πρέπει να ξεκινήσουμε γιατί έχουμε περιορισμένο χρόνο στη διάθεσή μας και έχει κατανεμηθεί ο χρόνος στους αγορητές με τρόπο ιδιαίτερα αυστηρό. Κυρία Υποψήφια Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, ο στόχος μας είναι να προχωρήσουμε στην ακρόαση της κυρίας Δαμανάκη που είναι υποψήφια επίτροπος για τη θέση του Επιτρόπου Θαλασσίων Ζητημάτων Βάσει των συνθήκων και του άρθρου 17 του κανονισμού μας θέλω να σας καλωσορίσω και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στην ακρόαση αυτή. Στην ακρόαση αυτή θα είναι παρόντες μαζί με τους βουλευτές Επιτροπής Αλίας και μια αντιπροσωπεία βουλευτών από την Επιτροπή Μεταφορών οι οποίοι και αυτοί θα λάβουν το λόγο, θα θέσουν ερωτήσεις στο τέλος της ακρόασης. Εμείς ε, αυτή η ακρόαση μας μάλλον μεταδίδεται κατευθείαν από το διαδίκτυο και θα παραμείνει διαθέσιμο το αρχείο της ακρόασης αυτής στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου. Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι γνωρίζετε τους κανόνες παρέμβασης από στην ακρόαση αυτή. Όλοι γνωρίζουν ακριβώ πώ θα διεξαχθεί η ακρόαση. Φυσικά και η κυρία Δαμανάκη. Δεν θεωρώ ότι είναι σκόπιμο να τη υπενθυμίσω. Απλώ σα λέω ότι θα είμαι πάρα πολύ αυστηρή στην τήρηση του χρόνου. Πριν από τις διακοπές των Χριστουγέννων. Η κυρία Δαμανάκη έδωσε την απάντησή τη στις έγγραφες ερωτήσεις οι οποίες είχαν διατυπωθεί από την Επιτροπή μας. Οι απαντήσεις αυτές έχουν διανεμηθεί σε όλους τους βουλευτές, βουλευτές μεταφρασμένες σε όλες τις επίσημες γλώσσες. Πριν δώσω το λόγο στην κυρία Δαμανάκη και στους συντονιστές των πολιτικών ομάδων και του υπόλοιπους βουλευτές, ως πρόεδρος θα ήθελα να κάνω ορισμένε εισαγωγικέ παρατηρήσει. Κυρία Δαμανάκη, όπως γνωρίζετε το ερωτηματολόγιο το οποίο αναφέρεται σε εσά ως υποψήφια επίτροπο θέτει ορισμένε ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με τις αρμοδιότητες των επιτρέπων. Λαμβάνοντα υπόψη την σημασία των προκλήσεων που προκύπτουν από την εφαρμογή τη συνθήκη τη Λισαβόνα, η Επιτροπή Αλία αποφάσισε να επικεντρωθεί σε θεσμικά θέματα θέτοντά σα πέντε συγκεκριμένα ερωτήματα σε σχέση με τι δεσμεύσει που περιμένουμε από εσά σε σχέση με τι σχέσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ημών συγκεκριμένα με το Κοινοβούλιο. Οι <clears throat> απαντήσει σα όμω, μου φαίνεται ότι είναι ασαφεί. δεν διαφαίνεται <clears throat> συγγνώμη, μια θέλησή σας να αναλάβετε συγκεκριμένες δεσμεύσεις εναντί του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρέπει να πω ότι είμαστε κάπως απογοητευμένοι. Αυτό δίνει την εντύπωση ότι η Κομισιόν δεν έχει λάβει υπόψη το γεγονός ότι ετέθησε εφαρμογή δίκη Λισαβόνα. Αυτό δεν είναι προσωπική παρατήρηση προ προς ε, εσά. Επομένω, θα θέλαμε με τι ερωτήσει μα να σα δώσουμε μια νέα ευκαιρία να έχετε μια σαφή στάση σε σχέση με τι δεσμεύσει που αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα θέματα αυτά. Και αφορούν πληροφορίες που θα έπρεπε να δοθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο και το γεγονό ότι θα πρέπει να δίνονται οι πληροφορίε αυτέ συγχρόνω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και επίση αφορούν τη συμμετοχή των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στι μεικτέ επιτροπέ για την εφαρμογή αλληλευτικών συμφωνιών, όπω επίση και σε συμμετοχή σε συνεδριάσει όπου εμπλέκονται διεθνεί οργανισμοί, όπου θέλουμε και διεκδικούμε ίση εκπροσώπηση με του εκπροσώπου του Συμβουλίου θα θέλαμε λοιπόν και πάλι να υπάρξει μια ανταπόκριση από την πλευρά της Κομισιόν δεδομένη και τη εφαρμογή τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Φυσικά δεν είναι τα μόνα ερωτήματα τα οποία θα τεθούν σε εσά κατά τη διάρκεια αυτή τη ακρόαση. Οι παρόντε βουλευτέ θα θέσουν ερωτήσει πιο ενδελεχεί και πιο συγκεκριμένε σε σχέση με την πολιτική αλλία και γενικά τι θαλάσσιε πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και <clears throat> εφόσον έχω ήδη καταλάβει δύο λεπτά χρόνο Θα σας δώσω το λόγο κυρία Δαμανάκη για τις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις κατά μέγιστο για 10 λεπτά. Έχετε το λόγο λοιπόν κυρία Δαμανάκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη Πρόεδρε κυρία Φράγα, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, είναι μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως υποψήφια επίτροπος. Πρόκειται για κορυφαία στιγμή στη ζωή κάθε πολιτικού όπως εγώ, με μακρόχρονη θητεία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, στο Κοινοβούλιο μιας χώρας που έχει βαθιές ρίζες στην Ευρώπη. Οι προσωπικές ευρωπαϊκές μου υποπιθήσεις είναι ισχυρές. Μπορώ να το πω αυτό διότι είναι αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης πολιτικής πορείας, η οποία δεν ήταν πάντα εύκολη. Είχε κόστος. Η Ευρώπη έχει μια ισχυρή πολιτική αλληλείας εδώ και δεκαετίες, μια από τις λίγες κοινέ πολιτικές. Θέλει επίσης να αναπτύξει τον τομέα της θαλάσσιας πολιτικής με τρόπο συνεκτικό και με αηφορία. Πρέπει να πετύχουμε. Καλωσορίζω θερμά το γεγονός ότι στο νέο θεσμικό περιβάλλον της συνθήκης της Λισαβόνας η αλία θα είναι στο εξής αντικείμενο συναπόφασης ως συνήθις νομοθετική διαδικασία. Έτσι διασφαλίζεται ένας ακόμη μεγαλύτερος ρόλος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στον τομέα αυτό τον οποίο συζητούμε, έχουμε μια στέρεη βάση να χτίσουμε, χάρη στη δουλειά που έκαναν οι προκάτοχοί μου και ιδιαίτερα ο κύριος Μπόρτζ. Ωστόσο υπάρχουν πλευρές όπου μπορούμε όλοι μαζί, όλοι μαζί εννοώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή, τα κράτη-μέλη, οι κοινωνικοί εταίροι, να αλλάξουμε προς το καλύτερο. Allow me now to touch on fisheries. Επιτρέψτε μου τώρα να ξεκινήσω με την αλία και να περάσω στην αγγλική γλώσσα γιατί θα πρέπει να χρησιμοποιήσω την τεχνική ορολογία όπως την έμαθα το τελευταίο καιρό από τα αγγλικά. Για την αλία λοιπόν πρώτα. Η τρέχουσα αναμόρφωση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής είναι ζωτική σημασία και θα αποτελέσει ασφαλώ κεντρικό ζήτημα τη δουλειά μου. Από τις 400 περίπου φορές που έχουμε λάβει στη διαβούλευση βλέπουμε ότι έχει επιτύχει αυτή η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης της Πράσινης Βίβλου. Και θα λάβω τα αποτελέσματά της πολύ σοβαρά υπόψη, όπως επίσης βέβαια και τις απόψεις της Επιτροπής σας. Έχει έρθει η ώρα για αποφάσεις και για εφαρμογή αυτών. Έχω τέσσερις κύριες λέξεις να σας δώσω. Καταρχάς, αηφορία που είναι μια λέξη κλειδί για τις προτάσεις που σας υποβάλλω, τόσο σε εσάς όσο και στο Συμβούλιο. Περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική αηφορία. Πιστεύω ότι μπορούμε να συγκεράσουμε τις τρεις αυτές μορφές και, και να βρούμε την ισορροπία μεταξύ των τριών αυτών και να εξασφαλίσουμε την αρμονική του συνύπαρξη και συνεργασία όχι μόνο μακροπρόθεσμα αλλά και εδώ και τώρα. Και πιστεύω ότι μπορούμε να αλλιεύουμε λιγότερο και να κερδίζουμε περισσότερα. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πλεόνασμα αλλιευτικής ικανότητας των στόχων μας, το overcapacity, ώστε να κάνουμε την αλλία μας περισσότερο προσοδοφόρα. Και ταυτόχρονα έχουμε υποχρέωση να ψωτεύσουμε την αλλία μικρής κλίμακας από αρνητικές συνέπειες. Η αλλία δεν είναι μόνο μια διατροφική πηγή. Για τις παράκτης περιοχές μας συνεπάγεται ασφάλεια, διαφύλαξη του πολιτισμού και της ιστορίας, είναι ένας τρόπος ζωής μια ζωή με πολλές δυσκολίες, τις οποίες γνωρίζω καλά, γιατί είμαι γεννημένη σε ένα ψαράδικο χωριό και μόνο η προσοδοφόρα αλληλεία μπορεί να διασφαλίσει το επίπεδο ζωής των ψαράδων και των οικογένειών τους. Για να είναι όμως προσοδοφόρα η αλληλεία θα πρέπει να έχουν οι θάλασσες ψάρια κατά τρόπον αιφόρο Μπορούμε λοιπόν να ψαρεύουμε λιγότερο και να αξιοποιούμε περισσότερο την αλία, να προωθήσουμε τις κατάλληλες μεθόδους διαχείρισης και να αναπτύξουμε ηχθειοκαλλιέργειες οικολογικές. Μπορούμε να αφήσουμε στο παρελθόν την πρακτική των απορρίψεων, discards, και πρέπει χρειάζεται να επενδύσουμε στην ποιότητα, στις, στα φρέσκα προϊόντα, στην πιστοποίηση για τα προϊόντα μας, ώστε να παρέχουμε καλή ποιότητα στροφή στις ευρωπαϊκές οικογένειες, στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Δεύτερη λέξη κλειδί, δημοκρατική υπευθυνότητα. Για όλους τους εταίρους στον τομέα μας. Γιατί η αλληλευτική πολιτική είναι μια κοινή πολιτική που μπορεί να επιτευχθεί κατά την έποψή μου μόνο εάν συμφωνήσουμε ότι δεν θα λαμβάνονται όλες οι αποφάσεις στο ύψιστο δυνατό επίπεδο, σε κάθε λεπτομέρειά τους. Πρέπει δηλαδή να προχωρήσουμε στην αποκέντρωση, στην περιφερειοποίηση της πολιτικής μας. και να εξασφαλίσουμε την ενεργό εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων με απόλυτο βέβαια σεβασμό στις συνθήκες. Η παγκόσμια διάσταση τώρα είναι η τρίτη λέξη κλειδί Πρέπει να προσαρμοστούμε στον 21ο αιώνα. Χρειάζονται καλύτερα αποτελέσματα από τις, για τις αλληλευτικές συμφωνίες με ένα διεθνές περιβάλλον ασφαλές και αποτελεσματικό και ταυτόχρονα θέλουμε και πλεονεκτήματα αναπτυξιακά και για τις χώρες εταίρους. Αηφορία νέε θέσει εργασία, προποθέσει ανάπτυξη για τη συνδυαστική του βιομηχανία και σεβασμό των δημοκρατικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτοί είναι οι τομεί στου οποίου το Κοινοβούλιο έχει και τι γνώσει και την ισχυρή παρουσία, που θα μπορούσε όμω και να ενισχύσει. Η σύνθηκη τη Λισαβόνα που θέτει σε βάση ισοτιμία στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, απαιτεί εδώ μια ποιοτική αλλαγή και συμφωνώ εδώ με την κυρία Πρόεδρο Πλην όμω, το θέμα αυτό δεν είναι αποκλειστικά δική μου ευθύνη, Είναι θέμα εγκάρσιο, οριζόντια όπω λέμε πολιτική που αφορά όλη την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Και αυτό που θα ήθελα να πω εγώ είναι ότι θα προσπαθήσω να εξαντλήσω κάθε περιθώριο, κάθε περιθώριο, το εννοώ αυτό, ώστε να έχουμε μια καλύτερη ανταπόκριση στο νέο και απάντηση στο νέο κανονιστικό πλαίσιο συμφωνία. Η τέταρτη λέξη κλειδί, η συμμόρφωση. Εξίσου σημαντική με τι προηγούμενους. Εδώ κρίνεται η αξιοπιστία της πολιτικής μας και χρειαζόμαστε εγγυήσεις για υγιή ανταγωνισμό με τα γειτονικά μας κράτη, με τα κράτη που αλλιεύουν στα ίδια ύδατα. Στηρίζομαι λοιπόν και στη δική σας ρητή υποστήριξη για ένα πλαίσιο ελέγχου. Χρειάζεται συνεργασία με τα κράτη-μέλη, ώστε να επιτύχουμε στενή παρακολούθηση της βιομηχανίας μας και να εξασφαλίσουμε την ουσιαστική απαγόρευση των εισαγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προϊόντων που προέρχονται από παράνομη, αδευκρινιστική και αδήλωτη δραστηριότητα και αν μου επιτρέπετε τώρα θα περάσω στα θέματα της ναυτιλίας, της θαλάσσιας πολιτικής. Η γαλάζια βίβλος διαθέτει τη στήριξη και την προωθητική βούληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Έχει έρθει λοιπόν η ώρα τώρα να προχωρήσουμε περισσότερο από την απλή αναζήτηση συμφωνιών και συνεργασιών και να προχωρήσουμε περισσότερο σε μια ολοκληρωμένη πολιτική διαχείριση των θαλάσσιων λέκανων με συγκεκριμένε απαντήσει στα συγκεκριμένα προβλήματα, όπως άλλωστε έχει περιγράψει και ο πρόεδρο Μπαρόσο στι πολιτικέ του κατευθύνσει. Εγώ προερχόμενη από νησί με πλούσια ναυτική παράδοση, που ανέρχεται στα βάθη τη αρχαιότητα, στα βάθη τη ιστορία, του μονοϊκό πολιτισμό, είμαι υπερήφανη αν μου δοθεί ευκαιρία να συμβάλλω και ε, από πλευρά μου στη γαλάζια ανάπτυξη στην Ευρώπη. Μπορούμε να εστιαστούμε λοιπόν σε ευκαιρίε για γαλάζια ανάπτυξη, και να ναυτιλιακή χωροταξία μπορεί να απελευθερώσει τι δυνατότητε των θαλάσσιων πόρων για εναλλακτική ενέργεια, για μεταφορέ με χαμηλέ εκπομπέ άνθρακα, για διευρωπαϊκά ενεργειακά δίκτυα και γαλάζια βιοτεχνολογία. Η λεωφόρη τη θάλασσα, η ενδοευρωπαϊκή ναυσιπλοεία και ο παράκτιο τουρισμό μπορούν να αποκτήσουν και να προσφέρουν νέε προοπτικέ. Δημιουργία γαλάζων θέσεων εργασία Στην κατεύθυνση αυτή μπορεί να συνεισφέρει η προώθηση και η ανάδειξη των δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη θάλασσα και την αυτιλία και η θεσμοθέτηση πιστοποιητικού ναυτιλιακή αριστεία. Τρίτο θέμα στη θαλάσσια πολιτική, η ασφάλεια των πολιτών τη Ελία και των μεταφορών. Η ανάπτυξη ενό νέου ε, ολοκληρωμένου συστήματο θαλάσσια επιτήρηση αποτελεί μια βασική πρόκληση για τη δημιουργία ενό ευρωπαϊκού θαλάσσιου χώρου χωρί εμπόδια, χωρί φραγμού. Και τέταρτον, η ενίσχυση τη οικονομία τη γνώση χάρη στην ε, πρωτοποριακή ευρωπαϊκή έρευνα για τη θάλασσα μπορούμε να συμβάλλουμε στη δημιουργία και την ε, απρόσκοπτη λειτουργία νέων ολοκληρωμένων δικτύων θαλάσσιας παρακολούθησης με το Emodent και με το Mar Atlas, τον Ευρωπαϊκό Χάρτη δηλαδή Θαλασσών. Και έτσι, εάν επικυρωθεί η εκλογή μου ως Επιτρόπου Ναυτιλίας και ε, Αλίας. Θα δουλέψω σκληρά για να επιτύχουμε μια πραγματική και θετική διαφορά στην καθημερινή ζωή όσων εξαρτώνται από την αλληλεία και το παράκτιο περιβάλλον μας. Θα το θεωρήσω μέγιστη τιμή το να μου επιτραπεί να συμβάλλω από πλευρά μου σε εταιρική, ουσιαστικά εταιρική σχέση μαζί σα, σε στενή συνεργασία μαζί σα, έτσι ώστε η αλληλεία μα, έτσι ώστε το θαλάσσιο περιβάλλον μα να έχει ένα πραγματικό μέλλον. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία υποψήφια. Στη συνέχεια θα περάσουμε τον πρώτο γύρο ερωτήσεων από τους συντονιστές. Καταρχήν, για δύο λεπτά ο κύριο Αντινόρο έχει το λόγο. Ε. Καλημέρα σα, Κύριε Επίτροπε, να σας καλωσορίσω στην Αλλιευτική Επιτροπή. Εσεί ε, σταθήκατε στα, σαν από τα πρώτα ζητήματα τα οποία θα ήθελα να θίξω κι εγώ. Μιλήσατε για την ε, σημαντική στιγμή που διαβιούμε, διότι στα πλαίσια της συναπόφασης η Επιτροπή Αλίας θα διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο και ελπίζω να μπορέσουμε να συνεργαστούμε πολύ καλά μαζί σας. Ξέρετε ε, ότι εργαζόμαστε για την πράσινη βίβλο, για τη σύνταξή της και ελπίζω να μπορέσουμε να συνεργαστούμε και για τη Λευκή Βίβλο, την οποία και αναμένουμε από εσά συγκεκριμένες απαντήσεις. Ως προς την περιφερειοποίηση, στην οποία αναφερθήκατε και εσείς, θα θέλαμε να ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να συνεπάρξει η κοινή ευρωπαϊκή πολιτική αλίας και η περιφερειοποίηση της, διότι θα πρέπει να έχουμε έναν μακρόπνο ορίζοντα για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Ως προς τη σήμανση, χαίρομαι που αναφερθήκατε στο ζήτημα αυτό, αλλά θα πρέπει να δούμε ποια οδό θα πρέπει να ακολουθήσουμε και στο θέμα της ε, σήμανσης μακροχρόνια. Κυρία Δαμανάκη, για τρία λεπτά έχετε το λόγο. Ε, ευχαριστώ τον κύριο συνάδελφο, τον κύριο Αντινόρο για την ερώτηση. Ε, πράγματι αυτά τα ζητήματα μας απασχολούν. Ε, σας είπα ήδη ότι έχουμε 400 συνεισφορές ε, στη συζήτηση από το κοινό και τους stakeholders για την Πράσινη Βίβλο. Πάρα πολλές από αυτές τις συνεισφορές αναφέρονται σε αυτή τη λέξη, decentralization, αποκέντρωση. Και υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές απόψεις για το πόσο καθένας εννοεί αυτή την αποκέντρωση. Θέλω να κάνω ευθύ εξ αρχή σαφέ ότι μιλώντας για αποκέντρωση δεν αναφέρομαι σε μία επανεθνικοποίηση της κοινοτικής πολιτικής. Η πολιτική αλίας είναι κοινή και θα παραμείνει κοινή. Αναφέρομαι όμως στην προσπάθεια να δούμε ποιες από τις αρμοδιότητες στα πλαίσια των συνθήκων και μπορούν, θα το δούμε αυτό όλοι μαζί σε μια πραγματική συνεργασία μπορούν να μεταφερθούν σε κατώτερα δυνατά επίπεδα. Δεν μπορώ να αντιληφθώ δηλαδή παραδείγματος χάρη για ποιο λόγο πρέπει το Συμβούλιο και εμείς και όλοι μας και η Επιτροπή να ασχολούμαστε με το μέγεθος ακριβώς που έχει το δίκτυ για τον ψαρά που ψαρεύει στη σκοτία το συγκεκριμένο είδος χάντοκ μπορούμε να πάμε σε μια λογική πιο αποκεντρωμένη, αλλά επαναλαμβάνω σε πλήρη σεβασμό προς τις συνθήκες. Διότι αυτό επιβάλλει, αν θέλετε, και η υποχρέωση που έχω εδώ ως υποψήφια επίτροπος. Επομένως, μπορούμε να συζητήσουμε αναλυτικά με ποιες μορφές θα το πετύχουμε αυτό. Πώς θα καταφέρουμε ώστε να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Ο στόχος θα είναι, αυτό που είπα, να έχουμε tailor-made solutions for sea basins δηλαδή να έχουμε ειδικέ λύσεις για κάθε θαλάσσια λεκάνη, για κάθε θαλάσσια περιοχή, από όλους τους ενδιαφερόμενους. Και είμαι πρόθυμη να συζητήσω μαζί σας το σχήμα αυτό, όπως είμαι πρόθυμη να συζητήσω ως ποιο σημείο θα μεταφέρουμε αρμοδιότητες. Όσον αφορά το labeling, τη σήμαση και την πιστοποίηση, είναι πολύ σημαντική, διότι θα μας δώσει τη δυνατότητα να συναγωνιστούμε με ίσους όρους ψαράδες από γειτονικέ χώρες που δουλεύουν στα δικά μας νερά για την Ιταλία, όπως και για την Ελλάδα, όπως και για άλλες μεσογειακές χώρες, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όπως και για άλλες χώρες όπου αντιμετωπίζουν ένα unfair competition από ψαράδες άλλων χωρών. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Δαμανάκη, ο κύριος ε, Αντινόρο θα ήθελε να δευτερολογήσει. Φαίνεται πως όχι. Περνάμε στην κυρία Ρόντας από τη Σοσιαλιστική Ομάδα. Έχετε δύο λεπτά για να διατυπώσετε την ερώτησή σας. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κυρία Δαμανάκη, καλώς ήρθατε. Χαίρομαι ιδιαίτερως που σας βλέπω εδώ και που θα έχουμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε. Για τον εξή λόγο. Ήσασταν για πολλά χρόνια βουλευτής και ξέρω ότι, έχετε αντιμετωπίσει τα προβλήματα μεταξύ βουλευτών αφενός και κυβερνήσεων υπουργών αφετέρου. Είστε εξοικειωμένοι με αυτές τις αντιπαραθέσεις και έχετε επιδιώξει πολλές φορές να εξασφαλίσετε καλή συνεργασία όσο δύσκολο και να ήταν αυτό. Και μια και έχετε πολλά χρόνια ε, κοινοβουλευτικού βίου, ξέρω ότι θα μας βοηθήσετε στο δικό μας έργο. Η ερώτησή μου λοιπόν, η μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής, όπως κάθε μεταρρύθμιση, είναι μια, μια μεταρρύθμιση με στόχους, δεν είναι δηλαδή τυχαία, και πλέον πολλά κοστίζει και πολλά χρήματα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι για την αντιμετώπιση των πιθανών οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών της μεταρρύθμισης. Με ολοκληρωμένη πολιτική για τη θάλασσα και την αναθεώρηση της, τη μεταρρύθμισή της, ασφαλώς και πάλι θα χρειαστούν πόροι αν και χρειάζεται μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική ασφαλώς, διότι χωρίς αυτή δεν μπορούμε να έχουμε την εξορρόπηση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών συνθήκων, γιατί διαφορετικά θα μας μείνει ούτε ψάρι στη θάλασσα. Γι' αυτό λοιπόν θα σας ρωτήσω πώς σκοπεύετε να πείσετε τους συναδέλφους σας, τόσο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και στο Συμβούλιο, για την χρηματοδότηση μιας επιτυχούς πολιτικής και μιας αηφόρας ε, μεταρρύθμισης, έτσι ώστε να μην θελήσουν να την κάνουν μηδενικά έξοδα. Έχετε τρία λεπτά για να απαντήσετε. Μπορούσα να πω ένα στίχο. With a little help from my friends. And I believe that uh, you will be my friend. Και πιστεύω ότι οι φίλοι μου θα είσαστε εσεί, Με λίγη βοήθεια από τους φίλους μου. Σε αυτόν τον αγώνα φίλοι μου θα είστε εσεί, γιατί αγώνα θα γίνει. It's all about economy, after all. Τελικά για την ε, οικονομία πρόκειται. Ασφαλώς ασφαλ... Ε, χρειαζόμαστε χρήματα και είμαι πολύ ευτυχή που οι συνάδελφοι έθεσε το θέμα. Ε, στην συζήτηση που θα κάνουμε για τα new perspectives ε, financial perspectives για τα επόμενα χρόνια, πιστεύω ότι θα μπορούμε να συνεργαστούμε ώστε να προβάλλουμε μια σοβαρή πολιτική χρηματοδότησης. Θα έχουμε τη δυνατότητα να πετύχουμε καλά αποτελέσματα αν είμαστε τεκμηριωμένοι και μπορούμε να πείσουμε ότι τα χρήματα που θα μας δοθούν θα αξιοποιηθούν. Το πρώτο λοιπόν στο οποίο νομίζω ότι πρέπει να επιμείνουμε είναι ότι χρειαζόμαστε χωριστό κονδύλι για το maritime policy, για, την, για τη θαλάσσια πολιτική, για την πολιτική ναυτιλίας. Δεν θα ήθελα να δεχθώ ε, τα χρήματα της αλληλείας, τα οποία δεν είναι πολλά. Όπως ξέρετε έχουμε ένα ποσό περίπου ένα δισεκατομμύριο το χρόνο, ούτε καν αυτό. Δεν θα ήθελα αυτά τα χρήματα να διατεθούν και για, το, ε, για την υπόθεση ναυτιλίας. Θα πρέπει να έχουμε ένα ξεχωριστό κονδύλι, ελπίζω ότι θα το διεκδικήσουμε μαζί και αυτή είναι μια πρώτη απάντηση στο ερώτημά σας. Από εκεί και πέρα για τα υπόλοιπα. Ε, είπα ότι θα κάνουμε προσπάθεια να διεκδικήσουμε χρήματα σε συνέργεια και με άλλες διευθύνσεις. Να πω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή με τη Διεύθυνση Έρευνας, DG Research και τον Επίτροπο, την αντίστοιχη Επίτροπο με την οποία έχω μιλήσει, ε, ετοιμάζουμε πρόγραμμα για τη θαλάσσια έρευνα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αναφέρεται στην κατάσταση των ωκεανών μα, θα δημιουργήσει, μάλλον είναι τρία προγράμματα. Ένα από αυτά αναφέρεται στην κατάσταση των ωκεανών μα, θα δημιουργήσει καινούργιε προποθέσει στην αξιοποίησή του και θα είναι ένα πρόγραμμα του οποίου τα κονδύλια δεν θα τα επιβαρυνθούμε εμεί, Με τη στενή έννοια μιλώ, θα είναι κοινοτικά κονδύλια από τον προπολογισμό τη ε, Επιτρόπου για την έρευνα. Αντίστοιχα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα, 10 δισεκατομμύρια ευρώ για την Αρκτική, το οποίο ετοιμάζεται. Θέλω να πω μπορούμε να εξασφαλίσουμε καλή συνεργασία και με άλλε διευθύνσεις για χρήματα, όπως επίσης με την Διεύθυνση Μεταφορών και την DG Transport, όπου έχουμε πολλά κοινά στο θέμα ε, maritime ε, και, άλλε και άλλες Από εκεί και πέρα το τελευταίο, στο οποίο θέλω να σταθώ, είναι ότι χρειάζεται να αξιοποιήσουμε τα δικά μας χρήματα καλύτερα. Όπως ξέρετε έχουμε το EFFF, το European Fisheries Fund, έχουμε επίσης και ένα δεύτερο εργαλείο για χρηματοδότηση. Τα χρήματα αυτά ε, στο πρώτο ταμείο κατανέμονται με βάση πέντε άξονες. Πολύ συνοπτικά θα μπορούσα να πω ότι θα ρίξω μεγάλο βάρος στον τέταρτο άξονα που αναφέρεται στο Sustainable Development. Είναι ανάγκη να αξιοποιήσουμε και τα λίγα χρήματα που έχουμε, όσα έχουμε, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να είναι πιο συμβατά με την ε, δική μας πολιτική. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Eh, Ευχαριστούμε κυρία Κύριε, κύριε Ρόντους, θέλετε να κάνετε ένα συμπληρωματικό ερώτημα. Όχι, δεν έχω να κάνω κανένα ερώτημα. Απλώς θέλω να διορθώσω αυτό το οποίο ελέγχθη προηγουμένως. Γιατί εγώ είπα νομίζω κάποια στιγμή για κοινή αγροτική πολιτική. Προφανώς εννοούσα την αλλιευτική πολιτική. Συγγνώμη για το θέμα αυτό. Eh, ευχαριστώ. Ακολουθεί ο συντονιστής της φιλελεύθερης ομάδας, ο κύριος Γκάλχερ, δύο λεπτά για να διατυπώσει το ερώτημά του. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να συγχαρώ την ε, υποψήφια Επίτροπο για τον διορισμό της και της εύχομαι κάθε επιτυχία. Εγώ θέλω να αναγνωρίσω την ε, έννοια αυτή της εταιρικής σχέσης που ανέφερε γιατί αυτό είναι απαραίτητο λόγω της συνθήκης της Λισαβόνας και χωρίς ακόμα τη συνθήκη Λισαβόνας θα ήταν απαραίτητο να αναπτυχθεί μια εταιρική σχέση. Πρέπει να γίνει ακουστή η άποψη της Επιτροπής Αλίας, η οποία εξάλλου αντιπροσωπεύει ένα πλούτο εμπειρία στον αλληλευτικό τομέα. Αναφερθήκατε σε μια στερεά βάση, αυτό είναι πολύ γενναιόδωρο εκ μέρου σα το αναφερθήκατε στο έργο του κυρίου Μπόρτ, ότι δημιούργησε στερεό έδαφο επί του οποίου μπορείτε να κτίσετε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η συνθήκη τη Λισαβόνα μα έχει δώσει ένα ενισχυμένο ρόλο στη λήψη αποφάσεων στον τομέα των αλλιευτικών θεμάτων με συναπόφαση. Επομένω, αναφερόμενο στην κοινή αλλιευτική πολιτική, αναφερθήκατε εσεί στο ρόλο των τριών θεσμικών οργάνων και αναφερθήκατε στον ίδιο τον αλληλευτικό τομέα και θα ήθελα εδώ να φέρω στην προσοχή σας κάτι το οποίο σίγουρα γνωρίζετε ότι πριν από τα Χριστούγεννα δεν ευδοκίμησαν οι διαπραγματεύσεις με τις νήσεις Φερόε έχουν εντωμεταξύ καταλήξει όχι ίσως με ιδιαίτερα επιτυχή τρόπο Ίσως όμως θα πρέπει να εστιάσετε την προσοχή σας στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν συμφωνίες με παράκτιες χώρες για τα θέματα του γάδου και αυτή τη στιγμή μπορούν οι χώρες αυτές να καθορίσουν μονομερώς τα αποθέματά τους. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει εδώ πέρα δυνατότητα να υπάρξουν συμφωνίε για αποθέματα τα οποία επικαλύπτονται των θαλασσίων περιοχών, μάλλον περνούν από μια θαλάσσια περιοχή στην άλλη. Και αυτό αφορά ιδιαίτερα την Νορβηγία και τα πελαγικά είδη. Ελπίζω λοιπόν ότι στο μέλλον θα έχετε μια πρακτική αντιμετώπιση για τα θέματα αυτά και την κατανομή των τάξεων των ε, συνολικών αλλιευμάτων. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τα καλά τους λόγια. Θέλω να επιβεβαιώσω αυτό που είπε πριν και η κυρία Ρόντας, ότι σε όλη μου την ε, ενήλικη ζωή ήμουν βουλευτής. Και αυτό σημαίνει ότι καταλαβαίνω πόσο σημαντικό και πόσο δύσκολο συγχρόνως είναι για τους βουλευτές να προσπαθούν να σταθούν με έναν τρόπο ε, ουσιαστικό, πολιτικό, αλλά συγχρόνως δημιουργικό απέναντι στην εκτελεστική εξουσία, αν μπορεί να θεωρηθεί ε, η Κομισιόν ότι έχει εκτελεστική εξουσία. Ε, γι' αυτό ελπίζω να εξακολουθήσω να έχω τη συνήθεια για μεγάλο διάστημα να βλέπω τα πράγματα από την άλλη πλευρά του λόφου, από την κοινοβουλευτική πλευρά. Τώρα όσον αφορά και αυτό, το λέω σε σχέση με την ανάγκη να υπάρξει πραγματική συνεργασία, real partnership, ανάμεσα σε εμά, στην Κομισιόν, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και να μπορέσουμε στο New Framework Agreement πραγματικά να βρούμε τον καλύτερη δυνατή λύση. Όσον αφορά το δεύτερο θέμα που έθεσε ο, κύριος, ο αξιότιμος κύριος βουλευτής, ε, θέλω να σας πω ότι σήμερα, κατά ευτυχή συγκυρία, ξαναρχίζουν οι συνομιλίες της Κομισιόν με την Ορβηγία. Η DG Mare από σήμερα αρχίζει τις συνομιλίες με την Νορβηγία. Είχαν διακοπεί για ένα μεγάλο διάστημα και αυτό είναι, ήταν μια δυσκολία που είχαμε ε, στις διαπραγματεύσεις που είχαμε με την Νορβηγία. Ε, είναι, η Νορβηγία, όπως ξέρετε, είναι μια μεγάλη χώρα, ε, γειτονική χώρα, μας ενδιαφέρει, ενδιαφέρει την Κομισιόν και όχι μόνο από την άποψη της Αλίας. Ε, την ενδιαφέρει και από άλλες απόψεις, όπως καταλαβαίνετε, που έχουν σχέση με την ενέργεια στην περιοχή, το maritime, τη δυνατότητα να υπάρχει διέλευση γενικότερα υπάρχει ένα θέμα καλών σχέσεων το οποίο πρέπει να σεβαστούμε. Χαίρομαι λοιπόν που επιτέλους ξαναρχίζουμε αυτές τις διαπραγματεύσεις που είχαν διακοπεί. Και είχαν διακοπεί για λόγους του οποίους υπενήχθηκε ο αξιότιμος κύριος Βουλευτής. Υπήρχε μία δυσαρμονία στη συζήτηση που κάναμε σε σχέση με το πώς ακριβώς θα κατανείμουμε τα αλλιευτικά δικαιώματα με δεδομένο ότι τα pelagic stocks και άλλα είδη, όχι μόνο τα pelagic, μετακινούνται προς βόρεια και διάφορων και των κλιματικών αλλαγών αλλά και εξαιτία ε, συγκυριακών αλλαγών. Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα πώς ε, σε, αυτή την περιοχή θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή λύση για όλους. Η Νορβηγία, επειδή ακριβώς είναι μια μεγάλη χώρα και γνωρίζει τη σημασία της για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητά να ε, υπησέρχεται και στην περίπτωση που έχουμε multi-annual planning, δηλαδή στην περίπτωση που έχουμε μακρόχρονα σχέδια, στον καθορισμό της ποσόστοσης που αντιστοιχεί σε κάθε χρόνο στα σχέδιά μας. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε ώστε να καταλήξουμε σε συμφωνία. Οι γειτονικέ χώρες είναι ανάγκη να βρίσκονται σε διάλογο μαζί μας και να καταφέρνουμε να έχουμε συμφωνία. Πιστεύω ότι η συμφωνία στην οποία θα καταλήξουμε θα λύνει με, το καλύτερο, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και την quota ε, του code, την ποσόστοση για το γάδο και όλα τα προβλήματα που έχουν σχέση με τα Faroe Island και την Ορβηγία. Eh, eh, eh, Ένα λεπτό συμπληρωματική ερώτηση, κύριε Γκάλεχερ, θέλετε. Ευχαριστώ, κύριε υποψήφια επίτροπε. Εάν σκεφτώ τη δική μου χώρα, 80% των αλλιευτικών σκαφών είναι κάτω από 15 μέτρα ίσαλης γραμμής, κάτι το οποίο σημαίνει ότι έχουμε αλληλεία μικρής κλίμακος και έχουμε επομένως τις παράκτιες αυτές νήσους οι οποίες έχουν πολύ σημαντική αλληλευτική δραστηριότητα που είναι σημαντική για τι κοινότητε αυτέ. Δεν υπάρχουν εναλλακτικέ πηγέ πλούτου για αυτέ τι περιοχέ. Θα ήθελα απλώ να μα πει η κυρία υποψήφια επίτροπο αν κατά τη διάρκεια τη αναθεώρηση τη κοινή αγροτική αλληλευτική πολιτική θα υποστηρίξει το να εισαχθούν σαφεί και συγκεκριμένε εξαιρέσει για την αλληλεία σε μικρά παράκτια νησιά. Και επίση τα περιφερειακά συμβούλια έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο τα τελευταία χρόνια και θέλω να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξη που έχετε πει ότι θα δώσετε στα περιφερειακά αλλιευτικά συμβούλια ώστε τα συμβουλευτικά αυτά συμβούλια να μπορέσουν να τεθούν και επιθεσμική βάση, γιατί νομίζω ότι μπορούν να παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Χαίρομαι λοιπόν που υποστηρίζει αυτή την προσέγγιση. Eh, για ένα λεπτό μπορείτε να απαντήσετε, κυρία Δαμανάκη. Ο αξιότιμο κύριο Βουλευτή έθεσε πολύ σημαντικά θέματα. Ε, περιορίζομαι να πω ότι όχι μόνο στη χώρα του, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα μικρά σκάφη είναι πλειοψηφία. Τα στοιχεία που ζήτησα δείχνουν ότι το 80%, το 80% συνολικά του ευρωπαϊκού ελευτικού στόλου είναι σκάφη κάτω από 12 μέτρα. Άρα μιλούμε για αυτό που λέμε small scale fisheries. Και επομένως χρειάζεται μία πολιτική. Δεν έχω το χρόνο να αναπτύξω λεπτομέρειες, ίσως και στη διάρκεια της συζήτησης, αλλά θα υπάρξει χωριστή πολιτική για τα μικρά σκάφη. Είναι ένα βασικό θέμα που πρέπει να συζητήσουμε και στα πλαίσια της, ε, ε, ε της αναμόρφωσης της πολιτικής αλληλείας που έχουμε μπροστά μας. Ε, νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε τις ε, καλύτερες λύσεις ώστε να προχωρήσουμε σε συνεργασία σε τέτοια κρίσιμα ζητήματα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, Θέλω να σας πενθυμίσω ότι η δευτερολογία δεν μπορεί να εισαγάγει μια νέα ερώτηση. Είναι απλώς συμπληρωματική ερώτηση. Η κυρία Λόβεν έχει το λόγο για δύο λεπτά. Συντονίστρια της ομάδας των Πρασίνων. Ευχαριστώ πολύ κυρία Δαμανάκη και συγχαρητήρια για την ε, υποψηφιότητά σας στην πολύ σημαντική αυτή θέση. Θα σας υπενθυμίσω ότι 71% του πλανήτη μας καλύπτεται από τους ωκεανούς. Και κέριος παράγων στα θαλάσσια συστήματα από τα οποία όλοι μας εξαρτώμεθα, ε, περιλαμβανομένης και της απορρόφησης διοξιδίου του άνθρακα, είναι η ε, με την υπεραλίευση λοιπόν έχουν μειωθεί κατά 70 ή 90% ακόμη μέσα σε 50 χρόνια τα αποθέματα ε, των ηχθείων στις θάλασσές μας και ιδιαίτερα στην περιοχή μας έχουμε προκαλέσει σημαντική αποσταθεροποίηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Κυρία Δακμανάκη, πιστεύετε ότι οι επιδοτήσεις ήταν κύριος μοχλός στην υπεραλίευση και πώς προβλέπετε την μείωση της υπεραλίευσης έτσι ώστε να διατηρήσουμε τους αλευτικούς μας πόρους αφού είναι ίδιος σπόρος οι ήχθιες και εφόσον πρόκειται για ένα βασικό πόρο της θάλασσας πώς θα πρέπει να κριθεί το ποια σκάφη θα πρέπει να αποσυρθούν και σε ποια θα δοθεί η δυνατότητα τη ε, αλίευσης. Δεν θα πρέπει αυτοί που έχουν τις βέλτιστες αλλιευτικές πρακτικές ε, με χαμηλέ επιπτώσει, ε, είτε στο βυθό είτε στα αλλιευτικά οικοσυστήματα, με χαμηλή κατανάλωση καυσίμων, με καλή κάλυψη των προϋποθέσεων και κανόνων, με καλή συμβολή στις τοπικές ε, κοινότητες. Δεν θα έπρεπε αυτά τα σκάφη λοιπόν να έχουν την προτεραιότητα της αλλιευτικής δραστηριότητας ή θα έπρεπε η αγορά μόνη της να κρίνει ποιος θα αναλάβει αυτή τη δραστηριότητα. λεπτά κυρία Δαμανάκη. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Ε, κυρία Λέβεν, συμφωνώ απολύτως με τα στοιχεία τα οποία παρουσιάσατε. Έτσι είναι τα πράγματα. Πράγματι έχουμε μία υπεραλίευση, ε, μία δραστική υπεραλίευση. Αυτά είναι τα στοιχεία τα επιστημονικά τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας και την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με έναν τρόπο ώστε ο πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εδώ θέλω να σας πω ότι 40% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζει σε παράκτιες κοινότητες. Ο πληθυσμός λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορέσει να αντεπεξέλθει σε αυτή την αλλαγή. Πρέπει λοιπόν όλη μας η πολιτική να είναι επιλεκτική, να καταλήγει στο στόχο της αηφορίας, συνδυάζοντας συγχρόνως και κοινωνικά μέτρα, ώστε οι κοινωνικές επιπτώσεις να μην είναι πολύ σκληρές για τους ασθενέστερους. Συμφωνώ ότι γι' αυτό δεν αρκεί μόνο η αγορά και γι' αυτό είμαι εδώ. Γι' αυτό είμαστε όλοι εδώ. Γι' αυτό η πολιτική της Κομισιόν, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια πολιτική που θέλει να ρυθμίσει την κατάσταση ώστε να οδηγηθούμε σε μια αηφορία, να οδηγηθούμε σε ένα μέλλον το οποίο και εγώ ονειρεύομαι, όπου θα υπάρχουν ψάρια για να ψαρεύουμε με ένα επικοδομητικό τρόπο, χωρίς να υπάρχουν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και οι επιπτώσεις ιδιαίτερα στα φτωχότερα στρώματα που ζουν στις παράκτιες περιοχές. Πώς θα το πετύχουμε αυτό. Ε, δώσατε μερικές ιδέες με τις οποίες συμφωνώ. Θα έλεγα ότι στο μέλλον πρέπει η χρηματοδότησή μας να γίνει πιο επιλεκτική. Δεν έχει νόημα, παραδείγματο χάρη, να χρηματοδοτούμε συνεχώς την ε, ε, δημιουργία νέων σκαφών, όπως κάναμε στο παρελθόν. Δεν έχει νόημα αυτό. Αυτό το οποίο χρειάζεται όμως να χρηματοδοτήσουμε είναι το, το modernization, τον εκμοντερνισμό των σκαφών μας, ώστε να έχουν τα κατάλληλα εργαλεία. Αν έχουμε παραδείγματος χάρη selective, gears, δηλαδή να το πω ελληνικά και δεν ξέρω πώς θα μεταφραστεί, ε, εργαλεία τα οποία μπορούν να κάνουν επιλογή, που έχουν μεγαλύτερη selectivity, τότε τα discards, οι απορρίψεις θα είναι πολύ λιγότερες το να έχουμε λιγότερες απορρίψεις είναι ένα στοιχείο κλειδί. Και άρα πρέπει η χρηματοδότηση να πάει επιλεκτικά σε αυτούς που κάνουν μοντερνισμό, εκμοντερνισμό των σκαφών τους. Είτε είναι μικρά είτε είναι μεγάλα. Ένα άλλο παράδειγμα. Εάν υπάρχουν ε, ψαράδες που ψαρεύουν σύμφωνα με τις διαδικασίες και σέβονται τους κανονισμούς, αυτοί θα πρέπει να επιβραβεύονται. Συμφωνώ μαζί σας. Και γι' αυτό αυτή η φράση που λέω decentralization και regionalization δεν είναι κενή περιεχομένου. Αποσκοπεί στο να δούμε και επιτόπου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πώς θα επιβραβεύουμε αυτούς που συμμορφώνονται. Ακόμα και στον καινούριο κανονισμό, το IU, ε, ε, Control, έχουμε παρόμοιες προβλέψεις. Ε, Ευχαριστώ. Ένα λεπτό συμπληρωματική ερώτηση, αν θέλετε, κυρία Λεβέν. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα <clears throat> να, να αναφερθείτε λίγο περισσότερο αν θέλετε για τις ιδέες σας για το πώς θα υπάρξει η μείωση του αληφτικού στόλου. Φαίνεται ότι έχουμε μια υπερβολική ικανότητα κατά 50% σε ορισμένους τομείς. Ποιος θα ήταν ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσετε να μειώσετε την αληφτική ικανότητα. Θεωρείτε ότι θα ήταν χρήσιμο να χρησιμοποιήσουμε το κριτήριο της περιβαλλοντικής αηφορίας σε ό,τι αφορά τη μείωση του αλευτικού στόλου. Ένα λεπτό. Που θέλω να πω είναι ότι τα εργαλεία που χρησιμοποίησαμε στο παρελθόν, όπως ήταν παραδείγματο χάρη το scrapping, δεν απέδωσαν αυτά τα οποία θα θέλαμε. Και καταλαβαίνω ότι η κριτική της ε, κυρίας Βουλευτού αναφέρεται και σε αυτό. Δεν μπορούμε λοιπόν να πάμε με τον ίδιο τρόπο, αυτό είναι βέβαιο πρέπει να πάμε με έναν τρόπο ώστε να χρηματοδοτούμε επιλεκτικά αυτά τα μέσα που βοηθούν ε, στο sustainable, στην αηφορία του τομέα. Το δεύτερο το οποίο επίσης μπορώ να πω είναι ότι η προσπάθειά μας πια έχει γίνει πιο συγκεκριμένη και αναφέρεται στον περιορισμό των ε, opportunities ε, for fisheries της ε, αλλιευτικής προσπάθειας, ακόμα και το σύστημα των tax and quotas είναι προσαρμοσμένο έτσι ώστε να εξασφαλίζει λιγότερες απορρίψεις. Άρα συνολικά η πολιτική μας μπορεί να φαίνεται πολύπλοκη, αλλά είναι μια πολιτική που εν τέλει καταλήγει στο να προστατεύσει την αηφορία. Ευχαριστώ. Στη συνέχεια ε, ε, παρέμβει ο κύριος Ζουκρόβαρτσίκη για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφια Επίτροπε, μετά όσα μας είπατε τώρα, για τον κατακαιρματισμό της πολιτικής για τις ποσοστώσεις και τη διαχείριση των αλληλευτικών αποθεμάτων, θα ήθελα να σας ρωτήσω από τα όσα έχουμε δει ως αποτέλεσμα των πολιτικών που έχει επιλέξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπό το φως της αποτυχίας του συστήματος των ποσοστώσεων. Δεν είναι η ώρα να σταματήσουν όλα αυτά, όπως άλλωστε είχε προεξαγγείλει και ο Επίτροπος Μπόρτς, και είσαστε διατεθειμένοι να εγκαταλείψετε το σύστημα των ποσοστώσεων και να προχωρήσετε μάλλον σε άλλα εργαλεία, όπως επί παραδείγμα τη διαφορετική κατανομή των αλλιευτικών σκαφών Και αναφέρομαι και στην ε, γραπτή σας απάντηση, τη σχετική με την ε, Βαλτική θάλασσα, για να ρωτήσω εάν τα πελαγικά είδη, στα οποία αναφερθήκατε κυρίως ε, της βιομηχανικής χρήσης, όχι προς κατανάλωση, θα τα αντιμετωπίσετε, θα τους επιφυλάξετε ειδική μεταχείριση. Γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με είδη τα οποία χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφή, ως ε, ε, ζωάλευρα, ηχθιάλευρα συγκεκριμένα και αποτελούν για μας ιδιαίτερα επικίνδυνα είδη. Ερωτώ λοιπόν εάν ε, θα, θα προτιμήσετε να στρέψετε αυτή την παραγωγή στην κατανάλωση προσβρόσεων και όχι βιομηχανική χρήση. Ο βουλευτή έθεσε ζητήματα τα οποία βρίσκονται στο κέντρο της συζήτησης που κάνουμε για την αναθεώρηση της πράσινης βίβλου. Έθεσε το θέμα της ενδεχόμενης αντικατάστασης του συστήματος των ποσοστώσεων από το σύστημα του περιορισμού της αλληλευτικής δραστηριότητας Παρόλο που δεν θέλω να προκαταλάβω τη συζήτηση, θέλω να απαντήσω όμως με όσο δυνατόν πιο ευθύ τρόπο απέναντι στο ερώτημα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να ανταποκριθεί σε όλες τις περιστάσεις και σε όλες τις ε, δυνατότητες αλίας που έχουμε στην Ευρώπη. Εάν υπήρχε και αν προκύψει από τη συζήτηση ή από τις δικές σας προτάσεις, να είστε βέβαιος ότι θα είμαι αμέσως πρόθυμη να το υιοθετήσω αλλά δεν έχω πιστεί και έχω πολύ ασχοληθεί με το θέμα, σας διαβεβαιώ, ότι μπορούμε τόσο απλά να αντικαταστήσουμε τις ποσοστώσεις με, τον περιορισμό της αλλιευτικής προσπάθειας. Δέχομαι ότι ο περιορισμός της αλλιευτικής προσπάθειας έχει πάρα πολλά θετικά και κυρίως βοηθά στο να μειώσουμε τα discards, τις απορρίψεις, το οποίο είναι θετικό. Αλλά δεν είναι τόσο απλό. Για να, το πω, για να πω, γίνω πιο συγκεκριμένη. Σε περίπτωση που έχουμε mixed fisheries, δηλαδή αλληλεία που συλλέγει πολλά διαφορετικά είδη, διαφορετικά είδη, θεωρώ ότι ο περιορισμός της αλληλευτικής προσπάθειας είναι το καλύτερο εργαλείο. Στην περίπτωση που έχουμε αλληλεία ενός μόνο είδους και υπάρχουν, έχουμε τέτοια αλίεια, και υπάρχουν εργαλεία που αφορούν ένα μόνο είδος, τότε ίσως για ένα διάστημα ακόμα θα πρέπει να μείνουμε προσιλωμένοι στο σύστημα tax and quotas θα πρέπει να δούμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο πώς θα συνδυάσουμε τα διάφορα εργαλεία που έχουμε. Προσωπικά επαναλαμβάνω, αντιλαμβάνομαι ότι το εργαλείο των, ε, του περιορισμού της αλληλευτικής προσπάθειας, αυτό το είδος management προσφέρει πλεονεκτήματα και είμαι πρόθυμη να το δώσω σε περίπτωση που πραγματικά αυτά θα φανούν. Όσον αφορά τη Βαλτική, Θέλω να πω ότι εδώ έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με το τοπικό ΡΑΚ, με το τοπικό συμβουλευτικό όργανο. Πολύ καλή συνεργασία και υπήρξαν περιπτώσεις όπου η διεύθυνση, ε, της οποίας έχω τη φιλοδοξία να προείσταμαι, ε, δέχθηκε πολύ σοβαρά υπόψη προτάσεις του Συμβουλίου της Βαλτικής. Και όσον αφορά την επιστημονική συμβουλή και όσον αφορά τα άλλα. Σκοπεύω μέσα στον επόμενο χρόνο να εξαγγείλω ειδικό μακρόχρονο πρόγραμμα για τα pelagic stocks της Βαλτικής. Θα έχουμε ένα καινούριο multi-annual program. Και στα πλαίσια αυτά θα μπορούμε να δούμε με έναν καλύτερο τρόπο τι μπορούμε να κάνουμε για το θέμα το οποίο θέσατε. Είμαι υπέρ των μακροχρόνιων προγραμμάτων γιατί αυτά εξασφαλίζουν μεγαλύτερη σταθερότητα και για την αλληλεία μας και για όλους τους εταίρους. Ε, και δίνουν τη δυνατότητα να συζητήσουμε καλύτερα και στο Συμβούλιο σας. Σε κάθε περίπτωση θέλω να πω ότι το Συμβούλιο της Βαλτικής θα ληφθεί σοβαρά υπόψη τις προτάσεις μας. Ευχαριστώ. Θέλετε να δευτερολογήσετε για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υποψηφία Επίτροπε, σε ένα θέμα στις γραπτές απαντήσεις αναφέρεστε στο πολιετές σύστημα για τον ε, Σολομό στην ε, Βαλτική θάλασσα. Αλλά ο γάδος είναι το πιο σημαντικό είδος ψαριού στη Βαλτική. Σκοπεύετε λοιπόν το ίδιο σύστημα το χρησιμοποιήσετε και για τον ε, μπακαλιάρο της Γλυλανδίας, κοντ ή μόνο για τον Σολομό. Ένα μακρόχρονο πρόγραμμα για τον γάδο, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη είναι ένα πρόγραμμα το οποίο εκτιμούμε συνεχώς σε συνεργασία με το Συμβούλιο και θα συνεχίσει η εφαρμογή του. Εάν χρειαστεί οτιδήποτε θα το δούμε μαζί. Αλλά το πολιετές πρόγραμμα για το Σολομό δεν υπάρχει και γι' αυτό το εξαγγέλλω. Είναι μια καινούργια πρωτοβουλία, πρέπει να υπάρξει. Ευχαριστούμε για την ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς για το λεπτό κύριος Φεραίρα. Ευχαριστώ. Κύριε, κυρία Επίτροπε, πολλές φορές αναφερθήκατε για την υπεραλίευση των αλλιευτικών στόλων και είπατε ότι είναι δυνατόν να αλλιεύσουμε λιγότερο ε, αυξάνοντας την αποδοτικότητά μας. Όπως ξέρετε, στην Πορτογαλία, στη χώρα μου, μετά από την ένταξή μας στην κοινή αλλιευτική πολιτική, μειώσαμε τον αλλιευτικό στόλο κατά 36% σε 10 χρόνια και το αλίευμα κατά 40%. Άλλες χώρες όμως, η Ολλανδία, η Γαλλία και η Ολλανδία αύξησαν τον αλλιευτικό στόλο από 12 έως 37%. Η Ισπανία αύξησε την παραγωγή κατά 10%. Η κατάσταση λοιπόν, κάτι το οποίο δεν προβλέπεται από, το, από την πράσινη βίβλο. Η κατάσταση διαφέρει από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Σε ε, μας η μείωση του ελευτικού στόλου δεν αύξησαν την παραγωγικότητα. Είχαμε και αύξηση του κόστους παραγωγικότητας και του κόστους εμπορίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο, στην κορύφωση της κρίσης το μόνο μέτρο που προέβαλε ήταν ο παροπλισμός του αλλιευτικού στόλου. Ποια μέτρα προβλέπετε έτσι ώστε να αυξήσουμε την αλλιευτική παραγωγικότητα. Κυρία Δαμανάκη, για τρία λεπτά. Η πολιτική αλληλείας είναι μια κοινή πολιτική. Αναφέρεται ως τέτοια ειδικά στις συνθήκες και εγώ αυτό θα το σεβαστώ απολύτως. Πρέπει όμως να κάνουμε την προσπάθεια να δούμε τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας. Συμφωνώ. Και να δούμε τα ιδιαίτερα προβλήματα, ώστε να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πράγματι, η Πορτογαλία είχε μία πολύ μεγάλη μείωση του δικού της στόλου. Μεγαλύτερη από τη μέση κοινοτική μείωση. Η μέση κοινοτική μείωση είναι περίπου 2% το χρόνο. Εσείς είχατε μεγαλύτερο ρυθμό. Περίπου διπλάσιο. Πράγματι, υπάρχει θέμα παραγωγικότητας. Είδα τα στοιχεία και πρέπει να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε όμως στα πλαίσια της κοινή πολιτικής που έχουμε. Σε αυτό θέλω να επιμείνω. Δεν μπορώ να υποστηρίξω επανεθνικοποίηση της κοινή αλλιευτικής πολιτικής. Όχι μόνο επειδή θεωρώ ότι θα είναι αντιπαραγωγικό και αντιοικονομικό, αλλά δεν το πιστεύω. Δεν μπορούμε να πάμε πίσω. Τι μπορώ να απαντήσω συγκεκριμένα στην ερώτησή σας. Έχω την εντύπωση ότι τα κακά οικονομικά στοιχεία στα οποία αναφερθήκατε συνδέονται με το γεγονός ότι το πολύ μεγάλο μέρος του πορτογαλικού αλλιευτικού στόλου είναι μικρά σκάφη. Πολύ μικρά σκάφη. Πρέπει λοιπόν να δούμε την χωριστή πολιτική, όπως είπα ήδη πριν, για τα small scale fisheries, που θα δίνει κίνητρα κυρίως στην ε, ανανέωση των εργαλείων και την ανανέωση του στόλου. Πρέπει να δούμε επίσης πώς μπορούμε να δώσουμε κίνητρα ώστε να υπάρχουν καλύτερες συνθήκες διατήρησης των αλλιευμάτων. Παραδείγματος χάρη θα μπορούσαμε να δώσουμε κάποια κίνητρα αν μπορούμε ή να συνεργαστούμε με, το regional, με τη διεύθυνση regional, με, το regional development ώστε να υπάρξουν κίνητρα για να υπάρξουν εγκαταστάσεις ψυγείων ε, ή αντίστοιχες καταστάσεις που θα βοηθήσουν στο να έχουμε καλύτερη παραγωγικότητα. Πρέπει να έχουμε καλύτερη συνεργασία στα πλαίσια της νέας χρηματοδοτικής πολιτικής με τους producers organizations, με τα συστήματα των παραγωγών. Ξέρω ότι οι ενώσεις παραγωγών δεν καλύπτουν όλους τους παραγωγούς, όλους τους αλείς, αλλά καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο μέρος, γύρω στο 57% σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και πιστεύω και στην Πορτογαλία το ποσοστό το οποίο δεν έχω υπόψη μου είναι αντίστοιχο. Πρέπει λοιπόν να δούμε με ποιο τρόπο εφαρμόζοντας τα κοινά μας εργαλεία θα βοηθήσουμε χωριστά κάθε περιοχή και κάθε χώρα. Έχω την εντύπωση πάντως ότι τα προβλήματα στις πορτογαλικές ακτές είναι παρόμοια με αυτά που είναι στις ακτές και άλλων χωρών της Μεσογείου και άλλων ευρωπαϊκών χωρών πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να βοηθήσουμε τα, αυτό που λέμε small scale fisheries, τα μικρά σκάφη, να επιβιώσουν. Με εξαιρέσεις, επαναλαμβάνω θα υπάρχουν εξαιρέσεις, παραδείγματο χάρη στο IUU Control προβλέπουμε ήδη μια εξαίρεση. Δεν είναι υποχρεωμένα αυτά τα σκάφη να εφαρμόσουν τη νέα τεχνολογία αμέσω. Και άλλες εξαιρέσεις τις οποίες θα δούμε. Ευχαριστώ. Eh, Δευτερολογία για ένα λεπτό. Επιμένω στην αύξηση της ε, παραγωγικότητας και θα ήθελα να σας ρωτήσω πότε προβλέπεται η μεταρρύθμιση της κοινή οργάνωσης της αγοράς. Αναφέρομαι στο έγγραφο το οποίο μας απεστάλει όπου αναφέρεται ότι η μεταρρύθμιση θα πρέπει να αποτελώσει μέρος μιας συνολικής, ενός συνολικού πακέτου. Εκεί θα υπάρξει διαφοροποίηση αναχώρα, δηλαδή η κοινή οργάνωση της αγοράς μεταρρυθμίστηκε στο παρελθόν, αλλά ε, αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε πότε προβλέπεται η μεταρρύθμιση της κοινή οργάνωσης της ε, αλλιευτικής πολιτικής. Κύριε Αδαμανάκη, για ένα λεπτό. Η μεταρρύθμιση του Common Market Organization για τα fisheries έχει καθυστερήσει. Ε, αλλά είπαμε και αποφασίσαμε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας κοινός νέος οργανισμός με βάση και την συνολική μεταρρύθμιση της αλλιευτικής πολιτικής θα ήταν λάθος να προχωρήσουμε στη μεταρρύθμιση αυτού του οργανισμού και μετά την αναθεώρηση της κοινή αλλιευτική πολιτικής να έχουμε μια νέα μεταρρύθμιση. Όπως καταλαβαίνετε θα είχαμε δύο διαφορετικά πράγματα που θα έπρεπε να συνδυαστούν και να έχουμε νέα μεταρρύθμιση εκ των υστέρων. Ε, αλλά πάντω, θέλω να επιμείνω σε αυτό που είπα. Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητή. Θα, έχουμε μεταρρυθμίσει, αλλά οι μεταρρυθμίσει θα οδηγούν στο να έχουμε τα καλύτερα όργανα, εργαλεία, instruments για κοινή αλλιευτική πολιτική. Για κοινή αλλιευτική πολιτική. Θα πάρουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητες, όλες τις ιδιαιτερότητες και τη διαστρωμάτωση, ε, τα διαφορετικά συμφέροντα και υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα, δεν το αγνώ, Άλλα είναι τα συμφέροντα των μεγάλων σκαφών, άλλα των μικρών, άλλα των χωρών, ώστε να το εφαρμόσουμε. Ευχαριστώ. Στη συνέχεια έχει το λόγο για δύο λεπτά ο κύριος Φάρατς από την ομάδα Ελευθερίας και Δημοκρατίας. Σα ευχαριστώ κύριε Δαμανάκη. Φαίνεται να υποστηρίζετε ότι η κοινή αλευτική πολιτική είναι επιτυχημένη. Είπατε ότι έχει μια στερεά βάση από μια βρετανική όμως οπτική γωνία. Ήταν μια συνολικά ολέθρια κατάσταση. Χαθήκανε δεκάδε χιλιάδων θέσεων εργασία όταν μπήκαμε στην ενιαία αγορά τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα ο Βρετανικό στόχος, στόλος μπορεί να συλλέξει μονάχα το 1 πέμπτο κατά αξία των ε, ηχθείων που κυκλοφορούν στα ύδατά μας η κοινή πρόσβαση σε ένα κοινό πόρο έχει μειωθεί από τη δική μας πλευρά και έχουμε κατέβει σε ένα ελάχιστο επίπεδο όπου έχουμε τη δυνατότητα μόνο 7% των ηχθείων στην, ε, στο διάβλο της μάχης μπορούν να συλλάβουν. Όλα αυτά λοιπόν είναι ικτρά. Το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν ο κυρίως ιτημένος αυτής της ε, διαδικασίας. Υπάρχει και ένα θέμα, το, υπάρχει κάτι το πυροθετικό, ότι η αθλητική αλληλεία στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε πολλά άλλα μέρη, ανθεί. Υπάρχει πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπων οι οποίοι ασκούνται στην ερασιτεχνική αλληλεία και είμαι ένα από αυτού. Τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλά ή πηγαίνανε πολύ καλά μέχρι ότου εμφανιστεί το άρθρο 47. Η πρόταση να αρχίσει να υπάρχει ρύθμιση και έλεγχο τη ερασιτεχνική αλληλεία. Και για μια φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λειτουργήσε πολύ λογικά και είπε ότι πρέπει να υπάρχουν εξαιρέσει και απόφαση σε επίπεδο κράτου μέλους, αλλά η Κομισιόν χτύπησε το χέρι στο τραπέζι, είπε όχι, αυτό πρέπει να ρυθμιστεί από ένα, σε ένα κεντρικό επίπεδο και πρέπει να το κάνει η Κομισιόν. Θέλω να σα ρωτήσω, εσεί έχετε την πρόθεση τα επόμενα πέντε χρόνια να εφαρμόσετε ένα συνολικό κανονισμό τη ερασιτεχνική αθλητική αλληλεία σέβομαι απολύτως τα στοιχεία του κυρίου βουλευτή όσον αφορά την κατάσταση στη χώρα του. Δεν θα συμφωνήσω όμως μαζί του ότι η κατάσταση αυτή, η χειροτέρευση της κατάστασης οφείλεται στην ευρωπαϊκή πολιτική, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν δυσκολίες ε, σε όλο τον πλανήτη, σε όλες τις χώρες και προσπαθούμε να τις αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ε, δεν θα κάνω διακρίσεις αν με τιμήσετε με την ε, υποστήριξή σας, αν με τιμήσετε με την αποδοχή σας, δεν θα κάνω διάκριση ανάμεσα σε καμιά χώρα και επομένως δεν μπορώ να δεχθώ τη λογική ότι κάποια χώρα είναι ιτημένη και κάποια άλλη είναι κερδισμένη από την πολιτική. Θα κάνουμε προσπάθεια ώστε να έχουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις για όλες τις θαλάσσιες λεκάνες, παίρνοντας υπόψη και τις ανάγκες περιφερειοποίησης της πολιτικής μας. Όσον αφορά το θέμα το οποίο θέσατε για την εραστεχνική αλία, θέλω να σας καθησυχάσω. Δεν σκοπεύω σε καμία περίπτωση να εντάξω την εραστεχνική αλία στα πλαίσια μιας κοινή ρύθμισης από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Θέλω να είμαι σαφή στο θέμα αυτό. Υπάρχουν αρκετοί κανονισμοί ε, σε επίπεδα κρατών μελών. Ε, κάθε κράτος μέλος μπορεί να ρυθμίσει το θέμα. Ε, θέλω να είμαι κατηγορηματική. Βεβαίως, για να είμαι επίσης απολύτως σαφής, τα αποτελέσματα και της εραστεχνικής αλίας οι επιστήμονές μας θα παίρνουν υπόψη στον υπολογισμό των στόξ των διάφορων ψαριών, στον υπολογισμό των αποθεμάτων μας. Ε, έτσι ώστε να μας δώσουν την καλύτερη δυνατή εικόνα για τα αποθέματα που υπάρχουν και στη χώρα σας και αλλού. Αλλά δεν θα υπάρξει κοινοτική ρύθμιση για την αεραστεχνική αλία. Θέλετε να θέσετε συμπληρωματικό ερώτημα. Ίσως θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο, λέει ο κύριος Φάρτς, αν για μια φορά κάναμε μια πραγματική ανάλυση, μια πλήρη ανάλυση κόστους κόστους-οφέλους για το κατά πόσο η ψυχαγωγική, η αεραστεχνική αλληλεία συμβάλλει στην ε, οικονομία μας. Γιατί δεν είναι μονάχα οι αλλοίς, είναι αυτοί οι οποίοι φτιάχνουν δολώματα, φτιάχνουν ε, εξοπλισμό αλλοίας. Είναι ένας τομέας λοιπόν ο οποίος έχει οικονομική άνθηση. Θα έπρεπε λοιπόν να έχουμε μια πλήρη ανάλυση κόστους ωφέλους και αντικτύπου για να δούμε κατά πόσον οι προτάσεις αυτές οι οποίες έχουν προταθεί θα έχουν άχθος για τον οικονομικό αυτό τομέα. Γιατί κινδυνεύουν να χαθούν εκεί θέσεις εργασίας και οικονομική δυνατότητα. Μπορούμε να έχουμε λοιπόν μια τέτοια ανάλυση. Ένα λεπτό, κυρία Δαμανάκη. Θα ήμουν πολύ ευτυχή, κύριε Φάρατζ, αν είχα μία ανάλυση και μία εκτίμηση εκ των υστέρων για όλε τι πλευρέ τη πολιτική μα. Και θέλω μάλιστα να πω ότι ε, θεωρώ πως αυτό είναι ένα δύνατο στοιχείο στην πολιτική μας που πρέπει να το ε, εμπλουτίσουμε. Πρέπει δηλαδή να προχωρήσουμε περισσότερο σε αυτό που λέμε ex post assessment κάθε πλευρά της πολιτικής μας, ώστε να έχουμε πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα. Θέλω να σας υποσχεθώ ότι στη διάρκεια της θητείας μου, εάν με επιβεβαιώσετε τον ορισμό μου, θα κάνω ό,τι μπορώ ώστε να έχουμε ε, τέτοια ex post ανάλυση για κάθε πλευρά της πολιτικής. Αλλά για την εραστεχνική ελεία είμαι λίγο διστακτική να προχωρήσουμε σε impact assessment ε, και ανάλυση ανάλυση τέτοιου τύπου, γιατί όπως καταλαβαίνετε <laughs> αυτό θα δώσει το μήνυμα ότι ενδεχομένως θέλω να υπαχθεί η αλία σε κοινό δίκαιο και θέλω να αποφύγω αυτή την εντύπωση. Σας ευχαριστώ. Τέλος, για να τελειώσουμε με τον πρώτο γύρο, εξ ονόματος των μη εγγεγραμμένων και για δύο λεπτά έχει το λόγο ο κύριος Λεπέν. Κυρία Επίτροπε, στην ανακοίνωσή σας αναφέρετε τις προτεραιότητες σας για να επανεξισορροπήσετε τα αλλιευτικά σκάφη και την εραστεχνική ε, αλία. Στον Οκτώβριο όμως πέρσι ε, ορίστηκε ένα χρονοδιάγραμμα σε σχέση με τα τέλη στα αλλιευτικά ε, σκάφη και τα αλλιεύματα. Όπως ξέρετε όμως διανύουμε μια περίοδο κρίσης και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό αποτελεί προδοσία στην ερασιτεχνική αλία. Έχουν δρακόντια μέτρα που πρέπει να υφίστανται οι αλίες και αυτό δεν ισχύει για τους αλιευτικούς πόρους γενικότερα. Τι θα γίνει σε σχέση με τις μεγάλες πολυεθνικές και τις μεγάλες βιομηχανίες μεταπίσεις σε σχέση ε, με τις, ε, με τις χώρες του Βορρά και τι θα γίνει σε σχέση με το γεγονός ότι οι μικροί αλληλείς ε, είναι ιδιαίτερα ανήσυχοι με τα αλλιεύματα, τα παράνομα αλλιεύματα. Τι θα κάνετε για να αντιμετωπίσετε την ε, παράνομη αλλία και τι θα κάνετε σε σχέση με τους δασμούς που τάσσονται υπέρ αυτού του είδους αλλίας. Η κυρία Δαμανάκη για τρία λεπτά. Ευχαριστώ τον κύριο Λεπέν για την ερώτηση. Ε, γνωρίζω και σέβομαι την οικογενειακή του παράδοση στον τομέα της ελίας όπως γνωρίζω επίσης ότι ο ίδιος είναι ερασιτέχνης, ψαράς και, ελπίζω, και επομένως αντιλαμβάνομαι ότι ξέρει πολύ καλά την κατάσταση. Δεν θα ήθελα η Κομισιόν να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη για το θέμα αυτό. Τα κράτη-μέλη έχουν την ευθύνη, δεν είναι ένας τομέας που έχει κοινοτικοποιηθεί και δεν θα ήθελα να εμφανιστώ κάνοντας προσπάθεια να τον κοινοτικοποιήσω. Τι θέλω όμως να πω. Ε, ως Επίτροπος είμαι υποχρεωμένη να αντιμετωπίσω τις συνέπειες όλων των σκαφών και όλων των αλλιέων στο περιβάλλον μας. Και θέλω να διαβεβαιώσω τον κύριο Λεπέν ότι δεν θα κάνω καμία διάκριση. Είτε μεγάλα σκάφη, είτε μικρά σκάφη, εφόσον ρηπαίνουν αναλογικά, η ρήπανση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, και θέλω να το πω με πολύ σαφή τρόπο, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε με προκαταλήψεις ένα μεγάλο σκάφος δεν ρηπαίνει πάντα πάρα πολύ αν έχει τα κατάλληλα εργαλεία. Όπως επίσης και ένα μικρό σκάφος, εάν δεν έχει τα εργαλεία, μπορεί να ρηπαίνει. Οι εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα είναι σχετικές και πρέπει να δούμε κάθε περίπτωση. Άρα, στο σημείο αυτό θα είμαι απολύτως δίκαια. Θα προσπαθήσω τουλάχιστον να είμαι απολύτως δίκαια. Τώρα, όσον αφορά τα θέματα εφαρμογής της πολιτικής μας, αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα Θέλω μόνο να πω ότι ο νέος κανονισμός, ο οποίος έχει εισαχθεί, δίνει τη δυνατότητα να έχουμε ένα καλύτερο σύστημα, έχουμε ένα point system στο θέμα εφαρμογής των αλλιευτικών κανόνων και νομίζω ότι η εφαρμογή του θα βοηθήσει πολύ ώστε να είμαστε όλοι περισσότερο αποτελεσματικοί. Ο νέος αυτός κανονισμός ε, ουσιαστικά ελέγχου, κανονισμός ελέγχου ουσιαστικά ενσωματώνει πάρα πολλούς κανονισμούς που είχαμε απλοποιεί την κατάσταση, δίνει δυνατότητα στους επιθεωρητές μας να κάνουν πραγματικό έλεγχο και δίνει επίσης κίνητρα επιβράβευση σε περίπτωση που κάποιος συμμορφώνεται με τις υποδείξεις που του γίνονται. Είναι ένα μοντέρνο και πιστεύω αποτελεσματικό εργαλείο και έτσι ακόμα και ε, στην περίπτωση της ε, εφαρμογής της νομοθεσίας μας όπου είχαμε τεράστια προβλήματα και το παραδέχομαι πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να έχουμε μια καλύτερη κατάσταση. Λέω είχαμε τεράστια προβλήματα διότι όπως ξέρετε κύριε Λεπέν και το Court of Auditors ε, έχει μιλήσει πολύ αρνητικά για την εφαρμογή της πολιτικής αλίας, πολύ αρνητικά και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε ώστε με τον καινούριο κανονισμό να απαντήσουμε και να ανταποκριθούμε στις απαιτήσει του. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό κύριε Λεπέν μπορείτε να δευτερολογήσετε. Θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτό το δικαίωμα κύριε Λεπέν. Σας ευχαριστώ πολύ που αναφερθήκατε στις οικογενειακές μου ρίζες. Κύριε Δαμανάκη, είχαν ε, δραστηριότητα ε, όχι εραστεχνική, ο πατέρας μου και ο παππούς μου. Εγώ ίδιος είχα επαγγελματική στη, στανιάτα μου και γνωρίζω καλά αυτό το σκληρό επάγγελμα του ψαρά. Αντιμετωπίζουν λοιπόν το πρόβλημα των μεταβιβάσιμων ποσοστώσεων ε, οι Γάλλοι αλης ε, λόγω της ε, διάλυση των, παλαιών, των μικρότερων σκαφών ήταν υπέρ αυτών των ατομικών μεταβιβάσιμων ποσοστώσεων ο προηγούμενος επίτροπος. Εσάς ποια είναι η θέση σας και θα θεσπιστεί το σύστημα αυτό μόνο για τους Ευρωπαίους γιατί τότε τι θα εμπόδιζε μια ευρωπαϊκή επιχείρηση να εξαγοράσει ποσοστό αλληλευτικέ και να τι πωλήσει σε ένα κράτο έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να αναλάβει αυτή τη δραστηριότητα μια έξω ευρωπαϊκή επιχείρηση. Κυρία Δαμανάκη, για ένα λεπτό. Όταν αναφέρθηκα στι οικογενειακέ σα παραδόσει, αναφέρθηκα κυρίω, κύριε Λεπέν, στο γεγονό ότι ο πατέρα σα άσκησε αυτή τη δραστηριότητα κάτω από δύσκολε συνθήκε, πραγματικά δύσκολε. Αλλά α έρθουμε στο παρόν. Ε, αναφερθήκατε στο ζήτημα των ITQs, των transferable quotas. Ε, είναι πολύ μεγάλο θέμα. Πολύ μεγάλο θέμα. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα, όπως ξέρετε πολύ καλά. Υπάρχει όμως σε ορισμένες χώρες, εφαρμόζεται σε ορισμένες χώρες, όπως παραδείγματος χάρη η Δανία, η οποία κρίνει ότι το σύστημα με την εφαρμογή και με τους κανόνες και με τους περιορισμούς που έχει βάλει στην μεταβίβαση των ITQs, το σύστημα είναι επιτυχές. Έχουμε και άλλα παραδείγματα. Έχουμε το πολύ αρνητικό παράδειγμα της Ισλανδίας, όπου πράγματι η εισαγωγή του κεφαλαίου με έναν βάρβαρο τρόπο στην Αλία οδήγησε στην κατάρρευση συνολικά του συστήματος. Ε, αυτό το οποίο έχω να πω είναι ότι το θέμα θα συζητηθεί πολύ διεξοδικά στα πλαίσια της ε, συζήτησης για το πράσινο βιβλίο. Ε, δεν μπορώ εκ των προτέρων να είμαι εναντίον οποιασδήποτε χρήσης αυτού του δικαιώματος εφόσον τα κράτη-μέλη το χρησιμοποιούν και είναι στην αρμοδιότητά τους να το χρησιμοποιήσουν. Δεν μπορώ να παρέμβω. Αλλά συμφωνώ ότι θα πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να εξασφαλίσουμε ώστε να μην οδηγηθούμε σε μια υπερσυγκέντρωση και καταστροφή ουσιαστικά της αλίας και ιδιαίτερα του small scale fisheries. Ευχαριστώ. Στη συνέχεια προχωρούμε στο δεύτερο γύρο ερωτήσεων εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων. Η κυρία Πατράου Νέβες έχει το λόγο για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Να καλημερίσω και την κυρία Δαμανάκη. Της εύχομαι κάθε επιτυχία και επιτυχία του τομέα. Η τελευταία μεταρρύθμιση του 2002 του τομέα όρισε και ανείχνευσε σοβαρές δυσχέρειες. Η υπεραλίευση, οι υπερβολικές επενδύσεις η κατάτμιση του αλλιευτικού στόλου χωρίς να μπορέσουμε να εντοπίσουμε αυτά τα δύο φαινόμενα. Επίσης υπάρχει υπερεκμετάλλευση ορισμένων αποθεμάτων και όχι σωστά πρότυπα διαχείρισης. Πιστεύω ότι θα πρέπει να προβούμε σε μια εκβαθέων μεταρρύθμιση αυτή τη φορά. Ποιες θα είναι οι προτεραιότητες θα προωθήσετε μία αποκέντρωση των αποφάσεων, ε, μία ε, διαφοροποίηση των μοντέλων διαχείρισης. Η κυρία Δαμανάκη για δύο λεπτά. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. ευχαριστώ και την κυρία Νέβες για την ερώτηση. Γνωρίζω ότι είναι υπεύθυνη για μια πολύ σκληρή δουλειά. Πολύ σκληρή δουλειά πραγματικά το να ετοιμάσει την έκθεση για το πράσινο βιβλίο και ξέρω ότι ήδη έχει να κάνει με πολλές εκατοντάδες τροπολογίες που έχουν κατατεθεί. Δεν έχω μπορέσει να δω αναλυτικά όλες τις τροπολογίες, είναι κάπου 300 τόσες, αλλά έχω δει το, τη δουλειά που έχει γίνει μέχρι τώρα, την έκθεσή της, τον draft της έκθεσής της και θέλω να πω ότι έχει πολλές καλές ιδέες τις οποίες σκοπεύω να αξιοποιήσω. Πώς θα προχωρήσουμε. Ε, οι προτεραιότητες θα είναι τέτοιες ώστε να απλοποιούν κατά το δυνατόν την νομοθεσία που έχουμε και συγχρόνως να την κάνουν ε, πιο αποτελεσματική. Θα μου πει κάποιος ότι αυτό που ψάχνω είναι πραγματικά να τετραγωνίσω τον κύκλο, αλλά εν πάση περιπτώσει θα καταφύγω στην ελληνική παράδοση στη γεωμετρία ελπίζοντας ότι θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ είναι πράγματι δύσκολο να συνθέσουμε τα διαφορετικά συμφέροντα που συγκρούονται σε αυτό το τομέα. Γιατί υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα και νομίζω όλοι το καταλαβαίνετε αυτό. Υπάρχουν τα συμφέροντα των καταναλωτών, υπάρχουν τα συμφέροντα των ψαράδων, τα συμφέροντα των μικρών ψαράδων, τα συμφέροντα της βιομηχανίας, τα συμφέροντα της βιομηχανίας μεταποίησης, τα συμφέροντα των ε, περιοχών, των coastal regions, τα τουριστικά συμφέροντα. Είναι δύσκολο. Ε, και φαντάζομαι ότι και η κυρία συνάδελφος, η κυρία αυτό το αντιλαμβάνεται. Οι προτεραιότητες ε, περίπου ανάγονται στις τέσσερι λέξεις τις οποίες ανέφερα ως λέξεις κλειδιά στην ε, ε, αρχική μου ομιλία. Θα, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για sustainability, για εφορία, ό,τι μπορούμε ώστε να αυξήσουμε την δημοκρατική ευθύνη, ε, καλύπτοντας και τα θέματα αυτά του decentralization και regionalization τα οποία αναφερθήκατε. Θα κάνουμε μία προσπάθεια να έχουμε καλύτερη συμμόρφωση στις αποφάσεις μας. Θα κάνουμε προσπάθεια ώστε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά εργαλεία πολιτικής. Ε, καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο, αλλά θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε ε, σε συνεργασία μαζί σας. Για μισό λεπτό η κυρία Πατράου μπορεί να δευτερολογήσει αν θέλει να χρησιμοποιήσει αυτό το δικαίωμα. Ευχαριστώ. Αναφέρθηκα στον εντοπισμό και χαρακτηρισμό του αλληλευτικού στόλου. Θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο στη διάκριση μεταξύ ερασιτεχνικού και βιομηχανικού στόλου μπορείτε να προβείτε σε μία ουσιαστική διάκριση για ιδιαίτερα ευαίσθητα θέματα σε σχέση με τα διαχειριστικά πρότυπα. Δεν ξέρω κατά πόσο προβλέπετε επενδύσεις για τη διενέργεια ε, μελετών ως προς τις ε, διάφορες ε, προδιαγραφές και μοντέλα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ενδεχομένω. Κύριε Δαμανάκη, για μισό λεπτό. Η διάκριση ανάμεσα στον ερασιτέχνη ψαρά και αυτόν που κάνει βιομηχανική αλία είναι σχετικά απλή. Περιορίζομαι να πω ότι για μένα ερασιτέχνης ψαράς είναι αυτός που δεν πουλά το προϊόν του δεν θα μπορεί να πουλά το προϊόν του. Η διάκριση ανάμεσα σε αυτό που λέμε small ε, scale fisheries και, τους, και την ε, βιομηχανία είναι πιο δύσκολη. Εδώ τα κριτήρια είναι πιο σύνθετα και πρέπει να το συζητήσουμε στα πλαίσια της κοινή πολιτικής. Θα έλεγα ότι γενικά τα κριτήρια που μέχρι τώρα χρησιμοποιούμε είναι να μην έχουμε σκάφη μεγάλα, χρησιμοποιούμε το μέγεθος και συγχρόνως δεν επιτρέπουμε στα μικρά σκάφη να υπάρχουν σειρώμενα εργαλεία. Ε, είναι όμω μεγάλο θέμα. Και... Ε, κύριε Μιλάνα, για ένα λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Να σας καλωσορίσω κύριε Δαμανάκη και εγώ με τη σειρά μου. Νομίζω ότι πολλές φορές στον προφορικό λόγο απαντούμε διαφορετικά από ό,τι στο γραπτό. Στην Ευρώπη έχουμε κατανόληση 5 εκατομμυρίων τόνων ετησίως. Ω Ως προς την κατανάλωση τόνου υπάρχουν όμως ορισμένες ελλείψεις στοιχείων και η Επιτροπή μας είπε ότι θα δημοσιοποιήσει τις προθέσεις της σε αυτό το θέμα. Πιστεύετε ότι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειάζεται ένας ειδικό κανονισμός επί του θέματος σε σχέση με την ηχθειοκαλλιέργεια ή θεωρείτε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ειδικό ταμείο επί του θέματος. Κύριε Δαμανάκη για δύο λεπτά. Ευχαριστώ τον κύριο Μιλάνα για την ερώτηση. Το θέμα της ηχθειοκαλλιέργειας, το οποίο θέλω ευθύ εξ αρχής να αναφερθώ, γνωρίζω ότι αποτελεί αντικείμενο μιας έκθεσης, την οποία ετοιμάζεται να υποβάλει και την οποία επίσης έχω δει. Ε, θα ήθελα να πω πολύ καθαρά ότι χρειάζεται να αναπτύξουμε περισσότερο την ηχθειοκαλλιέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρκεί να σας πω ότι αυτή τη στιγμή παράγουμε μόνο 1,2 εκατομμύρια τόνους από ηχθειοκαλλιέργεια το χρόνο και εισάγουμε 5,5. Ε, και ενώ η χθιοκαλλιέργεια στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται με ρυθμό της τάξης τα τελευταία 7 χρόνια 0,1% το χρόνο, σε άλλες χώρες αναπτύσσεται με ρυθμό 7 και 8 το χρόνο. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει κεντρική πολιτική για την ηχθειοκαλλιέργεια, υπάρχουν πάρα πολλές διευθύνσεις οι οποίες αναμειγνύονται στο θέμα αυτό θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να συντονίσουμε την πολιτική των κρατών μελών. Θα επισκεφθώ τα κράτη-μέλη, θα προσπαθήσω να δω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πώς μπορούμε να συνεργαστούμε και θα συζητήσουμε στα πλαίσια του πράσινου βιβλίου το ενδεχόμενο να έχουμε μια κοινή πολιτική για την, ε, και ένα αντίστοιχο χρηματοδοτικό εργαλείο. Αυτά ως πιθανότητα. Μπορείτε να δευτερολογήσετε για μισό λεπτό. Σημερίζεστε την ιδέα ότι υπάρχει ανάγκη σε αυτό το τομέα να γίνει μια άρδιν ε, μεταρρύθμιση του ρυθμιστικού πλαισίου, διότι σήμερα η πολιτική ηχθειοκαλλιέργειας εντάσσεται σε δεκάδες κανονισμών στα πλαίσια εξορθολογισμού πιστεύετε ότι θα πρέπει να έχουμε ένα ενιαίο κείμενο. Για μισό λεπτό κυρία Δαμανάκη. Ναι, τη συμμερίζομαι αυτή την ιδέα. Υπάρχουν πάρα πολλές διευθύνσεις και πάρα πολλές υπηρεσίες οι οποίες ε, ασχολούνται με την ηχθειοκαλλιέργεια. Υγεία, ε, περιβάλλον, μεταφορές. Ασφαλώς δεν θέλει κανείς να υποκαταστήσει τη δραστηριότητα άλλων υπηρεσιών ή άλλων επιτρόπων. Αλλά πρέπει να κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Να υπάρξει μια ενιοποίηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και να υπάρξει μια ενίσχυση του τομέα αυτού. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό έχει το λόγο ο Αντιπρόεδρος κ. Χάγκλουντ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Υποψήφια Επίτροπε. Θα ήθελα να σας ζητήσω να πείτε λίγο περισσότερο για τις απόψεις σας σε σχέση με την σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες τις αλληλευτικές ε, συμφωνίες συγκεκριμένα και τα ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία θέλει να προωθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε παγκόσμιο επίπεδο. Αναφέρομαι κυρίως για τη συμφωνία με τη Γουινέα, την οποία εμείς έχουμε απορρίψει ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο παρελθόν. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η άποψή σας για αντίστοιχα θέματα στο μέλλον και επίσης θα ήθελα να, να έχω την άποψή σας για θηρευτές ε, ηχθείων όπως είναι οι κορμοράνοι και την ζημιά που μπορούν να προξενήσουν στην αλληλευτική δραστηριότητα στην Ευρώπη. Δύο λεπτά κυρία Ταμανάκη. Ευχαριστώ τον κύριο Χάγκλουντ. Να πω καταρχήν για το θέμα της, ε, των διεθνών συμφωνιών, των international agreements, ότι πράγματι χρειάζεται βελτίωση ε, η πολιτική μας και στα πλαίσια της ε, του, ε, συζήτησης για την μεταρρύθμιση είναι ένα κεφάλαιο που το συζητούμε. Οι, αυτές οι συμφωνίες είναι ένα σημαντικό εργαλείο ε, διαθέτουμε πολλά χρήματα, διαθέτουμε 15% του προϋπολογισμού μας κάθε χρόνο για αυτές τις διεθνείς συμφωνίες και επομένως μπορούμε να τις αλλάξουμε έτσι ώστε να έχουμε συγχρόνως και εξυπηρέτηση της, ε, ε, της fishery industry αλλά και εξυπηρέτηση των συμφερόντων των χωρών οι οποίες είναι, ε, βρίσκονται σε ένα καθεστώς πράγματι που πολλές φορές αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες και μεγάλες δυσκολίες επίσης στον τομέα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Καλωσορίζω την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη συμφωνία με τη Γουινέα. Θεωρώ ότι ήταν πολύ σημαντική συμβολή συμβολή του, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην πολιτική μας ε, πολύ σημαντική, το εννοώ και θέλω να πω ότι θα συζητήσουμε την πολιτική μας στο θέμα των συμφωνιών ώστε τα ανθρώπινα δικαιώματα να υπάρχουν ως απαράβατος όρος στα πλαίσια του συνόλου της πολιτικής που ασκούμε. Θέλουμε να συνεχίσουμε αυτή την πολιτική διότι μπορεί να είναι επωφελής για όλους και για την αλληλεία μας και για τις χώρες αυτές οι οποίες μπορούν να επωφεληθούν. Δεν επωφελούνται πάντα για πολλούς λόγους. Πρέπει να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, αλλά μπορούμε και πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την πολιτική. Ευχαριστώ κύριε Χάουγκλοντ. Έχετε 30 δευτερόλεπτα για συμπληρωματικό ερώτημα. Πάρα πολύ σύντομα κυρία Πρόεδρε. Θέλω να σας ευχαριστήσω κυρία Δαμανάκη για τη σαφή σα απάντηση, για τις συμφωνίες με τρίτες χώρες. Θα μπορούσατε να μας πείτε κάτι περισσότερο για τους διώκτες ηχθείων όπως είναι Κορμοράνη. κορμοράνοι. Ίσως το δεύτερο σκέλος που αφορά τις φώκες και τους κορμοράνους. Ε, αυτό δεν είναι, κοιτάξτε να δείτε, το θέμα αυτό δεν είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι θέμα της Κομισιόν. Είναι θέμα που αναφέρεται στα κράτη-μέλη τα οποία προσπαθούν με τον τρόπο που αυτά νομίζουν να το λύσουν. Όμως, όμως, όμως όσον αφορά τις, ε, τις δικές μου δυνατότητες. Αναφέρομαι, γι' αυτό το θέμα αναφέρομαι στους κορμοράνους. Αυτό είναι θέμα των κρατών μελών. Όσον αφορά τις φώκες υπάρχει η πολιτική μας η οποία πραγματικά πρέπει να εφαρμοστεί. Αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι τον επόμενο χρόνο θα έχουμε ίσως τη δυνατότητα να παραγγείλουμε μία μελέτη επιπτώσεων αυτών των καταστάσεων στα πλαίσια της αλληλείας αλλά και του περιβάλλοντος ώστε να πάρουμε τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Υποψήφια Επίτροπε. Είπατε προηγουμένως τα ενακτικά εναρκτήρια σχόλια σας αναφερθήκατε στην αξιοπιστία της πολιτικής μας η οποία διακυβεύεται όταν μιλούσατε για τα θέματα της συμμόρφωσης. Θα μπορούσα να σας, να σας αναφέρω ότι κατά την άποψή μου αυτή η πολιτική δεν έχει καμία αξιοπιστία. Στη Σκωτία έχουμε εμπειρία πάνω από 30 χρόνια με αυτή την ε, πολιτική η οποία οδήγησε μονάχα σε οικονομική κάμψη στις αλληλευτικές κοινότητές μας. Πώς θα μπορούσε να αναστραφεί αυτό το κλίμα στην Σκοτία με τη δική σας πολιτική. Επίσης αναφερθήκατε σε αποκέντρωση, είπατε ότι θέλετε να στοχεύσετε να υπάρχουν ε, λύσεις σε κάθε θαλάσσια λεκάνη που είναι προσαρμοσμένες στην ανάγκη αυτής της θαλάσσιας λεκάνης. Μήπως σημαίνει αυτό ότι τα αλληλευτικά έθνη τα οποία έχουν πρόσβαση σε αυτές τι θαλάσσιες λεκάνες να είναι αυτά τα οποία θα αποφασίσουν πώς θα λειτουργήσει αυτή η πολιτική στο μέλλον. Και αυτό περιλαμβάνει και την διατήρηση των ελευτικών ε, ειδών. Δύο λεπτά, ένα λεπτό, κυρία Δαμανάκη. Με τι απόψει του κυρίου συναδέλφου για την αποτυχία τη ε, αλλιευτική πολιτική. Θέλω απλώ να πω ότι έχουμε και ορισμένε θετικέ εξελίξει. Ορισμένε θετικέ εξελίξει που αφορούν και τη σκοτία. Παραδείγματο χάρη, έχουμε μία, εξαιτία και τη πολιτική μα, ε, μία βελτίωση της κατάστασης που έχουμε στο απόθεμα Northern Hake Εφαρμόζουμε ε, multi-annual plan από το 2004 και ήδη το απόθεμα αυτό βρίσκεται πάνω από τα όρια βιωσιμότητας. Έχουμε καλά αποτελέσματα στην πολιτική για solid and στο Βόρειο Ατλαντικό έχουμε εφαρμόσει μια πολιτική από το 2007 και μέσα σε δύο χρόνια έχουμε πετύχει μια βελτίωση του αποθέματος 40%. Έχουμε κάποια θετικά παραδείγματα. Δεν είναι όλα μαύρα στην εφαρμογή της πολιτικής. Έχουμε καλύτερα αποτελέσματα για τη γλώσσα στο βυσκαϊκό κόλπο. Όμως καταλαβαίνω ότι είναι πολύ σημαντικό για σας οι ψαράδες και η σκοτία να παίρνει μέρος, να αισθάνεται ότι είναι μέρος και ακούεται η άποψή της και ε, λαμβάνεται υπόψη και καταλαβαίνουμε αυτά που λέτε. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε στα πλαίσια της πρότασης για τη μεταρρύθμιση της πολιτικής αυτό που είπα regionalization. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Το ποιοι θα αποφασίζουν σε κάθε θαλάσσια λεκάνη, αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητήσουμε. Αντιλαμβάνομαι ότι εσείς θα θέλατε μόνο τα κράτη-μέλη που έχουν σύνορα στη συγκεκριμένη λεκάνη να μετέχουν. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό. Θα ήταν ουσιαστικά ενάντια στις συνθήκες και θα ήταν ουσιαστικά μια, ε, ένα, θα δημιουργούσε ένα πρόβλημα στο κατά πόσο κοινή είναι η πολιτική μας. Αλλά θα το συζητήσουμε και αυτό. Ε, όλα τα θέματα θα συζητηθούν και θα βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση. Ε, Έχετε δικαίωμα να δευτερολογήσετε για 30 δευτερόλεπτα. Δεν νομίζετε ότι θα ήταν λογικό να μην θέσουμε ένα αμφιβόλο κοινέ πτυχές της πολιτικής εάν δεν ήταν αποδοτικές όπως αποδείχτηκε. Δεν είναι δύσκολο να εξηγήσετε στις αλλιευτικές κοινότητες ότι πρέπει να δράσουμε κατά ένα συγκεκριμένο τρόπο διότι έτσι ορίζει η συνθήκη. Δεν δεχόσαστε ότι η ρόλος σας είναι να τονίζετε από καιρού εις ότι ίσως η συνθήκη, στη συνθήκη έγκυται το πρόβλημα. Κυρία Δαμανάκη, για 30 δευτερόλεπτα. Είμαι υποχρεωμένη να σεβαστώ απολύτως τη συνθήκη. Αλλά η ίδια η συνθήκη προβλέπει, η ίδια η συνθήκη προβλέπει ότι η πολιτική τίθεται συνολικά σε συζήτηση. Και αυτό κάνουμε. Όχι απλώς ορισμένες ε, πλευρές που δεν έχουν επιτύχει, αλλά με βάση τη συνθήκη θέτουμε όλη την πολιτική μας σε συνολική πρόταση αναδιαπραγμάτευσης. Αυτό είναι το νόημα του πράσινου βιβλίου. Μιλούμε συνολικά για CFP reform. Άρα λοιπόν θα τα συζητήσουμε όλα με αυτό το πνεύμα. Ευχαριστώ πολύ. Με ανακούφιση ακούω σκοπεύετε να προχωρήσετε στη μεταρρύθμιση τη κοινή αλληλευτικής πολιτικής και ιδιαίτερα με τι πτυχέ τη αποκέντρωση, τη περιφερειοποίηση ε, για τη λήψη αποφάσεων με συμμετοχή των ίδιων των εμπλεκομένων φορέων. Στο, στη συνθήκη του Άμστερνταμ και το πρωτόκολλο με την, για την επικουρικότητα ε, ρητά αποκλείεται η αποκέντρωση και η περιφερειοποίηση προς τα κράτη-μέλη. Πώς θα αντιμετωπίσετε αυτό το εμπόδιο και πώς θα φροντίσετε ε, ή καθημερινή λειτουργία της αλίας να μην μετατραπεί σε μικροδιαχείριση, micromanagement, που ήταν καταστροφική από πλευράς του Η κυρία Δαμανάκη για δύο λεπτά. Ε, οι συνθήκες προβλέπουν ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε επανεθνικοποίηση της πολιτικής μας και γι' αυτό ήμουν πολύ σαφής ευθύ εξ αρχής προσπαθώντας να κάνω διάκριση ανάμεσα στο ενδεχόμενο επιστροφής αρμοδιοτήτων στα κράτη-μέλη και αυτό που εγώ ονομάζω regionalization και ονομάζεται και στην Πράσινη Βίβλο και στις σχετικές εκθέσεις regionalization των αποφάσεων. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά θέματα. Δεν υπάρχει θέμα επιστροφής αρμοδιοτήτων στα κράτη-μέλη. Αλλά υπάρχει θέμα να έχουμε δυνατότητα ώστε λεπτομέρειες των αποφάσεών μας να λαμβάνονται σε τοπικό επίπεδο ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη συμμετοχή. Αυτό προβλέπεται από τις συνθήκες ε, οι νομικοί μας λένε ότι μπορούμε να το κάνουμε, γι' αυτό έχει μπει και στο πράσινο βιβλίο και γι' αυτό κάνουμε όλο αυτό το διάλογο για το ποιος, πώς θα το πετύχουμε. Αλλά συμφωνώ μαζί σας, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην κατεύθυνση της επιστροφής ε, αρμοδιοτήτων ε, στα κράτη-μέλη. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Μπορείτε να μας καθησυχάσετε, κυρία Δαμανάκη ότι δεν θα εφαρμόσετε σύστημα uniform ε, στη διαχείριση στα νέα σας αυτά καθήκοντα που να ασχεί για όλους δηλαδή. Ε, εσείς ο ίδιος είπατε πριν ότι πρέπει να αποφύγουμε το micromanagement και συμφωνώ Λέτε όμως και συμφωνώ επίσης ότι δεν πρέπει να εφαρμόσουμε ένα σύστημα uniform, αλλά πρέπει να έχουμε tailor-made solutions. Tailor-made solutions for uh, integrated tailor-made solutions for uh, για τις ε, ειδικέ περιπτώσεις και για τις θαλάσσιες λεκάνες. Ό,τι μπορεί. Χωρίς ε, λοιπόν στρατιωτικές ε, υποχρεωτικές νόρμες, αλλά χωρίς να φτάσουμε και στο επίπεδο του micromanagement. Θέλω πραγματικά, αισθάνομαι ότι αυτό θα είναι ένα δύσκολο ταξίδι και θέλω να αναζητήσω μαζί σας τις καλύτερες δυνατές λύσεις. Ε, Ευχαριστώ. Ο κύριος Φεραίρα πάλι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε κύριος Φεραίρα. Για το θέμα της αποκέντρωσης. Είπατε κυρία υποψήφια επίτροπε ότι είσαστε εναντίον μια επανεθνικοποίηση τη κοινή αλληλευτική πολιτική και υποστηρίζετε μια κοινή πολιτική αλλία. Αλλά γνωρίζοντας όπως γνωρίζουμε ότι ένα πράγμα είναι η πολιτική και κάτι άλλο είναι το κόστος αυτής της πολιτικής, ποιες είναι οι απόψεις σας για τον κίνδυνο να επανεθνικοποιηθεί το κόστος της κοινής αλληλευτικής πολιτικής. Κυρία Δαμανάκη, έχετε λόγια για ένα λεπτό. Ε, μίλησα για την ανάγκη να υπάρξει κοινή πολιτική και πραγματικά πιστεύω ότι το ευρωπαϊκό οικοδόμημα έχει τις προβλέψεις και τις διασφαλίσεις ώστε να υπάρχει δίκαιη κατανομή και βαρών σε όλους. Ε, υπερασπίζομαι αυτό το ευρωπαϊκό οικοδόμημα εδώ και πολλά χρόνια και νομίζω ότι έχουμε τις διασφαλίσεις. Στα πλαίσια άλλωστε της εφαρμογής της collegiality θα στηρίξω όλες τις αποφάσεις των επιτρόπων των αρμοδίων για το θέμα αυτό. 30 δευτερόλεπτα δευτερολογία κύριε Φεραίρα. Το ερώτημά μου σε συγκεκριμένο επίπεδο πώς θα αντιμετωπίσετε τις απειλές να μειωθούν τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλίας και επίσης στα πλαίσια της αποκέντρωσης τι πιστεύετε στο να δοθεί μόνιμος χαρακτήρας σε αυτό το οποίο το 2002 είχε θεωρηθεί μια προσωνή ρύθμιση, δηλαδή να παραμείνει η περιοχή παράκτια μέχρι 12 μίλια για τους αλληλείς κάθε κράτους και εάν θα πρέπει να επεκταθεί αυτή η, αυτός ο περιορισμός στην υφαλοκρηπίδα και πέραν των 12 μιλίων. Δηλώσει τον απόλυτο σεβασμό της στο δίκαιο της θάλασσας. Αυτόν τον σεβασμό θέλω και εγώ από αυτό το βήμα να ε, επαναδηλώσω. Ε, υπάρχουν διαφορετικές, διαφορετικά καθεστώτα στις διάφορες χώρες. Στη Μεσόγειο έχουμε κυρίως ε, αυτό το σύστημα όπου η ζώνη ελίας των χωρών είναι 12 και μερικές φορές 6 μίλια θα μπορούσα να πω αλλά υπάρχουν και άλλες χώρες όπου έχουν τις exclusive economic zones τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες που είναι 200 μίλια. θα γίνει σεβαστή η εξωτερική πολιτική της κομισιόν. Ε, Ευχαριστώ. Ο τελευταίος παρεμβαίνων σε αυτό το δεύτερο γύρο, ο κύριος Σαλαβράκος. Για ένα λεπτό, έχετε το λόγο. Κύριε Δαμονάκη, θεωρώ ότι η παρουσία σας εδώ ήταν πολύ ικανοποιητική και παρά το γεγονός ότι είμαστε σε διαφορετικούς πολιτικούς χώρους στην Ελλάδα δεν έπαψα ποτέ να θαυμάζω ε, την τελειότητα του μυαλού σας και των θέσεων όπως τις διατυπώνετε. Θα ήθελα να σας κάνω ένα ερώτημα ε, σχετικά με τη Μεσόγειο θάλασσα την οποία μοιράζονται πολλές χώρες μερικές από τις οποίες δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιπλέον δεν υπάρχουν αποκλειστικές οικονομικές ζώνες και ανοιχτές θάλασσες έτσι ώστε να ισχύουν τα σχετικά με τα 6 ή τα 12 μίλια των θαλασσίων συνόρων. Πώς σας διασφαλίσετε εσείς σαν Επίτροπος ισότιμες συνθήκες μεταξύ των ψαράδων μας που είναι υποχρεωμένοι να υπακούν σε λεπτομερή και αυστηρή νομοθεσία και των άλλων συναδέλφων τους που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν υπόκειται στους ίδιους κανόνες αλλά συχνά ψαρεύουν παρανόμως και μπροστά στην πόρτα των δικών μας ψαράδων. Δύο λεπτά κυρία Δαμανάκη. Άδελφο για τα καλά του λόγια. Ε, το πρόβλημα που θέτει είναι πράγματι πολύ σοβαρό. Ε, αφορά την Ελλάδα, αλλά όχι μόνο την Ελλάδα. Αφορά πολλές μεσογειακές χώρες, διότι πάρα πολλές μεσογειακές χώρες έχουν ε, οι ψαράδες μας σε πολλές μεσογειακές χώρες έχουν να αντιμετωπίσουν ένα unfair competition, ένα, πλαίσιο ενός μη υγιούς ανταγωνισμού, με δεδομένο ότι, όπως ξέρετε, στη Μεσόγειο δεν είμαστε μόνο εμείς, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πάρα πολλές χώρες, πάρα πολλές άλλες χώρες, ε, οι οποίες ε, δεν έχουν, αν θέλετε, την ίδια έτσι, διάθεση να συμμορφωθούν στους διεθνείς κανονισμούς αλλιές. Πώς μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Καταρχήν θέλω να πω ότι ο μόνος τρόπος, καλύτερος τρόπος είναι ο διάλογος και η προσπάθεια να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε. Ε, όπως ξέρετε η Ευρωπαϊκή Ένωση μετέχει στα όργανα της Μεσογείου που διαχειρίζονται την αλία της Μεσογείου, μετέχει και στο ICAT, μετέχει και στο GFCM, δηλαδή στην Επιτροπή για τη Μεσόγειο, την Αλλιευτική Επιτροπή για τη Μεσόγειο, όπου μετέχουν και όλες οι χώρες της Μεσογείου και η Τουρκία στην προκειμένη περίπτωση. Σημασία έχει εκεί να υπάρξουν μέτρα πίεσης ώστε να γίνει απολύτως σαφές ότι οι κανονισμοί πρέπει να τηρούνται από όλους από όλους. Και να γίνει επίσης σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ψαριών στον κόσμο, ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ψαριών στον κόσμο, δεν μπορεί να εισάγει προϊόντα παράνομης αλίας. Δεν μπορούν να έχουν IUU products πρόσβαση σε εμά. Εφαρμόζουμε τους κανονισμούς. Ανάγκη λοιπόν είναι στα διεθνή αυτά πλαίσια να βρούμε την καλύτερη ε, λύση ε, για όλους, έτσι ώστε πραγματικά να προστατευθούν οι δικοί μας ψαράδες. Και αυτό θα προσπαθήσω με ό,τι δυνάμεις διαθέτω να το επιτύχω. Κατά τα άλλα, ελπίζω να εφαρμοστεί το δίκαιο της θάλασσας σε όλη τη Μεσόγειο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με ειρηνικό τρόπο, ώστε να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα και για την αλληλεία μας. Ευχαριστούμε κύριε Δαμανάκη. Ο κύριο ε, Καλαβράκο θέλει να δευτερολογήσει ή όχι. Ευχαριστώ. Α, perfecto. Θαυμάσια σα Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε με τον ε, κύριο Κατέκ. Ευχαριστώ. Σα καλωσορίζω κυρία Δαμανάκη και εγώ με τη σειρά μου θεωρώ ότι θα ήταν απαράδεκτο να έχουμε μεμονωμένες μεταβιβάσιμες ποσοστώσεις για τη βιοτεχνική αλία. Στη Βρετάνη οι αλίες φοβούνται αυτή την πιθανότητα. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να έχουμε άμεση ανάθεση και απόδοση ποσοστώσεων. Στα πλαίσια της συνθήκης της Λισαβόνας είσαστε υπέρ μίας, ενός νέου ορισμού της βιοτεχνικής αλίας διαμέσου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έτσι ώστε να μπορέσει να επιβιώσει η βιοτεχνική αλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρία Δαμανάκη, για δύο λεπτά. Ε, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Καντέκ για την ερώτησή του. Ε, πράγματι, το θέμα της μεταβίβασης των ποσοστώσεων, αυτό που λέμε ITQ system και transferable quotas, για να συνοηθούμε, διότι ορισμένοι έτσι το καταλαβαίνουν, είναι ένα δύσκολο θέμα και καταλαβαίνω την ανησυχία που ε, ανέφερε για τους ψαράδες της Βρετάνης. Είπα και πριν, και μια και έχω λίγο χρόνο θέλω να το επαναλάβω, ότι υπάρχουν χώρες μέλη που το ε, εφαρμόζουν αυτό το σύστημα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να εφαρμοστούν ε, προϋποθέσεις και περιορισμοί στο σύστημα αυτό. Και υπάρχουν τέτοιοι μηχανισμοί. Παραδείγματο χάρη η Δανία δεν επιτρέπει να μεταβιβάζεται το δικαίωμα το ατομικό, παρά μόνο στα πλαίσια της μικρότερης αλίας. Δεν επιτρέπεται προς, μεγαλύτερε προς μεγαλύτερες βιομηχανίες να μεταβιβαστεί. Υπάρχουν επίσης όρια, 5%. Μπορούμε να βρούμε μηχανισμούς. Και νομίζω ότι τα κράτη-μέλη τα οποία προς το παρόν χειρίζονται το θέμα μπορούν να βρουν τον καλύτερο ε, τρόπο και εμείς βεβαίως θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια ώστε αυτό που λέμε small scale fisheries να προστατευτεί. Συμφωνώ με τον κύριο Καντέκ χρειάζεται ένας επίσημος ορισμός του τι εννοούμε όταν λέμε small scale fisheries. Και αυτό είναι ένα θέμα που θα το συζητήσουμε στα πλαίσια του CFP ε, reform, διότι υπάρχουν διάφορα στοιχεία τα οποία πρέπει να συνυπολογιστούν. Υπάρχει το μήκος του σκάφους, εμείς φάζουμε ως όρο να μην έχει σειρώμενα εργαλεία και πιστεύω το καταλαβαίνετε αυτό. Υπάρχει όμως επίσης και το θέμα της ιδιοκτησίας. Εάν δηλαδή κάποιος έχει πάρα πολλά μικρά σκάφη, εκατοντάδες, αυτό πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη. Άρα συμφωνώ, πρέπει να συζητήσουμε το θέμα, να προχωρήσουμε σε ένα ορισμό αυτού που λέμε small scale fishery και να εξασφαλίσουμε τις καλύτερες δυνατούς όρους γι' αυτό. Ο κύριος Καντέκ, ε, δευτερολογία. Υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα το οποίο έχουμε θίξει αρκετές φορές. Υπάρχει μια αντίφαση μεταξύ της βιώσιμης συνολικής διαχείρισης και του ανοίγματο της παγκόσμιας αγοράς. Το 60% των ε, ε, αλλιευτικών προϊόντων που καταναλώνουμε προέρχονται από τρίτες χώρες. Πώς μπορούμε να προωθήσουμε την ε, εμπορία των δικών μας αλλιευτικών προϊόντων και πώς μπορούμε να ορίσουμε κανόνες υγείας και υγιεινής για τα εισαγόμενα προϊόντα. Κανόνες που δεν τηρούνται πάντα μέχρι τούδε. Κυρία Δαμανάκη. Μα πιο σκληρά από τα δικά σας λένε ότι το 70% των εισαγωμένων των προϊόντων που καταναλώνουμε είναι εισαγόμενα. Άρα υπάρχει σοβαρό θέμα το οποίο θέτεται με την ερώτησή σας. Θα έλεγα ότι μπορούμε να είμαστε και αμυντικοί και επιθετικοί. Είμαστε αμυντικοί διότι έχουμε τον καλύτερο κανονισμό για τις συνθήκες υγιεινής για τα ψάρια, τον οποίο εφαρμόζει η αρμόδια, επιτροπή, η αρμόδια διεύθυνση υγείας. έχουμε αρκετά καλούς κανονισμούς στο θέμα του trade, στο θέμα του εμπορίου και μπορούμε να επιμείνουμε ώστε κανένα προϊόν παράνομης αλίας με βάση το IUU control να μην μπαίνει στη χώρα μας. Από εκεί και πέρα Υπάρχει θέμα και επιθετικής πολιτικής και αναφέρομαι στο labeling και eco-labeling των προϊόντων μας. Είναι πολύ σημαντικό ο Ευρωπαίος καταναλωτής να ξέρει ότι αυτό το οποίο τρώει έχει ψαρευθεί στα πλαίσια μιας υγιούς ε, αλίας που συμβάλλει στην αηφορία. Αυτό είναι μεγάλο όπλο και σκοπεύω να το χρησιμοποιήσω. Ε, Ευχαριστούμε πολύ. κυρία για ένα λεπτό. Καλημέρα και να σας καλωσορίσω και σας εύχομαι συγχαρητήρια. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μεγάλες προκλήσεις γιατί μιλάμε για αλία και για βιωσιμότητα. Βρισκόμαστε σε κατάσταση παγκόσμιας κρίσης. Μιλήσατε για την αξιοπιστία του τομέα ε, ενώπιον της ε, μεταρρύθμισης πιστεύετε ότι θα, θα μπορούσαμε να φτάσουμε στους στόχους της μελλοντικής αλληλευτικής πολιτικής με βάση τον ε, ενδελεχή έλεγχο. Πιστεύετε ότι μπορούμε, να, μπορούμε ε, να προωθήσουμε θέματα συμφωνίας και με βάση εκδημοκρατισμό τρίτων χωρών με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Επίσης, ο ρόλος της γυναίκας στην αλληλευτική πολιτική μπορείτε να αναφερθείτε σε αυτό το ρόλο. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε να απαντήσετε και στις τρεις ερωτήσεις, ε, κυρία Πίτροπε, παράλληλα. Ξεκινήσω από τις γυναίκες. Αν ε, δεν έχουμε χρόνο, τουλάχιστον έχω πει κάτι γι' αυτό. Ε, ζήτησα τα στοιχεία, γιατί πραγματικά είχα ένα ενδιαφέρον. δεν έχουμε πάρα πολλές γυναίκες ψαράδες. Έχουμε 4% περίπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε όμως συνολικά 26% στο σύνολο του τομέα, διότι έχουμε πάρα πολλές γυναίκες οι οποίες, οι ασχολούνται στη βιομηχανία, στο processing industry, στη μεταπητική βιομηχανία. Ε, οι γυναίκες θέλουν να συμμετέχουν ήδη ορισμένες από αυτές ε, στα RACS και θέλουν καλύτερη συμμετοχή. Έχω μάλιστα έρθει σε επαφή με ορισμένες γυναικείες οργανώσεις, οι οποίες ζητούν ένα καθεστώς καλύτερο ε, από αυτό το οποίο έχουν. Και στα πλαίσια της αναμόρφωσης των συμβουλίων θα πρέπει να το δούμε. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα θέματα, συμφωνώ ότι η κρίση έχει επηρεάσει και την αλληλεία, έχει επηρεάσει τις τιμές των προϊόντων, χωρίς αμφιβολία, και έχει μειώσει την κατανάλωση σε κάποιες χώρες. Ε, πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα προστατεύσουμε κατά το δυνατόν, διότι δεν μπορούμε να αποστούμε από την πολιτική της Κομισιόν, ε, τους πιο αδύνατους, δηλαδή τα small scale fisheries και τους αυτούς που πραγματικά δεν έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν, με εργαλεία μοντέρνα που θα είναι συμβατά με το κοινοτικό δίκαιο. Για τον εκδημοκρατισμό στις ε, συμφωνίες με τις τρίτες χώρες συμφωνώ απολύτως. Ευχαριστώ. Ήσασταν ε, πάρα πολύ γρήγορες στην απάντησή σας. Θα ήθελα να σας μιλήσω για το εξής. Μιλήσατε για ένα μετρήσιμο μέγεθος που είναι η πραγματική αλληλευτική πολιτική και ο αλληλευτικός στόλος. Πώς μπορούμε να κάνουμε πιο ορατό το ρόλο των γυναικών. Μου βάζετε δύσκολα αλλά πρέπει να το δοκιμάσουμε. Ξέρουμε ότι έχουμε 88.000 σκάφη, ξέρουμε ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά για το στόλο, δεν ε, έχουμε βρει πολύ συγκεκριμένα στοιχεία για το πώς προσδιορίζεται αυτό που λέμε over capacity, σε αυτό το θέμα θέλω να είμαι ειλικρινής. Ε, και συνήθως συγκρίνουμε και ε, σχηματίζουμε εντύπωση για το overcapacity σε σχέση και με τα διαθέσιμα αλλιεύματα. Θέλω να εισαχθεί η λογική του ex post assessment στην πολιτική αλλίας. Αυτό μόνο μπορώ να πω. Στη συνέχεια το λόγο έχει και για δύο λεπτά ο κύριος Ρέιμερς. Η κυρία Ράιμερς, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κυρία Δαμανάκη, το σύστημα ελέγχου των ε, αλλιευτικών μεθόδων και ποσοτήτων μέχρι στιγμής δεν έχει εξασφαλίσει τους επιδιωκόμενους στόχους. Ως εκ τούτου εγώ θα θεωρούσα πολύ πιο σκόπιμο να εμπλακεί ο ίδιος ο αλλιέας και ενδεχομένως με σύστημα κινήτρων, κυρώσεων ε, να τον πείσουμε, να τον φέρουμε μέσα στο σύστημα έτσι ώστε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Και γι' αυτό ερωτώ τι είδους κίνητρα θα μπορούσε ενδεχομένω να προβλέψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να τηρούνται οι προϋποθέσεις, οι ε, προδιαγραφέ της κοινή αλλιευτική πολιτικής από τους αλληλεί και πώς θα μπορούσε αυτή την ανακοίνωση να την ε, εφαρμόσει καλύτερα η Επιτροπή. Συμφωνώ με την κυρία Ρέιμερς ότι κάποιος ο οποίος μετέχει στη λήψη μιας απόφασης ε, είναι πιο εύκολο να την εφαρμόσει, είναι πιο πρόθυμος να την εφαρμόσει. Άρα πρέπει να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το τομέα. Στα πλαίσια όμως των συνθήκων. Ε, μιλήσατε για κίνητρα. Κίνητρα υπάρχουν ως λογική στην πολιτική μας. Σας είπα ήδη ότι ο νέος κανονισμός για τη συμμόρφωση, το IUU Regulation, προβλέπει ουσιαστικά ένα point system, δηλαδή προβλέπει να, υπάρχουν, να υπάρχει λογική των κινήτρων στις ποινές και στις, ε, στην όλη λογική του συστήματος συμμόρφωσης. Προβλέπει επίσης ότι αν κάποιος για ένα διάστημα, αν υπάρχει μια ορισμένη ποινή και αν κάποιο για ένα διάστημα συμμορφωθεί, μπορεί να αναιρεθεί αυτή η ποινή. Έχουμε πάει δηλαδή ακόμα παραπέρα. Υποθέτω όμως ότι κυρίως ενδιαφέρεστε ε, για κίνητρα στα πλαίσια των tax and quotas και, των, ε, και της εφαρμογής των αλλιευτικών εργαλείων πολιτικής. Τι μπορώ να πω γι' αυτό. Εμείς καθορίζουμε γενικά το ε, τάκ, της ποσόστοση που αντιστοιχεί σε κάθε κράτος μέλος. Τα κράτη-μέλη μπορούν να εφαρμόσουν τέτοιου είδους κίνητρα και ορισμένες χώρες ήδη το εφαρμόζουν. Εμείς θα ενισχύσουμε την πολιτική των κινήτρων ώστε ο ψαράς που ψαρεύει μέσα στα πλαίσια των κανονισμών να αμείβεται ανάλογα. Θέλετε να θέσετε συμπληρωματικό ερώτημα, κύριε Ρέιμερς, όχι. Ευχαριστώ. Στη συνέχεια, επειδή έχουμε και το χρόνο, θα είμαι λίγο πιο χαλαρή. Δεν θέλω να καταχραστείτε όμως της καλής μου θέλησης. Λοιπόν, θα δώσουμε και περισσότερο χρόνο λοιπόν στους ε, τελευταίους ομιλητές και η κυρία Πίτροπος στο τέλο τη παρέμβασή τη, θα έχει λίγο περισσότερο χρόνο γιατί έχουμε κερδίσει χρόνο. Ο κύριο Βαλέσα για ένα λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Δαμανάκη, είμαι Πολωνός από το Γκτάνσκ της Βαλτικής και γι' αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής για τη συγκεκριμένη αυτή περιοχή. Η Αλία στη Βαλτική, στην Πολωνία, έχει 900 περίπου μεγάλα και 400 περίπου μικρά σκάφη. 2.000 θέσει εργασία λίγο πολύ και επιπλέον ανά Αλία 7 περιφερειακές θέσει εργασία από τον αλλιευτικό τομέα. Άρα εξαρτώμεθα σε μεγάλο βαθμό από την αλία του γάδου της Βαλτική. Το, τα προγράμματα προστασίας όμως ε, δεν έχουν φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα και έτσι διαρκώ μειώνονται τα αποθέματα γάδου στη Βαλτική. Πώ θα μπορούσατε να προβλέψετε και τι είδου μέτρα θα μπορούσατε να προβλέψετε έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η επιλεκτική αλία γάδου και βέβαια τι μέτρα προστασία για τι νέε γενναίε. Καταλαβαίνω την ιδιαιτερότητα της Βαλτικής και τη σημασία της αλίας για την πολωνική οικονομία που έθεσε ο κύριος Βαλέσα. Ε, ε, είναι όμως ανάγκη να δούμε και το μέλλον της Βαλτικής. Και το μέλλον της Βαλτικής, όπως και το μέλλον της πολωνικής αλίας, εξαρτάται από το κατά πόσο υπάρχουν επαρκή αποθέματα, ώστε οι αλλήλει να μπορούν να ζήσουν. Αυτές οι θέσεις εργασίας να διασφαλιστούν και για το μέλλον. Αναφερθήκατε στο πρόγραμμα του, του Baltic Code, του, του του Γάδου. Είναι ένα multi-annual πρόγραμμα που έχουμε, είναι μακρόχρονο πρόγραμμα, το οποίο μόλις τώρα έχει αρχίσει να αποδίδει. Ε, μόλις τώρα έχει αρχίσει να αποδίδει. Ε, ζήτησα τα στοιχεία, είναι απλώς ενθαρρυντικά. Κατά συνέπεια δεν μπορούμε να πάμε σε μια λογική απότομης ε, ανόδου των ποσοστώσεων. Ούτε μπορούμε να πάμε σε μια λογική ε, επανόδου ε, της χρήσης του εργαλείου αυτού του DRAFNET, του DRIFNET στη Βαλτική, γιατί όπως καταλαβαίνετε θα έχουμε πολύ μεγάλες συνέπειες σε άλλα είδη, όπως είναι τα θηλαστικά, όπως είναι τα πόρποϊζης, τα μικρά δελφίνια που υπάρχουν στη Βαλτική και που προστατεύονται από την Ατούρα 2000. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μία ισορροπία και αυτό που έχω να πω είναι ότι η ισορροπία αυτή μπορεί να βρεθεί και στο τοπικό συμβούλιο, στο οποίο η Πολωνία μετέχει και πολύ ζωηρά από ό,τι γνωρίζω, έτσι ώστε οι προτάσεις εκεί να συζητούνται και να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θα επιμείνουμε στα προγράμματα, ε, multi-annual ε, προγράμματα για το γάδο της Βαλτικής. ερώτημα. Ε, πάρα πολύ σύντομα κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή της κυρίας Υποψηφίου Επιτρόπου στο πρόβλημα το οποίο απορρέει από το ερώτημά μου, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί από όλους. Το γεγονός ότι ε, αλλιεύονται γάδι σε πολύ νεαρή ηλικία και γνωρίζει και η κυρία Επίτροπος ότι είναι ένα πρόβλημα αυτό. Είναι ότι δεν υπάρχει αρκετά επιλεκτικό το, επιλεκτικά τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε. Δεν είχα το χρόνο να απαντήσω στο συγκεκριμένο σκέλος και είναι πολύ σημαντικό. Συμφωνώ. Πρέπει λοιπόν αυτό το οποίο να κάνουμε είναι να επιδοτήσουμε συγκεκριμένα, να βοηθήσουμε οικονομικά στη Βαλτική τη χρήση εργαλείων που εξασφαλίζουν μεγαλύτερη ε, επιλεξιμότητα, selectivity εννοώ εδώ, ε, ε, ώστε τα μικρότερα τα μικρότερα είδη να μπορούν να διαφεύγουν από τα εργαλεία αυτά. Πρέπει επίσης να δούμε την ανάγκη να υπάρξουν προστατευόμενες περιοχές και απαγόρευση της ελίας για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αυτό το έχουμε δει, το διάστημα δηλαδή που τα μικρά κυκλοφορούν. Ε, αυτά, όλα θα πρέπει να, θα, αυτά όλα θα πρέπει να τα κάνουμε σε συνδυασμό. Ευχαριστώ. Στη συνέχεια έχει το λόγο για ένα λεπτό κύριο Σαρσένης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Δαμανάκη, σας γνωρίζω όπως όλοι και οι πολίτες της Ελλάδας για... ως ένα σύμβολο της δημοκρατίας, αλλά και μια πολιτικό με μεγάλη εμπειρία και μεγάλη προσφορά. Βλέπω σήμερα μπροστά μου έναν άνθρωπο με βαθιά γνώση των θεμάτων αλίας, έτοιμο να αναλάβει μια θέση ευθύνη τόσο απέναντι στου Ευρωπαίου πολίτε, όσο και απέναντι στι γενιέ που έρχονται. Η μεγάλη πρόκληση τη θητεία σα θα είναι η μεταρρύθμιση τη κοινή αλληλευτική πολιτική. Πολλά συζητήσαμε ε, στα πλαίσια της σημερινής ε, ακρόασης. Είναι γνωστό ότι η μεταρρύθμιση θα επικεντρωθεί ε, στη μείωση του ελευτικού στόλου και στη μείωση της συνολικά επιτρεπόμενων αλλοιωμάτων. Αυτό ε, ιδίως σε παράκτητες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου η αλληλεία είναι σημαντικό τμήμα της, ε, στο μέσα και εισοδήματος ενδεχομένως να έχει σημαντικές ε, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Θεωρείται ότι οι αλληλείς σε αυτές τις περιοχές θα πρέπει να τύχουν ειδικών ρυθμίσεων, μέτρων, προγραμμάτων, προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τι αρνητικέ επιπτώσει τη μεταρρύθμιση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Ε, δεν είμαι όπως καταλαβαίνετε ειδική στην Αλία και ούτε έχω την πείρα που έχετε εσείς. Ε, κάνω προσπάθεια να ενημερωθώ και με βοήθησαν πολύ και η διεύθυνση και η Πρόεδρος και ο προηγούμενος Επίτροπος, ο κύριος Μπόρτς, πρέπει να πω, ήταν πολύ βοηθητική στις πληροφορίες τους. Μπαίνω κατευθείαν στο θέμα γιατί είναι πολύ σοβαρό. Πράγματι θα υπάρξουν κοινωνικές επιπτώσεις. Πώς μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Είχα μια πολύ αναλυτική συζήτηση με τον συνάδελφο Commissioner Designate των κοινωνικών θεμάτων. Ε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να υπάρξουν χρηματοδοτήσεις από, τα, από το Κοινωνικό Ταμείο για τα θέματα αυτά. Χρηματοδοτήσει σε ανθρώπου που θα αναγκαστούν ίσω να εγκαταλείψουν τη δουλειά του. Δεν θα είναι εύκολο γιατί για του ψαράδε δεν είναι εύκολο να τους πει εγκατάλειψε τη δουλειά ούτε είναι εύκολο να του πει να σε εκπαιδεύσουμε ώστε να κάνει μια άλλη δουλειά. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να αυξήσουμε τη χρηματοδότηση και τη βοήθεια σε ανθρώπου που ενδεχομένω θα πληγούν. Πρέπει επίσης να, να δούμε το ενδεχόμενο να υπάρξουν συστήματα συνταξιοδότησης νωρίτερα Αυτά κοστίζουν, δεν είναι στη δική μου αρμοδιότητα, ούτε είναι καν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής, είναι στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Παίρνοντα υπόψη όμως τον διαχωρισμό όλων αυτών των αρμοδιοτήτων, και εδώ θέλω να είμαι σαφής, θα σεβαστούμε τις συνθήκες και η νομική υπηρεσία θα είναι απόλυτη και θα βοηθήσει, πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για αυτές τις περιοχές. Νομίζω ότι κυρίως Πρέπει να τους δώσουμε τη δυνατότητα πάντως να ασκούν αυτό το επάγγελμα του ψαρά τουλάχιστον οι μεγαλύτερες ηλικίε. Για τους νεότερους μπορούμε να δούμε την εκπαίδευση με ένα καλύτερο δυνατό τρόπο και το ενδεχόμενο να έχουν ένα δίπλωμα, ίσως υπάρχουν εδώ ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αυτική εκπαίδευση, με το δίπλωμα του Maritime Excellence. Ε, θέλω κλείνοντας να πω ότι θεωρώ ότι σε αυτόν τον διάλογο πρέπει να μετέχουν εκτός από τις περιοχές και, τους, ε, και τις οργανώσεις των παραγωγών και τα συνδικάτα των περιοχών. Υπάρχουν ε, συνδικάτα που εκφράζουν εργαζόμενους στην Αλία. Μέχρι τώρα δεν έχει συνεργαστεί η διεύθυνση αρμόδια με, ε, αυτά τα συνδικάτα. Πρέπει να ανοίξουμε διάλογο και με τα συνδικάτα αυτά. Θέλετε κυρία Σένη. Πολύ για την απάντηση. Ε, μια δύσκολη ερώτηση. Πραγματικά και σήμερα η η μείωση των ελαιωμάτων οφείλεται στην υπεραλίευση και στις μη βιώσιμες αλληλευτικές πρακτικές. Το μέλλον η κλιματική αλλαγή αναμένεται να επιδεινώσει περαιτέρω το αλληλευτικό απόθεμα. Αν και είναι δύσκολο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σα, τι μέτρα προτίθεστε να λάβετε προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσει τη κλιματική αλλαγή στα αλλιεύματα και στη ζωή στη θάλασσα. Ε, αυτό είναι ένα θέμα που πραγματικά δεν το έχουμε μελετήσει επαρκώς. Δεν έχουμε δηλαδή επαρκή επιστημονικά στοιχεία. Ε, δεν, έχουν, δεν έχουμε επαρκή επιστημονικά στοιχεία. Is the Λέω ότι δεν έχουμε επαρκή επιστημονικά στοιχεία ώστε να μπορούμε πώς επιδρά αυτή τη στιγμή η κλιματική αλλαγή στις θάλασσες και τους ωκεανούς μας. Έχω μία ε, πολύ αναλυτική συνεργασία με την Ιρλανδέζα Επίτροπο, η οποία θα είναι αρμόδια για την έρευνα και έχουν προβλεφθεί, όπως ήδη είπα, περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ στο 7ο πρόγραμμα, αυτό το πρόγραμμα ευνών, ένα μεγάλο πρόγραμμα από αυτά, είναι 35 ίσως εκατομμύρια, ένα μεγάλο πρόγραμμα, αν θυμάμαι καλά, είναι γύρω στα 10,5 εκατομμύρια ευρώ, έχει αυτό ακριβώς το περιεχόμενο. Αναφέρεται στην επίδραση που θα έχει η κλιματική αλλαγή στις θάλασσες και την, ε, τις ε, συνακόλουθες επιπτώσεις και στα θέματα της αλίας και στα θέματα τα κοινωνικά και οικονομικά στις παράκτιες περιοχές. Ελπίζω να έχουμε τη μελέτη και να μπορούμε να προχωρήσουμε. Μέχρι τότε θα στηριχθούμε σε όποια επιστημονική συμβολή διαθέτουμε από τις μελέτες που εμείς ως ε, Διεύθυνση Αλίας έχουμε με, τα επιστημονικά σώματα τα οποία συνεργαζόμαστε και τα οποία γνωρίζετε, το ISIS e και, το... και τη Scientific Committee την οποία διαθέτουμε. Για να τελειώσουμε με τον τέταρτο γύρο, ο κύριος Ντέιβις έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υποψηφία Επίτροπε, Προσπαθούμε να βελτιώσουμε τα αλληλευτικά αποθέματα με την αναθεώρηση της κοινή ε, αλληλευτικής πολιτικής, αλλά ταυτόχρονα βλέπουμε ότι προσπαθούν πολλά ε, σούπερ μάρκετ και πολλοί αλείς να πωλήσουν προϊόντα από λεγόμενες αηφόρες ε, πηγές αλίας και έτσι εξασφαλίστε ένα σύστημα, αναπτύσσετε μάλλον ένα σύστημα πιστοποίησης από το Αλληλευτικό Συμβούλιο, πράγμα το οποίο σημαίνει και επιπλέον χρήματα για τον αλληλεία και περισσότερη εμπιστοσύνη για τον καταναλωτή και αηφορία. Αυτή η εκπαραλλήλου ε, ανάπτυξη της πιστοποίησης της προέλευσης των νύχθειων είναι κατά την άποψη σκόπιμο να υποστηριχθεί. Ευχαριστώ τον κύριο Ντέβις για την ερώτηση που είναι πραγματικά ενδιαφέρουσα. Ξέρετε ότι ε, ο commissioner boards και η διεύθυνση είχαν κάνει μια προσπάθεια να προχωρήσουν αυτό το σύστημα το labeling, αυτό που λέμε labeling στο θέμα των ε, ε, ψαριών δεν είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα. Πρέπει να πω ότι αυτή η προσπάθειά μας ακόμα δεν έχει πάρει καλή έκθεση impact assessment. Δεν έχουμε καλή έκθεση από την αρμόδια επιτροπή που κάνει το impact assessment, ώστε να μας βοηθήσει να προχωρήσουμε μπροστά. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε ώστε να εξασφαλιστεί αυτή η έκθεση και να προχωρήσουμε με το σύστημα της υιοθέτησης ενός συστήματος ελάχιστων κριτηρίων, ελάχιστων κριτηρίων, ώστε ένα προϊόν αλίας που καταλήγει στο σούπερ μάρκετ να έχει την ετικέτα ότι έχει ψαρευθεί με έναν τρόπο που είναι συμβατός με sustainable fisheries. Όμως εσείς αναφέρεστε σε κάτι περισσότερο και πολύ πιο ενδιαφέρον. Αναφέρεστε στο λεγόμενο eco-labeling, δηλαδή στη δυνατότητα να υπάρχει μια ε, ετικέτα που να, κατά κάποιο τρόπο να πιστοποιεί την, ε, το eco-labeling του προϊόντος. Και γνωρίζω ότι υπάρχουν πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες στο θέμα αυτό. Υπάρχει και μια πρωτοβουλία στην οποία έχει εμπλακεί και το WWF, από ό,τι ξέρω. Είναι πρωτοβουλίες που είναι ενδιαφέρουσες, δίνουν το κάτι παραπάνω και νομίζω ότι ε, μπορούμε να συνεργαστούμε καλά με τους οργανισμούς οι οποίοι κάνουν αυτή την πολιτική, ε, ε, δημιουργώντας βέβαια ένα ενιαίο σύστημα πιστοποίησης δικό μας, ευρωπαϊκό, με βάση το οποίο και αυτοί θα κρίνονται. Eh, Ευχαριστώ. Από ό,τι βλέπω και η Ισπανική Προεδρία αναφέρεται στο eco-labeling, στην οικολογική σήμανση. Ε, μένα αυτό που με ενδιαφέρει όμως περισσότερο είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην καταλήξει να επανεφεύρει τον ε, τροχό και ε, να μην κάνει πράγματα τα οποία ήδη έχουν αναλάβει και κάνουν τα διάφορα όργανα πιστοποίηση. Απλώ να ενισχύσουμε και να βελτιώσουμε αυτή την πρακτική θέλω. Το σύστημα το οποίο εισηγείται η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα σύστημα προδιαγραφών το οποίο αναφέρεται στα ελάχιστα κριτήρια τα οποία είναι αναγκαία έτσι ώστε ο καταναλωτής να έχει την επίσημη πιστοποίηση από εμά, ότι το ψάρι που καταναλώνει έχει ψαρευτεί με σωστό τρόπο. Το ποιος θα εφαρμόσει αυτό το σύστημα. Αυτό είναι ένα θέμα ανοιχτό, όπου μην έχετε καμιά αμφιβολία, η Επιτροπή δεν προσπαθεί να υποκαταστήσει κανένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Στη συνέχεια έχει το λόγο. Άμε συγχωρείτε, διαδικαστικό. Κύριε Ρόντους Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Έχουμε ένα πολύ αυστηρό χρονοδιάγραμμα. Είχαμε τουλάχιστον ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα στην αρχή των εργασιών μα και ευχαριστώ πολύ. Χάρη στη δική σα επιδέξια καθοδήγηση των εργασιών έχουμε κερδίσει λίγο χρόνο. Από την ομάδα μου όμω υπάρχει και κάποιο ο οποίο δεν θέλει εξάπαντο να διατυπώσει ερώτηση, αλλά δεν είχε μπορέσει να βρει χρόνο μέσα στο πρόγραμμα αυτό. Θα μπορούσατε να προσθέσετε το όνομά του στο τέλο των εργασιών μα, εφόσον περισσέψει χρόνο, να έχετε δυνατότητα να μιλήσει. Eh, Κοιτάξτε κύριε Ρόντο, εγώ προσπαθώ να εξοικονομήσω χρόνο για να δώσω πιο πολύ χρόνο στην υποψήφια επίτροπο ώστε να μπορέσει να διευρύνει τι απαντήσει τη στο τέλο. Αυτό δεν μπορώ να, που δεν μπορώ να κάνω είναι να δώσω περισσότερο χώρο σε μια πολιτική ομάδα γιατί ο, ο χρόνο αγόρευση καθορίζεται βάσει του συστήματος DONT και πρέπει να εφαρμόσουμε επακριβώς τη μέθοδο DONT σε αυτή την ακρόαση. Λείπαμε πολύ, αλλά πρέπει να τηρήσω τους κανόνες που έχουμε θεσπιστεί για αυτή την ακρόαση γιατί πρέπει να είναι ίδιες οι συνθήκες για όλους και σύμφωνες με τους κανόνες που έχουμε. Και επομένως προσπαθώ απλώς να ξεκονομήσω χρόνο για την κυρία Επίτροπο και όχι για να αλλάξουμε την μέθοδο DONT. Στη συνέχεια λοιπόν έχει το λόγο ο κύριος Ριβελίνη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ποια πολιτική θα εισαγάγεται για την ε, αλία στη Μεσόγειο όπου ισχύουν κοινοτικοί κανονισμοί σε σχέση με το μέγεθος των ματιών των δικτύων για συγκεκριμένα αλλιευτικά είδη, ενώ σε άλλες χώρες οι οποίες δρούν σε διεθνή ύδατα, οι χώρες αυτές μπορούν να δρούν χωρίς ε, κανόνες με απώλεια του εισοδήματος της Ευρωπαϊκής Αλλιευτικής. Τι μπορούμε να κάνουμε με τις μη κοινοτικές χώρες που κατακλείζουν τις αγορές με αλλιεύματα σε βεβαίως καταστροφικές τιμές, πολύ χαμηλές τιμές. Κύριε Δαμανάκη. Ε, κύριε Ριβελίνη, ε, οι χώρες της Μεσογείου πράγματι υπόκεινται σε, οι χώρες της Μεσογείου που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπόκεινται σε ένα αυστηρό κανονισμό υπόκειται στους αυστηρούς κανονισμούς που έχουμε σε όλη την Ευρώπη και έχουμε ειδικά αυτό τον κανονισμό για τη Μεσόγειο. Ζητούμε από τα κράτη-μέλη να προχωρήσει στις προδιαγραφές που χρειάζονται για την εφαρμογή αυτού του κανονισμού. Θα κάνω ό,τι μπορώ ώστε μέσα στις συγκεκριμένες προθεσμίες αυτός να εφαρμοστεί. Καταλαβαίνω όμως τις δυσκολίες και καταλαβαίνω γιατί ορισμένες χώρες και πολλές χώρες θα έλεγα της Μεσογείου δεν, είναι ακόμα, δεν έχουν ακόμα ανταποκριθεί, δεν έχουν ακόμα συμμορφωθεί ε, στην εφαρμογή αυτού του κανονισμού. Δεν έχουν καθορίσει τις περιοχές που χρειάζονται μια ιδιαίτερη προστασία, δεν έχουν ε, καθορίσει ε, όλα όσα ζητούμε για την καταγραφή των ειδών κλπ. Αλλά το θέμα που θέτεται είναι ένα θέμα για το οποίο έχουμε όλοι ευθύνη και πρέπει να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Πράγματι ο Ιταλός ψαράς, πριν ρωτήθηκα κάτι αντίστοιχο για τον Έλληνα ψαρά, έχει την ανάγκη να συναγωνιστεί κάποιον άλλον από κάποια άλλη χώρα που βρίσκεται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο οποίος αισθάνεται μεγαλύτερη άνεση, ας το πω έτσι, εντός εισαγωγικών, να ψαρεύει χωρίς εφαρμογή κανονισμών. Ποια είναι η λύση. Η λύση είναι να προσπαθήσουμε να και ο άλλος ψαράς να εφαρμόζει το σωστό κανονισμό. Αυτή είναι η λύση. Πώς μπορούμε να το πετύχουμε. Μπορούμε να το πετύχουμε με μεγαλύτερη πίεση στους διεθνείς οργανισμούς όπου μετέχουμε και όπου μετέχουν και αυτές οι χώρες. Η Λιβύη, η Αλγερία μετέχει στον, ε, ε, στον περιφερειακό οργανισμό που έχουμε στη Μεσόγειο. Πρέπει εκεί να γίνει σαφές ότι ε, πρέπει να εφαρμόζονται οι κανονισμοί. Υπάρχουν άλλες χώρες με τις οποίες έχουμε συμφωνίες. Το Μαρόκο, παραδείγματος χάρη. Άρα έχουμε και ένα λόγο παραπάνω πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε στα πλαίσια των σχέσεων που έχουμε, των διεθνών σχέσεων, ώστε να εφαρμόσουν οι χώρες όλες τους κανονισμούς. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και αμυντικά αντανακλαστικά τα οποία μπορούμε να ασκήσουμε. Εάν γίνει σαφές ότι δεν θα επιτρέψουμε να εισάγονται παράνομα προϊόντα αλίας, ε, ε, IUU products, το οποίο έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε με βάση τον κανονισμό, τότε νομίζω ότι αυτό θα δημιουργήσει ε, ένα κίνητρο για συμμόρφωση. Το θέμα είναι να ελέγξουμε αποτελεσματικά την εφαρμογή αυτού του κανονισμού, του IUU, και εδώ πραγματικά και το πρακτορείο που έχουμε, το agency που έχουμε στο Βίγκο, και οι δυνάμεις που έχουμε, το πλοίο που έχουμε, έχουμε αγοράσει ένα πλοίο για τον έλεγχο, το οποίο είναι καινούριο και καλό, όλες αυτές οι δυνάμεις που έχουμε θα, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο θα εργαστούν ώστε να έχουμε εφαρμογή των κανονισμών. Αυτή, αυτός είναι ο μόνος δρόμος. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε, αλλά νομίζω ότι η απάντησή σας δεν είναι συγκεκριμένη, διότι μιλάμε για προάσπιση των κοινοτικών δικαιωμάτων. Ποιες δεσμεύσεις αναλαμβάνετε λοιπόν συγκεκριμένα για να προωθήσετε τα συμφέροντα του κοινοτικού αλλιευτικού στόλου σε σχέση με τις εξοκοινωτικές χώρες που χρησιμοποιούν επιθετικές πολιτικές. Εσείς θα αποφασίσετε για την Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν να προασπιστείτε την Ευρώπη με δυναμικότητα και χωρίς ιδεολογικές ε, προκαταλήψεις. Τι θα κάνετε με τον λιβικό αλλιευτικό στόλο και ιδιαίτερα ως προς την πολιτική του Καντάφη, ο οποίος αλλάζει τα χωρικά ύδατα και χρησιμοποιεί μεγαλύτερη εμβέλεια ε, υδάτων. Τι θα κάνετε σε σχέση με την πολιτική Μπορς όπως είχε οριστεί το 2008. Δώσω τον κύριο συνάδελφο ότι όλοι έχουμε ασφαλώς τις ιδέες μας, αλλά ως Επίτροπος θα εφαρμόσω απολύτως ε, τα εργαλεία που έχω στα χέρια μου σαν Επίτροπος. Εννοώ δηλαδή την επιστημονική τεκμηρίωση την οποία θα έχω, το, τις εισηγήσεις που θα έχω από τον κοινωνικό διάλογο ο οποίο θα υπάρχει και τις δυνατότητες της διεύθυνσης η οποία θα βρίσκεται ελπίζω αν με επιβεβαιώσετε ως επίτροπο κάτω από τις εντολές μου ώστε να είμαστε όλοι περισσότερο αποτελεσματικοί. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Δεν νομίζω λοιπόν ότι μπορώ να δεχτώ αυτά τα οποία υπόθηκαν για ιδεολογικές προκαταλήψεις. Είναι πολύ συγκεκριμένη η νομοθεσία, πολύ συγκεκριμένη και πρέπει να εφαρμοστεί. Πώς θα εφαρμοστεί και ποιες είναι οι δεσμεύσεις μου. Η δέσμευσή μου μπορεί να είναι η προσωπική ότι εγώ ίδια θα φροντίζω να είμαι εδώ στην Επιτροπή σας όποτε έχετε τέτοια θέματα. Η δέσμευσή μου μπορεί να είναι ότι εγώ ίδια θα φροντίσω ώστε στην συνεδρίαση του, της Επιτροπής για τη Μεσόγειο, στην οποία μετέχει και η Λιβύη, να τεθεί το θέμα και να δούμε τα μέτρα συμμόρφωσης των κανονισμών να δούμε πώς μπορούν οι διεθνείς σχέσεις να συνεργαστούμε με τις αντίστοιχες διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε στα πλαίσια της άσκησης διεθνούς πολιτικής να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ο στόχος θα είναι να εφαρμοστούν οι κανονισμοί από όλους. Δεν μπορούμε να αναιρέσουμε την εφαρμογή των κανονισμών και να καταστρέψουμε τα αποθέματα που έχουμε στις θάλασσές μας επειδή κάποιοι το κάνουν. Θα πρέπει να πείσουμε και ναι. αυτούς να οδηγηθούν στη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Για να κλείσουμε αυτό το γύρο, η κυρία Τρότμαν, για ένα λεπτό έχει το λόγο. Κύριε Επίτροπε, κύριε Υποψήφια Επίτροπε, η ομάδα μου από την ε, νέα Επιτροπή αναμένει να δει τι είδους θέση θα επιφυλάξει σε μια καλύτερη και περισσότερη ανάπτυξη, την αντιμετώπιση των κοινωνικών αποκλεισμών, στρατηγική του 2020 και επίσης όλα αποτελούν ένα κοινό περιβάλλον. Η κρίση που αντιμετωπίζουμε πρέπει να αντιμετωπιστεί, περιμένουμε τις προτάσεις σας, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και την περιβαλλοντική κρίση στην Αλία και των ακτών και των θαλασσών. Αυτό η ε, κρίση πλήττει όλη την αλυσίδα παραγωγής στην Αλία Ερωτώ λοιπόν πώς και τι συγκεκριμένα μέτρα μπορείτε να προτείνετε, αυτά που προεξαγγέλλετε ως προς την καινοτομία στις αγωγικές παρατηρήσει. παρατηρήσεις. Υποψήφια παρακαλώ. Ευχαριστώ την κυρία Τροτμάν για την ερώτηση και για τη φιλοξενία στην πολύ ωραία πόλη τη. Ε, πράγματι το θέμα ε, της ε, πλήρους απασχόλησης είναι πολύ μεγάλο θέμα και πολύ δύσκολο. Και πολύ δύσκολο στα πλαίσια μάλιστα της οικονομικής κρίσης ε, γίνεται ακόμα δυσκολότερο. Συζητήσαμε το θέμα της οικονομικής κρίσης ε, και με τον πρόεδρο Παρόζο και με το κολέγιο, το, κολέγιο, το designated κολέγιο, ε, σε μια πολύ αναλυτική συζήτηση και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι υπάρχει γενική άποψη ότι η απασχόληση πρέπει να εξασφαλιστεί. Θέλω εδώ να προσθέσω την προσωπική μου άποψη. Καταλαβαίνω ότι η απασχόληση δεν εξασφαλίζεται πάντα απλώς και μόνο από την ανάπτυξη. Μπορεί να έχουμε οικονομική ανάπτυξη και να μην έχουμε αύξηση της απασχόλησης ή να μην έχουμε καν σταθεροποίηση των θέσεων απασχόλησης. Άρα χρειάζεται να ασκηθεί ειδική πολιτική για την απασχόληση και ε, είμαι σίγουρη ότι ο αρμόδιος επίτροπος και η αρμόδια διεύθυνση θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί ώστε να εξασφαλιστεί αυτό. Εγώ θα συνεργαστώ όσο μπορώ μαζί, ώστε στον τομέα της αλίας να μην έχουμε απώλεια θέσεων εργασίας, να μην έχουμε απώλεια θέσεων εργασίας και να εξασφαλίσουμε μια καλύτερη κατανομή των δυνατοτήτων που έχουμε για την αλία, ώστε να εξασφαλίσουμε τις θέσεις εργασίας ε, του τομέα. Από εκεί και πέρα βέβαια είναι και θέμα συνολικά πώς θα εφαρμοστούν οι κανονισμοί ώστε η περιβαλλοντική κρίση, η οποία αμφισβήτητα υπάρχει, να συνδυαστεί με ε, στοιχεία οικονομικής ανάπτυξης και με τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας. Και νομίζω ότι εδώ μπορούμε να εξασφαλίσουμε και τη χρησιμοποίηση των εργαλείων που δίνει το Maritime Policy. Το Maritime Policy μας δίνει εργαλεία γενικότερης χωροταξικής κατανομής των δραστηριοτήτων και κινήτρων νέας ανάπτυξης με βάση τη γνώση Μπορούμε λοιπόν να δούμε και να έχουμε μια αντίστοιχη ερευνητική υποστήριξη για το πώς καλύτερα μπορούμε να ωφεληθούμε, ε, να εξασφαλίσουμε το συνδυασμό της απασχόλησης με τις άλλες δραστηριότητες. Όπως είπα και στην αρχή, αυτό που πιστεύω είναι ότι μπορούμε να συνδυάσουμε και τα τρία και την ε, περιβαλλοντική ε, αηφορία και την ε, κοινωνική και την οικονομική. Και πραγματικά θα μπορέσουμε να τα συνδυάσουμε αν καταλάβουμε ότι όλα πρέπει να πάνε μαζί και δεν ξεχωρίσουμε το προβάδισμα κανενός. Συμπληρωματική ερώτηση, κυρία Τρότσμαν. Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση σας, κύριε υποψηφία Επίτροπε. Θα συμμετάσχουμε και εμείς, θα μας επιτρέψετε να συμμετάσχουμε σε αυτό το πρόγραμμα εργασίας. Η έρευνα η οποία θα μπορούσε να αποδώσει πράσινες θέσεις εργασίας και η συζήτηση για τη δημιουργία αυτών των θέσεων εργασίας δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο σε σλόγγαν. Πρέπει να είναι μια ουσιαστική προτεραιότητα για την προσεχή θητεία, τη δική σας και τη δική μας, ιδιαίτερα και στην Αλία. Τι έχετε να μας προτείνετε. Ε, μακάρι η αποσχόληση να η απασχόληση στον ελευτικό τομέα να ήταν δική μας αρμοδιότητα μόνο ώστε να μπορούσαμε να κάνουμε, να μπορώ να δώσω τη δέσμευση, να, πω, να μιλήσω για δέσμευση και να είμαι σίγουρη ότι θα το εφαρμόσω, ότι οι βουλευτές θα συμμετέχουν πραγματικά. Αλλά στο βαθμό που είναι αρμοδιότητα της διεύθυνση employment και του commissioner του υπεύθυνου για την employment, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θα συνεργαστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό το οποίο μπορώ να διαβεβαιώσω την Επιτροπή είναι ότι ε, θα είμαι πραγματικά στη διάθεσή σας θα είμαι εδώ πολύ συχνά, σκοπεύω να είμαι τουλάχιστον τρεις φορές το χρόνο και θα είμαι εδώ όποτε νομίζετε ότι υπάρχει θέμα το οποίο πρέπει να συζητηθεί. Οπωσδήποτε πριν και μετά από μεγάλα γεγονότα ή την εφαρμογή πολιτικών, η Επιτροπή Ελίας θα ενημερώνεται χωριστά από μένα προσωπικά. Ευχαριστώ για να κλείσουμε τον τελευταίο γύρο ερωτήσεων που θα ακολουθήσει η σειρά των ερωτήσεων από τις μεταφορές. Ο κύριος Μάτο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρία ε, Επίτροπε. Οι περιφερειακές περιοχές έχουν ιδιαίτερες συνθήκες σε διάφορα επίπεδα και για την αλία ιδιαίτερα. Προβλέπει για αυτές οι συνθήκες της Λισαβόνας μια ιδιαίτερη μεταχείριση. Είναι πάρα πολλά τα εμπόδια τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε σε καθημερινό επίπεδο, αλλά η αλληλευτική δραστηριότητα ιστορικά είχε μεγάλη σημασία για την οικονομία αυτών των περιοχών και θέλουμε να συνεχίσει να έχει αυτό το ρόλο. Πιστεύετε, κύριε Επίτροπε, ότι για αυτό το λόγο είναι απαραίτητη όλη η υποστήριξη των θεσμικών οργάνων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ένα άλλο θέμα το οποίο συνδέεται με το προηγούμενο, κατά την άποψή σα, θα μπορούσε να γίνει για να βοηθήσουμε τον αλληλευτικό τομέα για στις υπερπεριφερικές περιοχές και την ηχθειοκαλλιέργεια ακόμα και θεωρείται ότι οι λύσεις οι οποίες εφαρμόζονται τώρα είναι επαρκείς για να υπερκεραστεί η μειορεκτική θέση αυτών των περιοχών. Τέλος, ποια είναι η θέση σας σε σχέση με μια ε, ενδεχόμενη ενίσχυση του σχεδίου για την αλία και την ηχθειοκαλλιέργεια που έχει τελματωθεί τα τελευταία χρόνια. Ε, Πράγματι, κύριε Μάτο, η συνθήκη προβλέπει ειδικό καθεστώς για τις outermost regions και είναι φυσικό διότι η απόσταση από το κύριο κορμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δημιουργεί ορισμένα προβλήματα τα οποία πρέπει να ξεπεραστούν. Αυτή τη στιγμή τρέχει ένα οικονομικό πρόγραμμα με ορίζοντα το, δύο, το POSEI πρόγραμμα, ε, ασφαλώς το ξέρετε, το οποίο τρέχει με ορίζοντα το 2013 ε, το οποίο εφαρμόζεται και το οποίο θα συνεχίσει να εφαρμόζεται και προβλέπει την οικονομική βοήθεια των χωρών αυτών, των ε, περιοχών αυτών. Το δεύτερο που έχω να πω είναι ότι υπάρχει, όπως ξέρετε, καθεστώς ειδικής πρόσβασης, exclusive access, ε, των περιοχών αυτών στα χωρικά ύδατα. Το καθεστώς αυτό ε, θα συνεχίσει να εφαρμόζεται. Μάλιστα στα πλαίσια του διαλόγου έχουμε και μία πρόταση ενδεχομένως στα πρώτα 12 μίλια να αφιερωθούν ειδικά για small scale fisheries, για μικρά σκάφη. Είναι μια πρόταση στα πλαίσια του διαλόγου την οποία επίσης θα εξετάσουμε. Ε, όσον αφορά την ε, περαιτέρω οικονομική ε, ενίσχυση των περιοχών αυτών, αυτό που μπορούμε να δούμε είναι οτιδήποτε να συζητήσουμε καλύτερο στα πλαίσια του, του, της συζήτησης για τα new financial perspectives, τις νέες οικονομικές προοπτικές τις οποίες έχουμε και όπου μπορούμε να δούμε και τις δικές σας προτάσεις. Εάν υπάρξει κονδύλι για την ηχθειοκαλλιέργεια μπορούμε να δούμε το θέμα της ιοχθακαλλιέργειας, αλλά προς το παρόν από τα κονδύλια τα οποία έχουμε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα καλύτερο. Τέλος, νομίζω ότι αυτές οι περιοχές έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και θα μπορούσαμε να δούμε μια καλύτερη συνεργασία μαζί τους. Μια καλύτερη συνεργασία μαζί τους. Δηλαδή σκέφτομαι ότι ίσως θα μπορούσαμε να καλέσουμε τους εκπροσώπους και τις διοικήσεις όλων αυτών των περιοχών και να συζητήσουμε στα πλαίσια της αναμόρφωσης της κοινή αλληλευτικής πολιτικής το ενδεχόμενο να έχουμε ένα συμβουλευτικό όργανο, ένα ΡΑΚ για αυτές τις περιοχές. Αλλά αυτά θα τα δούμε εφόσον και οι ίδιοι συμφωνούν, ε, θα πρέπει να έρθουν εδώ να δούμε πώς μπορούμε να βρούμε, ώστε να οδηγηθούμε σιγά σιγά στην επεξεργασία μιας πολιτικής για όλα τα outer ε, most regions συνολικά. Από εκεί και πέρα το μόνο που έχω να πω είναι ότι προσωπικά θα σεβαστώ τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Γνωρίζω ότι όχι τα Κανάρια από τα οποία από ε, ε. νομίζω προέρχεστε, αλλά οι αζόρε έχουν προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για ένα θέμα. Θα σεβαστώ την απόφαση του Δικαστηρίου. Ε, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πράγματι είναι σημαντικό το θέμα αυτό των υπερπεριφερειακών περιοχών και τη αλίας εκεί η οριοθέτηση των υδάτων είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Είπατε ότι εφαρμόσετε το POSEIP, αλλά τα κονδύλια του POSEIP είναι παγωμένα από το έτος 2001 και έχει χάσει ουσιαστικά την ε, σημασία του για την επίτευξη του στόχου αυτού. Πώς θα μπορούσε λοιπόν να τροποποιηθεί αυτή η κατάσταση, εσείς θα αναλάβετε ένα σημαντικό αξίωμα, αλλά πρέπει επίση να αναλάβετε και μια δέσμευση εναντί των υπερπεριφερειακών περιοχών, που είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την Ευρώπη και πρέπει να είναι και για εσά και για την Αλία επίση. Τα κονδύλια τα οποία εκταμιεύονται, εκταμιεύονται στη βάση ενός πολιετού προγράμματος. Δεν είναι παγωμένα, υπάρχει ένα πολιετές πρόγραμμα και από εκεί και πέρα οι ίδιες οι περιοχές τα κατανέμουν. Το πολιετές πρόγραμμα αυτό ε, βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν μπορεί να αλλάξει. Μπορούμε να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε στο νέο πρόγραμμα το οποίο θα υπάρχει. Όσον αφορά το καθεστώς το οποίο έχει να κάνει με την ε, ε, ειδική, το exclusive access σε αυτές τις, σε αυτές τις περιοχές, αυτό επαναλαμβάνω ένα καθεστώς το οποίο υπάρχει και το οποίο θα εφαρμοστεί. Υπάρχει μία προσφυγή των αζωρών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το θέμα, θα εφαρμοστεί η απόφαση του δικαστηρίου. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πρεζέδο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Κυρία Επίτροπε, μέσα στα πλαίσια, γνωρίζω ότι έχετε ε, πείρα σε ορισμένα θέματα και δώσατε σαφείς απαντήσεις. Πιστεύω ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια, την ποιότητα και τη συμπερίληψη. Πιστεύετε ότι μέσα στα πλαίσια της ασφάλειας θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την παρουσία του αλλιευτικού στόλου στο εξωτερικό και τι πρέπει να κάνουμε σε σχέση με τα εισαγόμενα προϊόντα. Δηλαδή θα πρέπει να πληρούν τις ίδιες προδιαγραφές για να υπάρχει πραγματική ανταγωνιστικότητα. Και τι θα γίνει σε σχέση με την βιοτεχνική αλληλεία σε αυτό το τομέα και στα προϊόντα που προβάλλουν. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Σε σχέση με την παρουσία του στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα, διεθνή ύδατα, αυτή η παρουσία είναι πολύ σημαντική. Έχουμε περίπου 340 πλοία που ψαρεύουν με βάση το καθεστώς των ε, ε, Fisheries Agreements, των διμερών συμφωνιών και έχουμε περίπου 6.000, κοντά 6.000, 5.800 πλοία τα οποία ψαρεύουν σε διεθνή ύδατα με βάση την συμμετοχή μας στα RFMO, στα, στους μεγάλους ε, Regional Fisheries ε, Management Organizations. Ε, είναι μια πολύ σημαντική δύναμη η οποία πρέπει να προστατευτεί. Συμφωνώ ότι πρέπει να εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες, οι ίδιοι κανόνες όπως είπατε, και στην περίπτωση των εισαγόμενων προϊόντων οι ίδιοι κανόνες αλίας. Γι' αυτό εξάλλου βρισκόμαστε σε μια προσπάθεια εφαρμογής του διεθνούς κανονισμού του iuu regulation είμαστε σε συνεργασία με 150 κοντά χώρες στην προσπάθεια να εφαρμοστεί αυτός ο κανονισμός θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Από εκεί και πέρα αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι όλα αυτά τα αποτελέσματα να έχουν αντίκτυπο, συμφωνώ μαζί σας, και στους ε, ε, ψαράδες που έχουν μικρά σκάφη. Διότι εκεί, αν θέλετε, κρίνονται τα προβλήματα και σε ορισμένες χώρες, ιδιαίτερα στις χώρες της Μεσογείου, αλλά και σε άλλες χώρες, έχουμε όχι το 80, το 90% των σκαφών μικρά σκάφη. Άρα το θέμα είναι πώς θα φτάσει όλη αυτή η νομοθεσία σε αυτά τα μικρά σκάφη χωρίς να δημιουργήσει συνθήκες απαγορευτικές για την επιβίωσή τους. Είπα πριν ε, ορισμένα μέτρα που μπορούμε να πάρουμε. Εξαίρεση από αυστηρή εφαρμογή ορισμένων κανονισμών. Ειδική χρηματοδότηση Θέλω να το δω αυτό το θέμα της ειδική χρηματοδότησης. Δεν μπορούμε να έχουμε χρηματοδότηση για νέα σκάφη, αλλά μπορούμε να δούμε ειδική χρηματοδότηση για τα μικρά σκάφη, ιδιαίτερα στο θέμα του, της ανανέωσης, του innovation, για να είμαι σαφέστερη, των εργαλείων τους, της τεχνολογίας τους. Μπορούμε να βρούμε τρόπους, έτσι ώστε να έχουμε πραγματικά καλύτερα αποτελέσματα. Ελπίζω ότι θα έχω τη συνεργασία σας στον τομέα αυτό. Έχετε δικαίωμα ε, συμπληρωματικής ερώτησης για 30 δευτερόλεπτα. Θα ήθελα να τονίσω ότι ως προς την παρουσία λιευτικού στόλου στα διεθνή ύδατα, όπως ξέρετε, ε, εγώ προέρχομαι από μία περιφέρεια που εξαρτάται από την αλία και οι αλληλείς ε, στις δική μου περιφέρειες βασίζονται πάρα πολύ στην ε, κοινή αλλιευτική πολιτική. Θέλετε να απαντήσετε κυρία Δαμανάκη. Μόνο μια συμπληρωματική φράση για ένα θέμα που δεν υπόθηκε. Ε, μας ενδιαφέρει η παρουσία των ε, αλλιευτικών σκαφών στα διεθνή ύδατα και θα ασχοληθούμε και με την αντιμετώπιση ενός καινούργιου φαινομένου που υπάρχει. Αναφέρομαι στο θέμα της πειρατείας. Ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το πρόγραμμα Αταλάντα. Το πρόγραμμα Αταλάντα αναφέρεται στην προστασία των merchant fleets, των ε, εμπορικών σκαφών των εμπορικών σκαφών ε, και ήδη υπάρχουν ορισμένα προβλήματα. Η Ισπανία και ε, η Γαλλία έχουν στείλει αντιπροσωπεία στην Αταλάντα. Θα πρέπει να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε ώστε η επιχείρηση να καλύψει και την προστασία των αλλιευτικών σκαφών. ευχαριστώ τέλος ε, το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Τσουκαλάς. Κύριε Τσουκαλάκη, το λόγο. Κύριε Επίτροπε, στο Ευρωκοινοβούλιο και να σας ευχαριστήσω για τις απαντήσεις που μέχρι σήμερα μας δώσατε. Προσωπικά είχα την ευκαιρία να απολαύσω τον συνδυασμό ενός τεχνοκράτη πολιτικά κοινοβουλευτικά ευαίσθητου και ενός πολιτικά, πολιτικού τεχνικά γράμματου. Με αυτή την έννοια θα ήθελα να σας θέσω ένα ερώτημα που έθεσε και ο κύριος Μιλάνα προηγουμένως Πολλοί υποστηρίζουν ότι η υδατοκαλλιέργεια έχει αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και βλάπτει ιδιαίτερα τον τουρισμό, παραβλέποντας ίσως ότι η βιωσιμότητα δεν περιλαμβάνει μόνο την οικολογική διάσταση, αλλά και την οικονομική και την κοινωνική. Πιστεύετε ότι η ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας και η βιώσιμη ανάπτυξη είναι έννοιες που μπορούν να συνεπάρξουν. Ποιες είναι οι δράσεις που προτίθεστε να αναλάβετε, εάν μπορείτε τώρα να το πείτε, για την πρόθεση της βιώσιμης και οργανικής υδατοκαλλιέργειας. Έχετε κυρία Δαμανάκη. Ε, ευχαριστώ, κύριε Τσουκαλά. Ε, η απάντηση στο ερώτημα αν μπορεί να συνδυαστεί η ηχθειοκαλλιέργεια με την αηφορία, ε, η απάντηση είναι ότι θέλω να το ελπίζω. Θέλουμε να, το, προσπαθήσουμε, θέλουμε να το καταφέρουμε. Οι επιστήμονες μας λένε ότι μπορεί να γίνει αυτό. Μπορεί να γίνει. Εφόσον το λένε οι επιστήμονες και εφόσον ε, έχουμε την επιστημονική βάση και την τεκμηρίωση ότι αυτό μπορεί να γίνει, πρέπει να το προχωρήσουμε. Βέβαια, εάν μιλούμε για ανάπτυξη της ηχθειοκαλλιέργειας σε συνδυασμό με την αηφορία, τότε χρειάζονται προϋποθέσεις. Υπάρχουν συνθήκες που πρέπει να εφαρμοστούν. Δεν είναι τόσο απλό. Ε, μιλήσατε για... και εν πάση περιπτώσει πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα εξασφαλίσουμε ώστε πραγματικά η χθιοκαλλιέργεια να είναι συμβατή με το περιβάλλον. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα εδώ, πάρα πολλά θέματα, περιβαλλοντικά θέματα. Οι επιστήμονες όμως λένε ότι έχουν τις λύσεις και νομίζω ότι σε συνεργασία και με την αρμόδια διεύθυνση περιβάλλοντος ή εν πάση περιπτώσει αν καταφέρουμε να υπάρξει μια ε, συνεκτική πολιτική για την ηχθειοκαλλιέργεια ε, με τη συνεργασία και του Κοινοβουλίου, το οποίο είναι ευαίσθητο στο θέμα αυτό, ε, θα έχουμε τη δυνατότητα να ελέγξουμε τα μέτρα αυτά. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα θέματα. Μιλήσατε για οργανική ηχθειοκαλλιέργεια. Αυτό είναι κάτι παραπάνω και οι επιστήμονε λένε ότι υπάρχουν τέτοιοι τρόποι. Έχει να κάνει με την τροφή που δίνουμε στα ψάρια. Θα μπορούσε ας πούμε, να μιλήσουμε για ειδικέ κατηγορίε ηχθειοκαλλιέργειας όπου η τροφή είναι αποκλειστικά φυτική, δεν είναι ζωική. Υπάρχουν πολλά, πολλά θέματα, πολλά ανοιχτά θέματα ε, ε, που μπορούμε να δώσουμε λύσεις έτσι ώστε να μιλήσουμε για ανώτερη ποιότητα και στον τομέα αυτό. Θα προχωρήσουμε με βάση τις δυνατότητες που έχουμε. Τέλος, θέλω να αναφερθώ στο θέμα της ε, συνεργασίας, θέλω να πιστεύω ότι είναι συνεργασία της εκδοκαλλιέργειας με τον τουρισμό. Μπορούν να συνεπάρξουν υπό Και εδώ ακριβώς είναι αυτό που μπορεί να κάνει, αυτό που λέμε, που λέμε Integrated Maritime Policy και Integrated Special Planning. Μπορούμε να εφαρμόσουμε τα εργαλεία ώστε η χωροταξία να δώσει θέση και για τον τουρισμό και για την αλεία. Eh, eh, Ευχαριστώ κύριε Αδαμανάκη. 30 δευτερόλεπτα συμπληρωματικό ερώτημα αν θέλετε. Η απάντησή σα μου δίνει το δικαίωμα να σα ρίξω μια μικρή παγίδα, μια που αναφέρατε για την επιστημονική έρευνα. Πάρτε λοιπόν την ερώτηση ως προς την έρευνα και την αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογικών μεθόδων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, τι πρόκειται να κάνετε. Η έρευνα είναι πολύ σημαντική κύριε Τσουκαλά. Ξέρω ότι εσείς από την πείρα σας το ξέρετε αυτό. Ε, δυστυχώς τα κονδύλια που έχουμε εμείς είναι μικρά. Αυτό πρέπει να το πω. Δεν είναι κονδύλια που ικανοποιούν τα κονδύλια που έχει η DG Mare στη διάθεσή της για την έρευνα είναι μικρά και ένα μέρος από αυτό είναι ανάγκη να δίνεται ευθύ εξ αρχής για να εξασφαλίσουμε την επιστημονική υποστήριξη από τον ISIS και από την Επιστημονική Επιτροπή που έχουμε, τη Scientific Committee for Fisheries. Άρα περιθώρια για να έχουμε μια ειδική μελέτη πάνω στην ε, ηχθειοκαλλιέργεια πιστεύω δεν υπάρχουν, άλλωστε αυτή θα πρέπει να είναι μια πολύ μεγάλη μελέτη. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ ώστε στα πλαίσια της συνεργασίας για το καινούργιο, το Fifth ε, Research Program, μαζί με, την, ε, με τον αρμόδιο, την αρμόδια συνάδελφο στην προκειμένη περίπτωση, αν επιβεβαιωθούμε όλοι ως κολέγιο, ε, ώστε να έχουμε ενδεχομένως ένα κονδύλι από, το, από τα κονδύλια της έρευνας. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε ακόμα ένα λεπτό που έχουμε κερδίσει. Τώρα θα είμαι πάλι πάρα πολύ αυστηρή για την Επιτροπή Μεταφορών. Όχι, έχετε ένα λεπτό περισσότερο από του υπόλοιπου. Αυτό το λεπτό το οποίο μας περισσεύει θα το δώσω στην κυρία Επίτροπο όμως. Πρώτα απ' όλα. Και για ένα λεπτό έχει το λόγο ο κύριος Κουμουτσάκος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μιλώντας πρώτος από την Επιτροπή Μεταφορών, καλωσορίζω και καλημερίζω την κυρία Δαμανάκη. Κυρία Δαμανάκη, συγκρατώ με ικανοποίηση τις συχνές και ουσιαστικές αναφορές σας στην ανάγκη στενής συνεργασίας δική σας και της Επιτροπής συνολικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βέβαια, ομολογώ ότι δεν ήταν έκπληξη, τουλάχιστον σε εκείνους που γνωρίζουν τη μακρά κοινοβουλευτική σας πορεία στην Ελλάδα. Στην εισαγωγική σα ομιλία αναφερθήκατε γενικά μόνο στην ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Αυτό που λέμε γαλάζια το γαλάζιο βιβλίο, τη γαλάζια βίβλο του 2007. Θα ήθελα να γίνετε πιο συγκεκριμένοι αν είναι δυνατόν. Δύο χρόνια μετά την υιοθέτησή της, πώς αξιολογείτε την εφαρμογή της, που έχετε εντοπίσει και ποια κενά, αδυναμίες ή καθυστερήσει στην εφαρμογή της. Τι θα κάνετε για να δώσετε λύσεις και με ποιες προτεραιότητες. Αλήθεια, πού βρίσκεται η ιστορία της διαμόρφωσης του Ευρωπαϊκού Άτλαντα Θαλασσών, αν μπορείτε να μας πείτε. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ τον κύριο Κουμουτσάκο. Ε, ευχαριστώ που ερώτησε για αυτό το θέμα, για το Integrated Maritime Policy. Είναι η πρώτη ερώτηση που δέχομαι για το θέμα αυτό και ε, είναι φυσικό γιατί μιλούμε για μια καινούργια πολιτική. Αναφέρθηκε στην Πράσινη Βίβλο του 2007, έχουμε ήδη το μπλε βιβλίο που εφαρμόζουμε. προσπαθούμε τέλος πάντων να προσπαθούμε να έχουμε την καλύτερη δυνατή συνέργεια και συνεργασία με άλλες διευθύνσεις και με άλλους επιτρόπους. Γιατί όπως ξέρετε η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική είναι μια πολιτική που για να εφαρμοστεί χρειάζεται τη συμμετοχή πολλών ε, ε, διευθύνσεων και πολλών επιτρόπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλούμε και για το ασφαλώς τη δική σας επιτροπή, την Επιτροπή Transport, μιλούμε και για τη διεύθυνση Environment, ε, έχουμε, το, τις, έχουμε τις μεταφορές, το περιβάλλον, τις εξωτερικές σχέσεις, έχουμε πάρα πολύ την εσωτερική αγορά, πάρα πολλά θέματα τα οποία συνδέονται με την εφαρμογή αυτού που λέμε Integrated Maritime Policy. Ποια είναι η εκτίμηση για τη μέχρι τώρα εφαρμογή. Είναι θαρρυντική αν έπρεπε να χρησιμοποιήσω μία μόνο λέξη θα έλεγα ενθαρρυντική. Υπάρχουν εργαλεία καινούργια τα οποία έχουμε αναπτύξει. Ε, έχουμε ε, το Maritime Special Planning. Έχουμε ε, χωροταξία στο θαλάσσιο χώρο. Έχουμε μια διαδικασία σε σχέση με ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης του θαλασσίου χώρου που θα είναι πάρα πολύ σημαντικό έχουμε το πρόγραμμα αυτό για τη γνώση στον τομέα των θαλασσών και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καταλήλως αυτές τις γνώσεις. Για τον ε, των Θαλασσών, το λεγόμενο Μαράτλας στον οποίο αναφερθήκατε. Είναι ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο και ελπίζω να ανακοινώσουμε την πρόοδο για το θέμα αυτό τον επόμενο χρόνο. Ελπίζω λοιπόν ότι εν καιρό θα έχουμε αυτό τον Ευρωπαϊκό Ατλάντα των θαλασσών και των ωκεανών που βρέχουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαι σίγουρη ότι αναγνωρίζετε τη μεγάλη σημασία αυτού του Άτλαντα θα είναι σημαντικό όχι μόνο για την αλληλεία αλλά για τις μεταφορές, για την πολιτική <clears throat> περιβάλλοντος, για όλους. Ελπίζω την επόμενη άνοιξη θα μπορέσω να σας δώσω μια συγκεκριμένη ανακοίνωση για αυτό το σχέδιο, για το Μαράτλας. Ε, δευτερολογία, κύριε Είχατε στο πλαίσιο της, Ευρωπα... της απάντησης για την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στην ανάγκη συνεργασίας με άλλους συναδέρφους σας και με άλλες διευθύνσεις, ειδικά για τα θέματα των θαλασσίων μεταφορών. Ε, που αφορούν τον επίτροπο ε, συνάδελφό σας και τον επίτροπο μεταφορών ε, τον κύριο Κάλλας σας ανησυχεί το ενδεχόμενο να υπάρξουν κάποιες επικαλύψεις αρμοδιοτήτων Πώ θα το αποφύγετε αυτό ή εν πάση περιπτώσει πώς θα το λύσετε εάν κάτι τέτοιο προκύψει Παραδείγματο χάρη αναφέρομαι στο θέμα των λιμανιών ξέρουμε τη στρατηγική του σημασία για τις θαλάσσιες μεταφορές και το διεθνές εμπόριο αλλά και τη σημασία τους ως κέντρα διαμετακόμιση για την αλληλεία πώς τέτοια ζητήματα μπορεί να προκύψουν θα τα λύσετε. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω ότι δεν θα προκύψουν, κύριε Κουμουτσάκο, και αν προκύψουν, ο μόνος τρόπος να τα λύσουμε είναι μια καλή συνεργασία ανάμεσα σε μένα και τον άλλον Επίτροπο. Θέλω να είμαι πολύ σαφής. Αυτή τη στιγμή ο Επίτροπος Αλίας και Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής προεδρεύει σε ένα όργανο που υπάρχει από 10 επιτρόπους, ε, οι οποίοι ασχολούνται με το πώς ακριβώς θα προχωρήσουν στην εφαρμογή μιας τέτοιας ολοκληρωμένης πολιτικής χωρίς να υπάρχουν αυτά τα, αυτές οι αλληλοεπικαλύψεις στις οποίες αναφερθήκατε. Πρέπει, θα προσπαθήσω να συνεχίσουμε τη λειτουργία αυτού του οργάνου ε, έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη δυνατή συνεργασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε μια εξαιρετικά κρίσιμη φάση. Δεν έχουμε την πολυτέλεια, we can afford it, να το πω αγγλικά, δεν έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε διαφωνίες μεταξύ μας ή να προσπαθούμε να πατήσουμε ένα στο πόδι του άλλου. Από τη μεριά μου δεν σκοπεύω να το κάνω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 1.200 λιμάνια. Είναι μεγάλος πλούτος, Όσον αφορά τα θέματα αλληλεία, θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Είμαι σίγουρη ότι και ο κύριο Κάλλα, εάν επιβεβαιωθούμε, θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Ε, στα θέματα που τον αφορούν, δεν έχω σκοπό να παρέμβω. Κύριε Τικάου, για ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, από την 1η ε, Ιανουαρίου του 2007 η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βρέχεται πλέον και από τον εύξηνο πόντο την Μαύρη Θάλασσα, που έχει τεράστια στρατηγική σημασία. Όπως άλλωστε και ο δούναβη. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω ποια μέτρα σκοπεύετε να λάβετε ποια δέσμευση ε, μπορείτε να αναλάβετε ήδη τώρα για την καλύτερη ενσωμάτωση, συμπεριλήψη του εύξηνου πόντου στην κυρία πολιτική. Ε, και θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι στην ιστοσελίδα για τα θαλάσσια θέματα Υπάρχουν αιτήματα ε, για μάλλον τη υπηρεσία, για θαλάσσια θέματα, ε, δεν προβλέπεται ανάπτυξη σχεδίων για διαδρόμους πρόσβασης προς τον εύξηνο πόντο. Αυτό νομίζω θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Το τελευταίο το οποίο αναφέρατε δεν το γνωρίζω, θα το ελέγξω. Ε, χαίρομαι που το θέτετε, θα το ελέγξω με τις υπηρεσίες μου και θα δω ε, ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει. Αλλά το θέμα της ε, Μαύρης Θάλασσας, το θέμα του ευξήνου πόντου είναι πολύ σοβαρό, πράγματι. Ε, και είναι, είναι πολύ μεγάλη ευθύνη γιατί είναι ένα καινούριο πεδίο, κατά κάποιο τρόπο, καινούριο εφαρμογή της πολιτικής. Όπως ξέρετε έχουμε δύο χώρες, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Προσπαθούμε διστακτικά να εφαρμόσουμε πολιτική. Ρώτησα από ό,τι με ενημέρωσαν μόνο σε δύο είδη μέχρι στιγμής εφαρμόζουμε, δύο είδη ψαριών δύο είδη ψαριών εφαρμόζουμε στη Μαύρη Θάλασσα συστήματα οργάνωσης πολιτικής, management, fisheries management, μόνο για δύο είδη. Ε, η υπόθεση είναι δύσκολη διότι δεν είμαστε μόνο εμείς στη Μαύρη Θάλασσα όπως πολύ καλά ξέρετε. Η Μαύρη Θάλασσα, στη Μαύρη Θάλασσα έχουμε κυρίως ε, πολύ μεγάλες χώρες με πολύ μεγάλη επιρροή, με πολύ μεγάλη δύναμη. Έχουμε τη Ρωσία, έχουμε την Τουρκία, έχουμε την Ουκρανία. Ε, και ε, ζήτησα τα στοιχεία μου είπαν ότι 85% των αλλιευμάτων που αλλιεύονται στην Μαύρη Θάλασσα αλλιεύονται από τουρκικά σκάφη που είναι σκάφη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει λοιπόν να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή συνεργασία με αυτούς, με όλους, αν θέλουμε να πετύχουμε κάτι καλύτερο. Σήμερα ε, η Βουλγαρία και η Ρουμανία και η Τουρκία εκπροσωπούνται στην Επιτροπή που έχουμε για τη Μεσόγειο, την General Fisheries Committee, Mediterranean Committee. Ε, και εκεί λύνουμε κάποια θέματα. Ε, καταλαβαίνω ότι θα θέλετε να έχουμε καλύτερα, μια καλύτερη συνεργασία για την, ειδικά για τη Μαύρη Θάλασσα. Υπάρχουν ήδη τέτοια σχήματα. Υπάρχει το, η ε, οικονομική συνεργασία, οικονομική συνεργασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μετέχει στο πλαίσιο αυτής της οικονομικής συνεργασίας που συμπεριλαμβάνονται όλες οι χώρες της Μαύρης Θάλασσας και θα έλεγα επιτυχώς έχουμε αποτέλεσμα. Υπάρχουν και άλλα σχήματα συνεργασίας. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι θα εξετάσω αυτό το οποίο λέτε. Αλλά θέλω να ξέρετε ότι τίποτα δεν θα είναι καλό εάν δεν μετέχουν και οι άλλοι με δύο μόνο χώρες σε αυτή την τεράστια σημασία θάλασσα, με σημασία και για τα αναλυεία αλλά και για την ενέργεια και γεωπολιτική σημασία, θα είναι δύσκολο να προχωρήσουμε συμπληρωματική ερώτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να δούμε εσάς ως εταίρο για τη διαμόρφωση της στρατηγικής για το Δούναβι, μια στρατηγική που ακόμα βρίσκεται εν εξελίξη, όσο δεν αφορά την κοινή ε, πολιτική για τις θάλασσες πρέπει να πω ότι δεν περιορίζεται μόνο, δεν εξαντλείται μόνο στην αλία. Ερωτώ λοιπόν τι είδους μέτρα θα αναλάβετε για την ανάπτυξη των θαλάσσιων λιμένων τόσο ε, και των ε, λιμένων στους ποταμούς και σε παραθαλάσσιες περιοχές, σε εκβολές ποταμών ε, και για την ανάπτυξη βέβαια των παράκτων περιοχών. Ξέρω ότι αναπτύσσονται προτάσεις και σχέδια μέσα από τα διευθυντικά ταμεία, τα οποία ορισμένοι εκμεταλλεύονται και ορισμένοι χρησιμοποιούν περισσότερο για την περιφερειακή ανάπτυξη. Ερωτώ λοιπόν τι συγκεκριμένα μέτρα μπορείτε να προτείνετε και να αναλάβετε για μια ολοκληρωμένη εγκάρσια πολιτική για τη θάλασσα. Αναφερθήκατε στο Δούναβι ε, και, στις, ε, και στην ανάπτυξη του Δούναβι. Καταρχήν θέλω να πω ότι βεβαίως δεν είναι δική μου αρμοδιότητα αυτό. Κυρίως είναι θέμα ε, της περιφερειακής πολιτικής, όπως είπατε, και άλλων επιτρόπων. Όμως ενδιαφέρει και εμάς και ενδιαφέρει γιατί λόγου χάρη από τα στοιχεία που υπάρχουν για τη ρήπανση στη Μαύρη Θάλασσα φαίνεται ότι το 50% του φωσφόρου, λέω κάτι που τυχαίνει να θυμούμε, το 50% του φωσφόρου που βρίσκεται σήμερα στη Μαύρη Θάλασσα το φέρνει ο Δούναβης άρα λοιπόν εάν μιλούμε για ε, πολιτική περιβάλλοντος στη μαύρη θάλασσα πρέπει να συμπεριλάβουμε και τις ε, ε, ποταμούς που να συνεργαστούμε ώστε να έχουμε μια καλύτερη ανταπόκριση και για τα ποτάμια που χύνονται στη μαύρη θάλασσα. η θαλάσσια πολιτική στη μαύρη θάλασσα μπορεί να συνεισφέρει πολύ συγκεκριμένα γιατί μπορεί να οδηγήσει σε αυτό που λέμε integrated management της θάλασσας δηλαδή εφαρμόζοντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα επιτήρησης εφαρμόζοντας ένα σύστημα χωροταξίας θαλάσσιας χωροταξίας μπορούμε να συνδυάσουμε τις δραστηριότητες ώστε να μην έχουμε επικάλυψη και επίσης μπορούμε να αξιοποιήσουμε την έρευνα για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. κυρία το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Δαμανάκη για την διάβγεια των απαντήσεων και την ειλικρίνειά σας. Συμφωνώ με την αποκέντρωση και περιφερειοποίηση της αλλιευτικής πολιτικής, διότι αυτό ορίζει και το πρωτόκολλο της συνθήκης της Λισαβόνας μέσα στα πλαίσια της επικουρικότητας. Μιλήσατε για ασφάλεια, θαλάσσια ασφάλεια, για τα πρόσωπα, για την μεταφορά, για τα πλοία. Μιλήσατε για διάρκεια και συνέχεια στις συμφωνίες με τρίτες χώρες Γνωρίζετε ότι εμείς αντιμετωπίζουμε μεγάλο πρόβλημα με την συμφωνία με τη Σομαλία στον Ινδικό ωκεανό, ε, δηλαδή των πλοίων που αλλιεύουν στον Ινδικό ωκεανό. Ξέρετε ε, ότι αντιμετωπίσαμε μια κατάσταση πειρατείας με ένα βασκικό αλλιευτικό πρόσφατα και θα ήθελα να σας ε, ρωτήσω το εξής, λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ατλάντα καλύπτει τα εμπορικά, τι θα κάνετε σε σχέση με την ανανέωση των συμφωνιών και τι θα κάνετε σε σχέση με τα αλλιευτικά που δρούν στον Ινδικό ωκεανό. Θα πρέπει <laughs> να απαντήσει κυρία Δαμανάκη, αλλά βλέπω ότι από την Επιτροπή Τράνη είσαστε οι χειρότεροι, μακράν χειρότεροι. Κυρία Δαμανάκη, Κυρία Δαμανάκη, έχει δύο λεπτά. Ε, θα ήθελα να απαντήσω στην κυρία συνάδελφο. Ε, πράγματι <coughs> ε, υπάρχει θέμα για την καλύτερη να εξασφαλίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση καθεστώς ασφάλειας ε, για τα πλοία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ψαρεύουν σε δύσκολες περιοχές όπως είναι ο κόλπος της Σομαλίας. Ε, έχω δε την εντύπωση ότι αυτό είναι ένας από τους κύριους στόχους που πρέπει να πετύχουμε στις διεθνείς συμφωνίες. Έχω την εντύπωση ότι και η δική μας βιομηχανία η αλληλευτική βιομηχανία ε, θέλει τις ε, συμφωνίες περισσότερο για λόγους ασφάλειας. Θέλει να εξασφαλίσει ότι υπάρχει ένα ασφαλές περιβάλλον μέσα στο οποίο μπορεί να ψαρεύει. Η πειρατεία είναι ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα. Ε, ε, βασικό πλοίο στο οποίο αναφερθήκατε έχω την εντύπωση ότι ανέβασε τον αριθμό των ανθρώπων που κρατούν οι πειρατές σε 273, αν δεν κάνω λάθος. 273-276 μιλούμε για ένα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων και σκεφτείτε τις οικογένειες και όλα τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Η επιχείρηση Αταλάντα δεν καλύπτει πράγματι τα αλλιευτικά πλοία. Δεν τα καλύπτει. Έχετε δίκιο, κυρία συνάδελφε, σε αυτό. Γίνεται μια προσπάθεια από τα κράτη-μέλη να λύσουν το πρόβλημα έχουν στείλει εκπροσώπους ε, στο αρχηγείο της ε, επιχείρησης Αταλάντα που είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Γίνεται μια προσπάθεια να συντονιστούμε καλύτερα. Κάποιες χώρες, η Γαλλία νομίζω σκέφτεται να έχει ειδική συνοδεία για τα σκάφη της. Άλλοι σκέφτονται να επιτρέψουν τη χρήση όπλων. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Ε, νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να δούμε πώς θα συντονιστούμε ώστε να έχουμε, αν είναι δυνατόν, κάλυψη και των ε, σκαφών από την από την Ευρώπη με έναν πιο ε, συστηματικό τρόπο. Κυρία Μπιλμπάου, σας παρακαλώ πολύ εν συντομία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και θα ήθελα να λάβετε υπόψη τη διεύρυνση της ε, προστασίας στα πλαίσια της επιχείρησης ε, Ατλάντα και στα αλληλευτικά, διότι μέχρι τώρα δεν έχουμε δράσει καθόλου επί του θέματος. Θέλετε να απαντήσετε κυρία Δαμανάκη, φαίνεται πως όχι. Ο κύριος Τούσας έχει το λόγο. Για ένα λεπτό. Ο διεθνής χαρακτήρας ε, της ναυτιλιακής βιομηχανίας καθιστά στρατηγική σημασία στο ρόλο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού και της Διεθνούς Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών του 1982, Ανκλός, για το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Είναι μια βασική παράμετρος που δεν, να μας, δεν πρέπει να μας διαφεύγει από κανέναν σε ό,τι αφορά αυτό. Η στρατηγική της κοινή ναυπηλιακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων των κρατών μελών με κριτήριο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ναυτιλιακών επιχειρήσεων με προκλητικές φοροαπαλλαγές κατάργηση του καμποτάζ και πακτολό επιδοτήσεων αύξησε σε αστρονομικά επίπεδα τα κέρδη του εφοπλιστικού κεφαλαίου και των μονοπαλιακών επιχειρήσεων και ομίλων του κλάδου. Από την άλλη πλευρά, σε ό,τι αφορά τους ναυτεργάτες, διαπιστώνεται με μεγαλύτερη ένταση ο μαζικός διωγμός τους από τα καράβια, χειροτέρευση των όρων δουλειάς και αμοιβή, εντατικοποίηση της δουλειάς στο έπακρο αυξάνοντας τους κινδύνους για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και την προστασία του περιβάλλοντος. Η πολιτική αυτή υποβάθμισε τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες και επέφερε ισχυρό πλήγμα στα κοινωνικά στρώματα που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Πώς αξιολογείται αυτό το απαράδεκτο καθεστώς των φοροαπαλλαγών που έχει νομοθετηθεί στα πλαίσια των 27 κρατών για το εφοπλιστικό κεφάλαιο, πώς τοποθετήστε πάνω στα αιτήματα των αυτεργατών και γενικότερα των εργαζομένων των κατοίκων των απομακρυσμένων περιοχών. Κύριε, Τούσα, δεν μπορείτε να δευτερολογήσετε διότι εξαντλήσετε το χρόνο. Κύριε Αδαμανάκη, για δύο λεπτά. Συμφωνώ με τον κύριο συνάδελφο ότι το διεθνές δίκαιο της θάλασσας πρέπει να εφαρμοστεί. Συμφωνώ επίσης ότι ο IMO, ο Διεθνής ε, Ναυτιλιακός Οργανισμός παίζει έναν κυρίαρχο ρόλο, ο οποίος είναι επίσης σεβαστός και θα πρέπει να συνεργαστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτά όλα, κατά τη γνώμη μου, δεν έρχονται καθόλου σε αντίθεση, αντίθετα βοηθούν και επισημαίνουν την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει τη δική της ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική και πολιτική για την ναυτιλία. Ε, έτσι ώστε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Ε, δεν θέλω να επισέλθω σε ζητήματα που έχουν σχέση με την άσκηση οικονομικής και φορολογικής πολιτικής από την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Κομισιόν. Ε, η αρχή της collegiality principle, η αρχή της συλλογικότητας στα πλαίσια της Επιτροπής με καλύπτει απολύτως το θέμα αυτό. Συμφωνώ όμω ότι πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για του ναυτικού μα και στα πλαίσια τη ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, εδώ μου πέφτει και εμένα κάποιο λόγο. Ε, πιστεύω πως όλοι έχουμε την ίδια ευαισθησία, κύριε Τούσα. Το ότι εγώ δεν μπορώ να αναφερθώ συγκεκριμένα στα θέματα που θέτετε λόγω αρμοδιοτήτων δεν σημαίνει ότι δεν συμμερίζομαι και τη δική σας ευαισθησία, όπως και πολλοί συνάδελφοι εδώ, συνάδελφοί σας και πιστεύω και η Επιτροπή. Ε, όσο με αφορά, θέλω να πω ότι θα εγκαινιάσω διάλογο με τα συνδικάτα αυτό είναι που μπορώ να δώσω στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μου. Δεν υπήρχε μέχρι τώρα διάλογος με τα συνδικάτα των ε, εργαζομένων στον τομέα της αλίας και της ναυτιλίας. Αυτό είναι ότι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε και θα κάνω επίσης ό,τι μπορώ ώστε να υπογραφεί η τελευταία σύμβαση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας για, το... για τα δικαιώματα των ναυτικών. Υπάρχει σύμβαση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας εδώ και δύο χρόνια δεν την έχει υπογράψει καμία χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την έχουν υπογράψει κάποιες άλλες χώρες. Θα συνεργαστώ με τον Επίτροπο τον Αρμόδιο για τα θέματα αυτά, τον Επίτροπο τον ε, Υπεύθυνο για τα κοινωνικά θέματα, ο οποίος επίσης έχει ενημερώσει ότι θα πάρει σχετικές πρωτοβουλίες στον τομέα αυτό. Έχετε 30 δευτερόλεπτα για, για συμπληρωματική ερώτηση κύριε Τουσο. Μόνο 30 δευτερόλεπτα. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ σε ένα ίσω τομέα που δεν είναι στους φακέλους που έχει αναλάβει η κυρία Επίτροπο, Αλλά παραμένει σοβαρό πρόβλημα σε ό,τι αφορά την προστασία τη ανθρώπινη ζωή στη θάλασσα και του περιβάλλοντο. Είναι διαπιστωμένο από τι αρχέ τη δεκαετία του 1980 στη Μεσόγειο θάλασσα, στη Βαλτική θάλασσα, ότι υπάρχουν μεγάλα ναυάγια που υπάρχουν, αποτελούν σαν την αποθήκη για τη μόλυνση του περιβάλλοντος. ποτίθεστε να συμβάλλετε έτσι ώστε να ανελκυστούν αυτά τα ναυάγια. Με απόλυτο σεβασμό της αρχής της κολεγιάλιτης στην Επιτροπή θα κάνω ό,τι μπορώ κύριε Τούσα. Πράγματι θα κάνω ό,τι μπορώ με σεβασμό όμως την αρχή της κολεγιάλιτης στα πλαίσια της Επιτροπής, ώστε να αποκρουστούν αυτές τις περιπτώσεις. Άλλωστε, αν πω τίποτα περισσότερο για τα ε, safety packages, τα οποία έχουμε στην ε, θάλασσα, το, τα, τα packages, οι συνάδελφοι από την Επιτροπή Transport ενδεχομένως θα με κατηγορήσουν ότι επισέρχομαι σε ζητήματα του Επιτρόπου Κάλλας. Θέλω να καταλάβετε τη δύσκολη θέση μου. Ευχαριστώ πολύ. Ακολουθεί για ένα λεπτό η κυρία Γόσμπαχ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι δύσκολο να είναι κανείς στο τέλος του καταλόγου αγοριτών μετά από άλλα 30 άτομα. Θέλω να πω κάτι για τις παράκτιες αλή, δραστηριότητες αλίας. Πρέπει να δούμε ότι και αυτό είναι μια δυνατότητα γιατί βοηθάει τη διατήρηση θέσεων απασχόληση σε τοπικό επίπεδο σε ό,τι αφορά τις ε, διαδικασίες αλίας. Μιλάμε μέχρι στιγμή πάρα πολύ για τη βιομηχανική αλία, αλλά θα θέλατε ένα τμήμα των ποσοστώσεων για την αλλία να διατηρηθεί αποκλειστικά και μόνο για την παράκτια αλία για να μπορέσουμε να έχουμε φιλική προς το περιβάλλον μεταχείριση και μεταφορές οι οποίες είναι φιλικές στις περιοχές αυτές στο περιβάλλον. Επίσης να έχετε με μέτρα προστασίας για τα νεαρά ψάρια για να μπορούν να μεγαλώσουν χωρίς να έχουν κίνδυνο αλλιεύση. Δύο λεπτά. Ε, θα ξεκινήσω από το τελευταίο που το θεωρώ πολύ σημαντικό. Είναι ανάγκη πράγματι να προστατεύσουμε τα νεαρά ψάρια. Γιατί αν ε, δεν ε, τα στείλουμε πίσω για να φέρουν τους γονείς τους <laughs> σε εμάς, πραγματικά τα αποτελέσματα της αλληλείας θα είναι πολύ πενιχρά. Πώς μπορεί να γίνει αυτό. Ε, νομίζω ότι οι επιστημονικές μέθοδοι και τα εργαλεία πολιτικής που έχουμε στα χέρια μας είναι συγκεκριμένα. Προϋποθέτουν βέβαια να έχουμε μια καλή χαρτογράφηση των περιοχών όπου γίνεται η αναπαραγωγή και θα μπορούσαμε ίσως να δούμε τα κράτη-μέλη να ε, δουν σε αυτές τις περιοχές να υπάρχει ένα ειδικό καθεστώς προστασίας για αυτές τις περιοχές όπου γίνεται η αναπαραγωγή. Θα μπορούσαμε επίσης να δούμε την απαγόρευση της αλίας στο διάστημα που τα νεογνά είναι πολύ μικρά, ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Πρέπει να εργαστούμε πιο συστηματικά και πιο συντονισμένα σε αυτή την κατεύθυνση με τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να κατανείμουν τις ποσοστώσεις, τις οποίες εμείς κατανέμουμε κεντρικά για τα διάφορα είδη. Επομένως, τα κράτη-μέλη μπορούν να πάρουν υπόψη την πολύ ε, ε, λογική πρόταση που κάνετε να υπάρχει ε, χρησιμοποίηση αυτών των ποσοστώσεων έτσι ώστε να ενισχυθούν τα μικρά σκάφη. Εμείς σε κεντρικό επίπεδο θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε η πολιτική μας να έχει τις, τα απαραίτητα εργαλεία, να δίνει τα απαραίτητα εργαλεία και τη χρηματοδότηση για την ανανέωση των μικρών σκαφών. Είμαι απόλυτα πεπισμένη ότι το κύριο πρόβλημα είναι αυτό το να έχουμε μικρά μοντέρνα σκάφη που να έχουν τα εργαλεία, να έχουν ε, ε, τις δυνατότητες που δίνει η νέα τεχνολογία, ώστε και να ξέρουν που ψαρεύουν και να ξέρουν τι ψαρεύουν, να βλέπουν το μέγεθος των αλλιευμάτων, να βλέπουν κατά πόσο υπάρχουν μικρά, να βλέπουν κατά πόσο υπάρχουν, θα υπάρχουν απορρίψεις και να κάνουν τις κατάλληλες ενέργειες για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Νομίζω μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ε, Eh, eh, Ευχαριστώ. Μπορείτε ε, να δευτερολογήσετε για ένα λεπτό. Και τώρα θα ήθελα να αναφερθώ και πάλι για τα νεαρά ψάρια, τα ηχθίδια και για τα μικρά σκάφη αλίες. Το ερώτημα μου είναι το εξής. Εσείς θα αγωνιστείτε ώστε να ακολουθηθεί μια πολιτική ώστε όλα τα ψάρια να εκφορτώνονται και να μην απορρίπτονται. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τροποποιηθεί και το όλο σύστημα των ποσοστώσεων. Έχετε μια λύση να προτείνετε για το θέμα αυτό. Ε, ε, η κυρία Ρόσμπας μεταφέρει εδώ την πολύ θετική πείρα της Δανίας ενδεχομένως. Ξέρετε ότι η Δανία έχει, ε, έχει, συνολικό, έχει απαγορεύσει συνολικά τις απορρίψεις ε, εμείς όμως χειριζόμαστε το ζήτημα πιο προσεκτικά διότι υπάρχουν άλλες χώρες όπου δεν είναι εύκολο να γίνει αυτό. Αυτό το οποίο προς το παρόν κάνουμε για τις απορρίψεις είναι ότι έχουμε απαγορεύσει την πολιτική του overgrading όπως λέμε. Απαγορεύουμε δηλαδή να ρηχτούν ψάρια στη θάλασσα και να μπουν άλλα μεγαλύτερου είδους προκειμένου να πετύχει καλύτερη τιμή στη σοδιά του ο ψαράς. Επίσης συζητούμε στα πλαίσια της αναμόρφωσης του ε, ε πράσινου βιβλίου, στα πλαίσια της αναμόρφωσης της ε, κοινή αλλιευτικής πολιτικής, όλο αυτό το θέμα των απορρίψεων, το οποίο πολύ σωστά θέτεται και νομίζω ότι θα πρέπει να οδηγηθούμε σε μια πιο αποτελεσματική πολιτική για τις απορρίψεις. Πιο αποτελεσματική πολιτική για τις απορρίψεις. Εάν ε, ψαρεύει ένας ψαράς ένα μόνο είδος, εάν δηλαδή κατατείνει σε ένα ε, ε μόνο είδος, πρέπει να δούμε ειδικά μέτρα που αφορούν την επιλεξιμότητα των εργαλείων. Εάν έχει περισσότερα είδη, περισσότερα είδη, τότε ίσως μπορούμε να πάμε σε μια μεγαλύτερη, πιο αυστηρή λογική απαγόρευση των απορρίψεων. Αλλά συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να κάνουμε προσπάθεια ώστε οι απορρίψεις να ανήκουν στο παρελθόν. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα, έχουμε λίγα ψάρια είναι πραγματικά εκτός λογικής, να μην πω ότι είναι ανήθικο, ίσως δεν έχει πολιτική σημασία όρος, να ρίχνουμε ψάρια που, πιάνουμε πίσω στη θάλασσα. Δεν μπορούμε να το αντέξουμε αυτό. Τέλος, για να κλείσουμε, με τις παρεμβάσεις των βουλευτών, ο κύριος Δεγράνδες Πασκουάλ, για ένα λεπτό. <clears throat> Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υποψήφια Επίτροπε. Στην προηγούμενη θητεία οι προσπάθειές μας για μια κοινή πολιτική μεταφορών δεν οδήγησαν σε μια επιτυχία, μάλλον σε μια ε, αποτυχία σε ό,τι αφορά τα θέματα της θαλάσσιας ασφάλειας. Η αποτυχία μας ήταν το ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεν μπορούσαν να επιτύχουν τη φιλελευθεροποίηση σε επίπεδο λιμένων με το πακέτο ΕΡΙΚΑ 3 κτλ. Και δεν μπορέσαμε να προχωρήσουμε σε διατροπικές πλατφόρμες για τις θαλάσσιες μεταφορές. Έχετε κάποια σχέδια για να μπορέσετε να αναπτύξετε περισσότερο τα λιμάνια και να ξεπεράσουμε αυτό το θέμα που έχει μείνει εκρεμές. Δύο λεπτά. Ε, ε, η οικονομική πλευρά της πολιτικής ε, των λιμανιών και το ιδιοκτησιακό του καθεστώς δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Περισσότερο θα έλεγα ότι είναι στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Μεταφορών και του Αρμοδίου Επιτρόπου. αυτό το οποίο ενδιαφέρει και αυτό το οποίο θα ήθελα να επιμείνω είναι πώς θα συνδυαστεί η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, αυτό που λέμε Integrated Maritime Policy, με συνθήκες ασφάλειας στα λιμάνια, με τη δυνατότητα πρόσβασης όλων στα λιμάνια και με τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια. Αυτά πρέπει να προσπαθήσουμε να τα εξασφαλίσουμε διότι αφορούν και την αλία μας. Έχω ενημερωθεί, για, έχω ενημερωθεί όσο μπόρεσα να ενημερωθώ για τα σχέδια της αρμόδιας διεύθυνσης μεταφορών και τα σχέδια του αρμόδιου επιτρόπου. Ε, θέλω να πω το εξή. Έχουμε συζητήσει το θέμα αυτό ε, και στο Κολέγιο των Επιτρόπων, στο Κολέγιο, το Designated College. Και θέλω να αναφερθώ σε αυτό που υπάρχει και στα guidelines του Προέδρου Μπαρόζο, στι κατευθυντήριε γραμμέ του Προέδρου Μπαρόζο, ο οποίο έχει πει ότι τον επόμενο χρόνο θα έχουμε να δώσουμε, να παρουσιάσουμε ως Επιτροπή πλέον, όχι ως Επίτροπος Αλίας, μία έκθεση για το καθεστώ της εθνικής βοήθειας ε, των κρατών μελών σε σχέση με τα λιμάνια, και μία δεύτερη έκδοση που θα αφορά τις επιχειρήσεις κοινή ωφελία. Θεωρώ τις εκθέσεις αυτές πολύ σημαντικές. Στα πλαίσια των συζητήσεων αυτών πιστεύω ότι η Επιτροπή θα καταλήξει στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αλλά πραγματικά δεν θέλω να επισέλθω σε θέματα που είναι αρμοδιότητες άλλων επιτρόπων αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Έχετε δικαίωμα δευτερολογία. Ναι, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρία Υποψήφια Επίτροπε. Ευχαριστώ για τα λόγια σα. Δυστυχώ όμω Νομίζω ότι όλοι μας θα φύγουμε από αυτή την ακρόαση χωρίς να ξέρουμε ακριβώς, επακριβώς ποιες είναι οι αρμοδιότητες για τη Γενική Διεύθυνση θαλασσίων θεμάτων και τα θέματα της δικής της αρμοδιότητας. Ελπίζω λοιπόν θα μπορέσει να υπάρξει επωφελή συνεργασία με τους άλλους επιτρόπους και η πολιτική ασφάλειας είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την θαλάσσια ασφάλεια και ελπίζω ότι το Σώμα των Επιτρόπων στο σύνολό του θα προχωρήσει στη σωστή ρύθμιση των θεμάτων των λιμένων. Κύριε Δαμανάκη, έχει το λόγο. Ότι χρειάζεται καλύτερη αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων ανάμεσα στις διάφορες διευθύνσεις και στους διάφορους επιτρόπους ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ειλικρινά ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Και να σας υπενθυμίσω ότι και στην προηγούμενη, στη διάρκεια της προηγούμενης επιτροπής, από ό,τι γνωρίζω έχετε ε, μακρόχρονη εμπειρία για το θέμα αυτό. Υπήρχε αυτό το steering committee, υπήρχε μια επιτροπή 10 επιτρόπων, όπου ήταν μετήχε και ο Επίτροπος από τις ε, μεταφορές, με την προεδρία του Επιτρόπου για τη θαλάσσια πολιτική, του κυρίου Μπόρτς, ε, η οποία έλυνε οποιαδήποτε ζητήματα ενδεχομένως ανέκυπταν. Ε, ελπίζω ότι θα συνεχίσει αυτή η λειτουργία και θέλω να σας πω ότι αν συνεχίσει να λειτουργεί αυτή η Επιτροπή, εάν επιβεβαιωθώ ως Επίτροπος και αν έχω την έγκρισή σας και επιβεβαιωθώ και έχω την ε, Προεδρία αυτής της Επιτροπής, θα κάνω ότι καλύτερο μπορώ ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα. Θέλω να πω επίσης ότι θεωρώ πολύ σημαντικό γιατί να απαντήσω στο ερώτημά σας, ίσως σημαντικότερο και από την παρουσία μου εδώ ή την αντίστοιχη παρουσία του κυρίου Κάλλας, τη συνεργασία των υπηρεσιών στον τομέα αυτό είναι ανάγκη να έχουμε καλή συνεργασία στι υπηρεσίε μα και να μην προσπαθήσει ο ένα να πατήσει το πόδι του άλλου. Και ίσω να χρειαστεί να υπάρξει ένα inter-service group, όπω λέμε, μια διαυπηρεσιακή συνεργασία, ώστε να εξασφαλίσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Δεν είναι το θέμα των αρμοδιοτήτων το κύριο. Το κύριο είναι ότι επιτέλου η Ευρώπη θα έχει ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική και είμαι περήφανη που μπορώ και εγώ να συμβάλλω σε αυτό. Ε, Ευχαριστούμε πολύ σε όλους. Τελειώσαμε στην ώρα μας. Ε, με μερικούς ήμουνα πιο αυστηρή, αλλά χρειάστηκε να γίνει κάτι τέτοιο. Θα ήθελα να δώσω τέλος το λόγο στην υποψήφια επίτροπο για 7 λεπτά, έτσι ώστε, εάν το επιθυμεί, να συνοψίσει και στη μηνιά μισή θα βρεθούμε στην αίθουσα 1-5 οι αντιπρόεδροι, οι συντονιστές και οι υπάλληλοι των πολιτικών ομάδων για να γίνει η αξιολόγηση. Έχετε το λόγο κυρία Δαμανάκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ το Προεδρείο για την διαδικασία και ευχαριστώ και όλους τους κυρίους βουλευτές για τις ερωτήσεις που μου έθεσαν Ευχαριστώ επίσης και όσους δεν έθεσαν ερωτήσεις και μας άκουσαν υπομονετικά. Ε, ε, το, ε, ευχαριστώ για τις ερωτήσεις και δεν το λέω μόνο τυπικά, το λέω και ουσιαστικά. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις γιατί ήταν πραγματικά σε ζητήματα ουσίας. Έτσι μου δώσατε τη δυνατότητα να σκεφτώ ότι άξιζε η πολύ σκληρή δουλειά των δύο τελευταίων μηνών για να ενημερωθώ για τα ζητήματα του χαρτοφυλακίου μου. Θέλω να σας εξομολογηθώ ότι όταν ανέλαβα αυτό το χαρτοφυλάκιο ε, με τρόμαξε η μεγάλη τεχνική λεπτομέρεια στην οποία έπρεπε να επισέλθω αλλά ε, εν τέλει ε, κατάλαβα ότι τα πράγματα έχουν μια ορισμένη λογική και ότι αν ξεκαθαριστούν οι στόχοι και οι αρχές που πρέπει να υπηρετήσουμε τα πράγματα μπορούν να γίνουν ευκολότεροι για όλους όλοι οι κύριοι βουλευτές έθεσαν ζητήματα τα οποία θα τα συζητήσουμε στα θέματα της αναμόρφωσης της κοινή αλλιευτικής πολιτικής όσον αφορά την αλληλεία. Ετοιμάζετε κι εσείς ως Επιτροπή μια έκθεση για την αλληλεία, για τον το Green Book που έχουμε, για το CFP Reform. Η κυρία Νέβες είναι εδώ. Θα ενημερωθώ και για τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί και πιστεύω ότι αυτή η έκθεση θα βοηθήσει πολύ και θα παίξει ασφαλώς πολύ σημαντικό και καθοριστικό ρόλο ε, τον επόμενο χρόνο ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Τον επόμενο χρόνο πρέπει να βάλουμε τον πύχη ψηλά. Το 2010 είναι έτος βιοπικιλότητας και πρέπει τουλάχιστον η Επιτροπή μας, θα έλεγα να συνεισφέρει θετικά, αλλά τουλάχιστον να μην απογοητεύσει αυτούς που περιμένουν να ανταποκριθούμε στο καθήκον αυτό. Να συμβάλλουμε κι εμείς στο να διατηρηθεί η βιοπικιλότητα του πλανήτη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και όπως ήδη υπόθηκε, 70% του πλανήτη είναι νερό. Και επομένως είναι θάλασσες, είναι ωκεανοί και επομένως η ευθύνη είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τα ζητήματα που έχουν σχέση με την άσκηση πολιτικής στην Αλία θα τα δούμε μαζί. Ξέρετε ότι το άρθρο 43, παράγραφος 3 της συνθήκης δίνει τη δυνατότητα στην Κομισιόν να αποφασίζει για τα ζητήματα αλίας θα εφαρμοστεί το άρθρο αυτό με τη μεγαλύτερη δυνατή αυστηρότητα, με τη μεγαλύτερη δυνατή αυστηρότητα, ώστε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή να συμμετέχει. Άλλωστε ήδη τον κανονισμό για τα technical measures, γι' αυτό που λέμε technical measures, θα τον συζητήσουμε μαζί το επόμενο διάστημα, τον έχουμε φέρει στην Επιτροπή, θα πάρουμε πολύ σοβαρά υπόψη τις γνώμες της Επιτροπής. Και οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με το management της πολιτικής, ε, στο βαθμό που δεν παραβιάζει τη συνθήκη, θα συζητείτε εδώ. Ε, υπήρξε πολύ μεγάλη συζήτηση για τη διεθνή παρουσία μας, τη διεθνή παρουσία της Ένωσης. Συμφωνώ, είναι πολύ σημαντική η διεθνής παρουσία. Ε, συμφωνώ επίσης ότι το Κοινοβούλιο έχει παίξει ένα εξαιρετικά θετικό ρόλο ε, στα θέματα των διεθνών συμφωνιών, των Fisheries Agreement, των Bilateral Fisheries Agreements που έχουμε υπογράψει. Ο ρόλος αυτός πρέπει να ενισχυθεί και θα κάνω ό,τι μπορώ στα πλαίσια των δυνατοτήτων μου για να ενισχυθεί. Πάντως εννοείται ότι οποιοδήποτε έγγραφο, ευρωπαϊκό έγγραφο, έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορά την άσκηση των αρμοδιοτήτων μου θα είναι στη διάθεσή σας. Όπως επίσης εγώ η ίδια προσωπικά θα είμαι στη διάθεσή σας για ενημέρωση εδώ στην Επιτροπή πριν και μετά από οποιαδήποτε διεθνή συμφωνία. Κατά τα άλλα θα ακολουθηθούν τα όσα θα αποφασιστούν με τις αρχές της collegiality στο New Framework Agreement ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Κομισιόν. Ε, υπήρξε επίσης πολύ μεγάλη αναφορά από πολλούς συναδέλφους στην ανάγκη από πολλούς ε, συγγνώμη λέω συναδέλφους γιατί νομίζω ότι είμαι ακόμα βουλευτής ε, ε, από πολλά μέλη, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου υπήρξε μεγάλη αναφορά στο θέμα της αποκέντρωσης των, της λήψης των αποφάσεων και της περιφερειοποίησης της πολιτικής μας. Decentralization και regionalization. Είναι πολύ δύσκολο θέμα. Είναι πολύ δύσκολο θέμα γιατί θέλουμε να τηρήσουμε τις ε, συνθήκες και συγχρόνως θέλουμε να δώσουμε έδαφος στις τοπικές κοινωνίες να αναπνεύσουν. Ε, μαζί με εσά, σε πραγματική συνεργασία και μαζί με την νομική υπηρεσία και την Επιτροπή όλοι, είμαστε φύλακες των συνθήκων, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Για να κλείσω, κυρία Πρόεδρε, Θέλω για μια ακόμα φορά να ευχαριστήσω την ε, Επιτροπή. Θέλω να σας βεβαιώσω ότι έχω αίσθηση των ευθυνών μου. Καταλαβαίνω ότι ο Επίτροπος Αλίας, εάν με επιβεβαιώσετε, αποφασίζει για πράγματα που έχουν πολύ συγκεκριμένες επιπτώσεις στη ζωή χιλιάδων ανθρώπων. Δεν αναφέρεται σε γενικές αποφάσεις. Αποφασίζει συγκεκριμένα μέτρα που μετρούν για χιλιάδες οικογένειες ψαράδων, ανθρώπων που εργάζονται σε αυτές τις περιοχές αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να έχουν μια καλή ζωή αυτή που η ζωή τους εξαρτάται από την αλία και θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να έχουμε μια καλή συνεργασία ώστε να εξασφαλίσουμε στην αλία ε, ένα βιώσιμο μέλλον. Θα κάνω επίσης ό,τι μπορώ ώστε αυτό το νέο μας παιδάκι, το Integrated Maritime Policy, να μεγαλώσει σωστά, να έχει την καλύτερη δυνατή μεταχείριση, να συνεργαστεί καλά με άλλες επιτροπές και άλλους επιτρόπους, έτσι ώστε να μπορέσει η Ευρώπη να έχει μια θαλάσσια πολιτική. Ε, έχω γεννηθεί στην Κρήτη. Ε, οι Μινοίτες ήταν από τους πρώτους λαούς στην Ευρώπη που έφτιαξαν καράβια και αρμένισαν στη Μεσόγειο. Θα είναι μεγάλη μου τιμή να δουλέψω μαζί σας για να προχωρήσουμε παραπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους τους συμμετέχοντες. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και τους διερμηνείς και φυσικά και την υποψήφια επίτροπο η οποία ήταν παρούσα μαζί μας και τέλος της συνεδρίασης. Bueno. <laughs> Yeah.